Ja. Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, ich begrüße Sie alle ganz herzlich zu unserer Sitzung. Σας καλωσορίσω στη συνεδρίασή μας. Δυστυχώς θα πρέπει να ξεκινήσουμε, γιατί έχουμε πάρα πολλά θέματα στην ημερήσια διάταξη. Ιδάλλως δεν θα προλάβουμε να τελειώσουμε όλα τα ζητήματα στην ημερήσια διάταξη. Wenn Sie einverstanden sind, ich empfehle das Αν συμφωνείτε και σας το συνιστώ επιφύλακτα, θα ήθελα να σας ανακοινώσω στο 2 μόνο ότι έχουμε πάρα πολλά θέματα στην ημερήσια διάταξη και το μόνο τρόπος να τα ολοκληρώσουμε όλα είναι να είμαστε όλοι σύντομοι και λακωνικοί. Ιδάλλως θα έχουμε πρόβλημα. Πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη, στο 3, το σημείο 3, ενδιάμεση επισκόπηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων πλοήγησης μέσω δορυφόρου. Ο κύριο Ρέμεκον είναι εισηγητής. Θα, θα πρέπει να το ολοκληρώσουμε γρήγορα το θέμα αυτό. Κύριε Ρέμεκ, σας δίνω το λόγο. Και θα, έχουμε, θα μετράμε το χρόνο ομιλία πάντα. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Φτάνουμε πλέον στο σημείο που έχουμε το σχέδιο έκθεσης. Είναι διαθέσιμο. Ελπίζω πως αυτή ήταν η τελευταία καθυστέρηση του ζητήματος, η τελευταία καθυστέρηση για ολόκληρο το πρόγραμμα Γαλιλαίο. Επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω διάφορους συναδέλφους, οι οποίοι εργάστηκαν πάνω στην έκθεση, καθώς επίσης και την Γραμματεία και τον Πρόεδρο της Επιτροπής, τον κύριο Ρόη, για τη στήριξη και την συνεργασία του. Επίσης θα ήθελα να πω ότι και οι συνεργάτες μας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπήρξαν ε, πραγματικά συνεργάσιμοι. Ε, Επειδή έχουμε πάρα πολύ λίγο χρόνο, Επιτρέψτε μου απλώς να πω ότι προφανώς ε, το σχέδιο έκθεσης περιλαμβάνει μόνο ένα μικρό μέρος από αυτό που και εγώ και άλλοι θα ήθελα να πούν πάνω στο ζήτημα. Ελπίζω ότι θα υπάρξουν πολύ επικοδομητικά σχόλια και προτάσεις για προσθήκες. Και στο τέλος ε, η έκθεση ελπίζουμε να εκφράζει την ε, συνένεση, την ομόφωνη γνώμη αυτής της Επιτροπής. Επιτρέψτε μου να υπενθυμίσω κάποια γεγονότα. Η απόφαση για, το σύστημα, για τη δημιουργία του συστήματος Γαλιλαίο βασίστηκε σε δύο λόγους. Στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη διασφάλιση σημαντικού μεριδίου αγοράς ε, στις κορυφαίες τεχνολογίες, στις πιο προηγμένες τεχνολογίες. Όλοι ξέρουμε ότι η οικονομική κατάσταση αυτού του σχεδίου, του προγράμματος δεν είναι η ιδανική, το οικονομικό του καθεστώς δηλαδή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι Σύμφωνα με τον παρόντα ε, προϋπολογισμό, μόνο 18 δορυφόροι μπορούν να λειτουργήσουν. Ωστόσο, για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε, να εκμεταλλευτούμε πλήρως το δυναμικό του προγράμματος Γαλιλαίο, θα έπρεπε να φτάσουμε στην ε, εκμετάλλευση της πλήρους λειτουργικής ε, δυναμικότητας του συστήματος. Επίσης, συνειδητοποιούμε ότι ο προϋπολογισμός, ότι είναι αναγκαίες κάποιες υπερβάσεις του προϋπολογισμού, και σίγουρα αυτές οι υπερβάσεις θα αποδώσουν, δηλαδή η απόδοση επί της επένδυσης θα είναι εξασφαλισμένη. Ε, θα έπρεπε να συζητήσουμε πώς να δημιουργήσουμε διαδικασίες για την υλοποίηση ενώ μιας τόσο εκτεταμένης και ολοκληρωμένης υποδομής αν θέλουμε να μην έχουμε παρόμοια προβλήματα στο μέλλον. Αυτά θα ήθελα να πω μόνο τώρα στην αρχή. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα σχόλια που ελπίζω πως θα επακολουθήσουν. Να σας ευχαριστήσω και για το ότι ήσασταν λακωνικός. Ο συνάδελφο Μπρεζίνα έχει πρώτο το λόγο. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο, Πρόεδρε. Στην, αφού διάβασα την, το σχέδιο έκθεσης, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ επαγγελματικό. Περιλαμβάνει πολλά χρήσιμα πράγματα και πολύ συνοπτικά αλλά και εύγλωτα συνοψίζει ε, τους κύριους άξονες πάνω στους οποίους πρέπει να προβληματιστούμε και στους οποίους πρέπει να προσφέρουμε λύσεις. Το σχέδιο έκθεσης δεν αποφεύγει κάποιες αμφιβολίες ε, για την λειτουργία του συστήματος μετά το 2014. Αναφέρει για παράδειγμα το θέμα του επιχειρησιακού κόστους και αναγνωρίζει και το γεγονός ότι ε, όταν μιλάμε για τόσο προηγμένες τεχνολογίες, τεχνολογίες εχμής, ε, η διαδικασία μερικές φορές είναι πιο σημαντική από τον στόχο από το σκοπό. Εκτός, δεν είναι μόνο το σύστημα που θέλουμε να εξασφαλίσουμε, αλλά και την διαδικασία ε, απόκτησης, πρόσκτησης ε, τεχνολογιών και μας, ενδιαφέρουν και μας ενδιαφέρει και ο αντίκτυπος που αυτό θα έχει στην οικονομία. Ε, έχει, έχει γίνει λόγος για τη διαχείριση του προγράμματος. Για παράδειγμα, δεν υπάρχει ένας κύριος διαχειριστής που θα λειτουργεί το σύνολο του Γκαλιλαίου, αλλά αυτό ισχύει για όλα τα μεγάλα ευρωπαϊκά προγράμματα υποδομών. Ευχαριστώ, κυρία Χόλ. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την εκθεσή του. Ευχαριστώ. Ε, συμφωνώ μαζί του με όσα λέει κυρίως στον παράγραφο 3 για την πρόθεση της διαφάνειας. Νομίζω ότι δεν είναι πολύ ικανοποιητική η κατάσταση σήμερα, καθώς η Κομισιόν λέει ότι χρειάζεται ακόμα 1,9 δις ε, ευρώ. Δεν έχουμε καμία πληροφορία για το πώς κατέληξε σε αυτά τα αριθμητικά στοιχεία και θα πρέπει να έχουμε στοιχεία επιτάπητος, θα πρέπει να μπορέσουμε ε, να έχουμε το νούμερο επί το οποίο συμφώνησαν τα τρία όργανα προς τιμών. Ε, είναι σαν να αναφέρεται κάτι έτσι στον αέρα. Και επίσης υπάρχει ένα κενό χρηματοδότησης και με ανησυχεί αυτό και ε, το πρόγραμμα πλαίσιο καλείται να καλύψει αυτό το κενό. Όμως ε, αυτό θα είναι κάτι ε, πολύ ακριβό αλλά είναι ζωτική σημασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την καινοτομία και για τη μελλοντική αποτελεσματικότητα του κόστους. Αν ε, δούμε τρόπους για το πώς μπορούμε να διαθέτουμε το Γαλιλαίο, θα προτιμούσα να εξετάσουμε ορισμένες από τις υπηρεσίες ε, που αναμένεται να προσφέρει σήμερα το Γαλιλαίο και κυρίως ε, την ασφάλεια των υπηρεσιών ζωής. Είναι κάπως επίμαχο το θέμα αυτό, γιατί πρόκειται για μία από την υπηρεσία που σημαίνει ότι απαιτείται ένα πλήρες πρόγραμμα Γαλιλαίο, αλλά υπάρχει επικάλυψη σε μεγάλο βαθμό σε σχέση με το τι θα προσφέρει και το έγνος έτσι λοιπόν, ε, μια υπηρεσία που σχεδόν έχει καταστεί ε, υπηρεσιακή για να βοηθά την ασφαλή προσγείωση των αεροσκαφών. Ε, και η ερώτηση είναι αν αυτή η πτυχή της ασφαλείας ζωής του Γαλιλαίου είναι απολύτως απαραίτητη και αυτό είναι κάτι που θα μπορούσε να διαρευνηθεί προκειμένου να μειώσουμε το κόστος του Γαλιλαίου. Από την άλλη, θα συμφωνούσα ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί να μην κάνουμε περικοπές χωρίς να σκεφτούμε τις συνέπειες και ανησυχώ κάπως ε, μήπως δεν έχει δοθεί επαρκής προσοχή στο ότι υπάρχει πραγματικός κίνδυνος για όλα τα παγκόσμια περιφερικά συστήματα, όχι μόνο για το Γαλιλαίο, ε, από ε, τον ε, ήλιο και αναμένεται ότι θα δημιουργηθούν κάποιες διαταραχές. Ε, θα ήθελα να υπάρχει σαφήνεια για το αν έχει ληφθεί υπόψη η πιθανή ζημιά που μπορεί να υποστούν ε, οι δορυφόροι, δηλαδή όταν ε, θα πρέπει να εξετάσουμε τον αριθμό των δορυφόρων προς εκτόξευση. Και θυμάμαι τι έγινε και με τους Κινέζους για το ραδιόφασμα, την ζώνη ραδιοφασμού που χρησιμοποιείται από τους Κινέζους ε, σήμερα και δεν έχει ξεκαθαριστεί από αυτού. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσει, αλλά νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να δεκτούμε ότι μπορεί οι Κινέζοι ε, να αρνηθούν ε, να υποχωρήσουν σε αυτό. Και τελικά πώ θα έχουμε ένα σύστημα Γαλλιό που να λειτουργεί πλήρω αν ε, υπάρχουν ε, παρεμβάσεις από τους Κινέζους ε, σε κάποια σημεία της ζώνης του ραδιοφάσματος. Αλλά επαναλαμβάνω, μου άρεσε πολύ η εκθέση του κυρίου Ρέμεκ και ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί του στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ πολύ. Κύριο Βέιμπερ είναι ο επόμενο που έχει το λόγο. Χαίρομαι και εγώ με την έκθεση του συναδέλφου Ρέμεκ που αναγνωρίζει την αναγκαιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση να δημιουργήσει μια υποδομή για τον Καλλιλέο τέτοια που να ανταποκρίνεται στους στόχους ούτω ώστε να μπορούμε να λειτουργούμε πλήρως. Δηλαδή, μια, ένας αστερισμός, θα λέγαμε 25 δορυφόρων, 27 δορυφόρων και όλα αυτά σε συνεργασία με τις υποδομές επιδάφους, όλα αυτά είναι απαραίτητα για να μπορέσει το πρόγραμμα Γαλιλαίο που είναι ε, πρόγραμμα φάρος να μπορεί να λειτουργεί με ακρίβεια, να εντοπίζει και να μπορέσει να υπάρξει συνέχεια στις υπηρεσίες. Σε αυτό το θέμα θα πρέπει εμείς να λάβουμε υπόψη ότι υπάρχει διεθνής ανταγωνισμό όπως υπογράμμιση προλαλήσασα, διεθνής συναγωνισμός όσον αφορά τα συστήματα δορυφόρων. Έχουμε τη Ρωσία Φερρυπίν, την Κίνα αλλά και την Ινδία Επίσης έχουμε το GPS της Αμερικής. Αυτή, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να επιταχύνουμε την προσπάθειά μας και το να το κάνουμε το 2019 όπως προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με την ανακοίνωσή της, νομίζω ότι αυτό μπορεί να είναι κάπως καθυστερημένα. Επιπλέον, να πω, επίσης υπάρχει θετική αντιμετώπιση της έκκλησης σε κομισιόν ούτως ώστε να δούμε τα θέματα που έχουν να κάνουν με το ρίσκο, το κόστος, όσον αφορά την, ε, το κόστος για την έναρξη του προγράμματος. Παράγραφος 4 στο κείμενο το οποίο έχει καταθεθεί και νομίζω εκεί πρέπει να κάνουμε μια τροπολογία. Υπάρχει το πρόβλημα του μονοπωλίου. Στα, στα πλαίσια αυτά που έχουμε το Σογιούς της Ρωσίας. Αυτό είναι αρνητικό. Και επιπτώσεις αρνητικές όσον αφορά το πρόγραμμα Γαλιλαίου. Πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Επίσης, κατ' εμέ, θα ήταν προτιμητέο για την Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει τη δυνατότητα να μπορέσει να κάνει κάποια επιλογή, να έχει δυνατότητες για να έχει μια ε, σταθερή, ένα σταθερό δορυφόρο. Έχουμε το, την Αριάδνη 5 που μπορεί να εκτοξεύσει το, το δορυφόρο. Όπως εξάλλου έγινε και με το Soyuz. Φαίνεται προσαρμογή της Αριάδνης 5 για το πρόγραμμα Γαλιλαίο είναι κάτι το οποίο είναι θετικό ε, στα πλαίσια του Arian Space όλα αυτά τα προγράμματα για να μπορέσει κανείς να ξεπεράσει τεχνικά προγράμματα. Το κόστος προβλέπεται μόνο στα 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Έχουμε δηλαδή τι συζητήσει οι οποίε συνεχίζονται ανάμεσα στην ΕΖΑ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ έχω καταταθέσει μια τροπολογία για την παράγραφο 4, έχει να κάνει με το βιομηχανικό χώρο, για να έχουμε μια σωστή ε, αντιμετώπιση του θέματος αυτού. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λάμπερτς, σας ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να εστιάσω σε δύο ζητήματα. Το πρώτο από αυτά Καταρχά θα πρέπει να ξέρουμε, αξιολογώντα τι διάφορες επιλογές που έχουμε, και αυτό το έχω επαναλάβει συχνά στο παρελθόν, αλλά δεν έχει έλθει ποτέ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας παρουσιάσει μια απλή δήλωση, η οποία να δηλώνει ότι αν επιλέξουμε το πλήρες σύστημα, αυτά είναι τα ωφέλη και ξέρουμε λίγο πολύ το κόστο ποιο είναι, αλλά ποια θα είναι τα επιπρόσθετα ωφέλη. Αυτό θέλω να μάθω αν μείνουμε που, όπου είμαστε σήμερα, ποια θα είναι τα ωφέλη με το αντίστοιχο κόστος και επίσης αν ακυρώσουμε όλο το project, όλο το σχέδιο, ξέρουμε φυσικά ότι δεν θα πετύχουμε, αλλά τι θα μας κοστίσει. Μόνο βάσει αυτών των κριτηρίων μπορούμε να πάρουμε μια σωστή απόφαση και ειλικρινά θα ήθελα τα αριθμητικά αυτά στοιχεία κάποια στιγμή να τα δω και μάλιστα σύντομα. Κατά δεύτερον, δεν υπάρχει σαφήνεια για την στρατιωτική χρήση του Γαλιλαίου. Κοιτάξτε, δεν λέω ότι είναι μη διοντολογικό, ανήθικο και απαράδεκτο να υπάρχει στρατιωτική χρήση ενός τέτοιου συστήματος. Άλλωστε και το GPS ξεκίνησε από το Υπουργείο Αμήνης ε, στην αρχή. Άρα αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα. Αν όμως αντιμετωπίζουμε ένα πρόγραμμα το οποίο έχει υπέρογκο κόστος, και το οποίο θα μπορούσε να έχει σημαντική στρατιωτική χρήση, ε, δεν καταλαβαίνω γιατί το κόστος του προγράμματος αυτό θα πρέπει να το αναλάβει μια πολιτική αρχή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηλαδή. Να είμαστε σαφείς δηλαδή. Α, αυτό που καθιστά το Γαλιλαίο πιο σημαντικό αν θέλετε και πιο θεμητό είναι οι στρατιωτικές του χρήσεις, λογικό μου φαίνεται να συνεισφέρουν και οι στρατιωτικέ αρχές προ αυτή την κατεύθυνση, προς τη χρηματοδότησή του. Αν όχι, να έχουμε στοιχεία. Το πρόβλημα όμως είναι ότι όλα αυτά είναι σκοτεινά. Θα θέλαμε λοιπόν να διελευκαθούν όλα αυτά για να καταλάβουμε τα επιχειρήματα. Αυτό που δεν μπορούμε να δεχτούμε είναι να προχωρήσουμε σε ένα σύστημα το οποίο ζητείται ουσιαστικά για στρατιωτικούς σκοπούς ενώ ουσιαστικά δεν θα είχαμε καθόλου στρατιωτική χρηματοδότηση και για την μηδενική λύση. Φυσικά ενδεχομένως να θέλουμε το Γαλιλαίο για να δείξουμε την ανεξαρτησία κατά κάποιο τρόπο της Ευρώπης. Ένα τέτοιο σύμβολο ασφαλώς και συνεπάγεται ένα μεγάλο κόστος, αλλά και από στρατιωτικής άποψης. Γιατί χρειαζόμαστε το σύστημα αυτό. Ενώ θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε άλλα συστήματα, κυρίως το GPS. Άρα δύο είναι τα ενδεχόμενα. Καταρχάς, είτε ως Ευρωπαίοι προχωραμένα ένα σύστημα το οποίο είναι αντίθετο ή εν δεν υποστηρίζεται από τη ΣΥΠΑ και γι' αυτό θέλουμε το ευρωπαϊκό σύστημα. Και τελευταία περίπτωση που συνέβη κάτι τέτοιο ήταν το 56 όταν οι Γάλλοι και Βρετανοί πήγαν στο Σουέζ. Ε, πόσο πιθανό είναι κάτι τέτοιο. Και ακόμα λιγότερο πιθανή θα ήταν η εναλλακτική λύση να προχωρούμε, δηλαδή ένα πρόγραμμα το οποίο ήταν αντίθετο στο συμφέροντα των ΗΠΑ. Αυτό δεν θεωρώ ότι είναι πιθανό. Ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Άρα αξίζει αυτό το σύμβολο την τιμή του Όλα αυτά αποτελούν κριτήρια βασικά για τη συζήτηση. Κοιτάξτε, γιατί 30 δισεκατομμύρια θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και για άλλους σκοπούς, εξίσου θεμητούς. Και δεν έχουμε, ξέρετε, όλα τα όλα τα στοιχεία της εξίσωσης για να μπορούμε να λάβουμε σωστή απόφαση. Ευχαριστώ, ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος και τώρα να δώσουμε στο λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι. Θα ήθελα καταρχά να ζητήσω συγγνώμη ε, εξ ονόματο του κυρίου Φαργούφ, του συναδέλφου μου, ο οποίο δεν έχει καταφτάσει ακόμα. Θεωρώ ότι η συζήτηση αυτή είναι μια συζήτηση μεταξύ ημών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα ήθελα να επικεντρωθώ σε κάποια βασικά ζητήματα. Να ευχαριστήσω καταρχάς τον κύριο Ρέμεκ για την εξαιρετική έκθεση και τους υπόλοιπους βουλευτές που συνεργάστηκαν για την έκθεση αυτή και κατά δεύτερον θα πρέπει να ζητήσουμε συγγνώμη. Να ζητήσουμε συγγνώμη που έχουμε καθυστερώσει για την έκθεση, με την έκθεση για την ανδιάμεση αν θεώρηση. Τουλάχιστον έχουμε καθυστερήσει πιο πολύ από ό,τι υπολογίζαμε στην αρχή και πολύ λυπάμαι που χρειάστηκε να περιμένει τόσο πολύ ο κύριος Ρέμε και κάτι που είχαμε υποσχεθεί ότι θα τηρήσουμε για τα θέματα επί της ουσίας τώρα τα οποία και αναφέρθηκαν. Θα ήθελα να αναφερθώ στο θέμα του, των λεπτομερών δαπανών πίσω από τα 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ για την ε, διάθεση του νέου συστήματος και για την κατανομή των ε, δαπανών αυτών. Μπορούμε να σας δώσουμε μια τέτοια κατάσταση και να σας αναφέρουμε για παράδειγμα σε ποιο πλαίσιο εντάσσονται όλες αυτές οι δαπάνες. Φυσικά αυτές οι πληροφορίες, ξέρετε, έχουν και μία αξία στην αγορά σε ό,τι αφορά και τη βιομηχανία και τους παράγοντες που συμμετέχουν στην κατασκευή όλων αυτών των ε, συντελεστών. Και άρα είναι λίγο λεπτό το θέμα. Δεν θέλουμε να σας ε, κρύψουμε τις πληροφορίες αυτές σε καμία περίπτωση, αλλά θέλουμε οι πληροφορίες αυτές να μην φτάσουν σε χέρια ε, εκείνων που θα μπορούσαν να τις καταχραστούν. Φυσικά όμως μπορούμε να σας διαθέσουμε αυτές τις πληροφορίες, αλλά θα πρέπει να συμφωνήσουμε επί του πλαισίου ε, στο οποίο μπορεί να γίνει αυτό. Μιλήσατε, κυρία Χόγκ, για το safety of life. Όντως, υπάρχει εδώ η δυνατότητα να γίνουν οικονομίες. Αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι το Safety for Life θα χρειαζόταν πολύ πιο πολλούς ε, σταθμούς ε, από ότι θα χρειαζόταν για παράδειγμα το έγνος. Ε, υπάρχει όντως η σκέψη να μην αφήσουμε κατά μέρος το Safety for Life, αλλά να βρούμε ένα σύστημα το οποίο θα ήταν διαλειτουργικό με το αμερικανικό GPS, θα λειτουργούσε δηλαδή σε όλο τον κόσμο, να υπάρχουν δύο διαλειτουργικά συστήματα. Αλλά να σας προειδοποιήσω, οι, σχετικές οικονομίες δεν είναι σαφείς, δεν είναι σαφές πόσο, τι, ποσό θα μπορούσαμε να εξοικονομήσουμε και εξακολουθούν να υπάρχουν εξάρτηση και από άλλες υπηρεσίες οι οποίες θα πρέπει να αντιρευνηθούν το θέμα, όμως ε, όντως είναι ένα θέμα το οποίο ε, θα χαρούμε να κοιτάξουμε, το έχουν δείξει άλλωστε και άλλοι. Θα εξετάσουμε λοιπόν τι δυνατότητες υπάρχουν για ποιο ποσό εξοικονόμησης δηλαδή. Τα Τελευταία παρατήρηση να απαντήσω σε αυτά που είπε ο κυρία Λάμπερτς. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και ποια τα μειονεκτήματα ενός ε, συνολικού συστήματος και όχι ενός μερικού συστήματος. Ε, δεν αποφάνθηκε ιδιαίτερα γι' αυτό η έκθεση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής. Να σα πω ότι υπάρχουν κάποιε εσωτερικέ σκέψει εσωτερικέ εσωτερικοί υπολογισμοί που υποδεικνύουν ότι σε ένα σύστημα 18 δορυφόρων, ένα ανεξάρτητο σύστημα χωρί να υπάρχει συνδυασμό και σύνδεση με το GPS, ε, η ακρίβεια θα ήταν 250 μέτρα. Ε, στα, 24 ε, δορυφόρους θα είχαμε ακρίβεια 16 μέτρων πιο μεγάλη δηλαδή από ότι με το GPS, με, τους 20, με 30 δορυφόρους θα είχαμε μια οριζόντια ακρίβεια 3 έως 4 μέτρων. Αυτό για να έχετε υπόψη σας λίγο ε, τα μεγέθη τα οποία συζητάμε. Φυσικά αυτά θα πρέπει να τα ερευνήσουμε μαζί με τους συναδέλφους και από την υπηρεσία για το διάστημα. Αλλά βλέπετε από τα στοιχεία αυτά ότι ένα ανεξάρτητο σύστημα, αν αυτό πραγματικά θέσουμε ως στόχο, θα πρέπει να αναπτυχθεί πλήρως 27, δηλαδή δορυφόροι συν κάποιοι δορυφόροι ε, ασφαλείας. Τώρα σε ό,τι αφορά για την χρηματοδότηση, τη στρατιωτική και την στρατιωτική χρήση, ξέρετε την χρήση των PRS για παράδειγμα, εμείς ε, ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορούμε να προδιαγράψουμε ποια θα είναι η χρήση και ο σκοπός χρήσης των συστημάτων αυτών μπορεί να είναι η προστασία από καταστροφές για την αστυνομία, μπορεί ασφαλώς να προορίζεται και για στρατιωτική χρήση. Και όντως, στην παρούσα φάση, θα πρέπει να κοιτάξουμε ε, ποια θα είναι η χρήση σε κάθε χώρα και ασφαλώς δεν θα υπάρχει χρήση σε κάθε χώρα. Πέρα από αυτό, θεωρώ ότι το πλαίσιο το οποίο θα καθορίσετε και καθορίζεται μάλλον μαζί με το Συμβούλιο στην ε, κανονισμό 683 του 2003 ότι πρόκειται για ένα πολιτικό σύστημα με πολιτικούς σκοπούς και ότι δεν είναι φαγητικό το σύστημα αυτό. Νομίζω ότι αυτό είναι βασικό και το διακρίνει από άλλα ε, διεθνή συστήματα. Εδώ θα περιοριστώ, Πρόεδρο, σε αυτά θα περιοριστώ και αν έχετε ασφαλώς άλλες ερωτήσεις, με χαρά μου να τις απαντήσω και να ευχαριστήσω και πάλι τον κύριο Ρέμεκ για την εξαιρετική του έκθεση. Σας ευχαριστώ. Κύριε Ρέμεκ, θέλετε να πάρετε και πάλι το λόγο για να ολοκληρώσετε. Ε, ε, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον Οικονομικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. καθώς ε, μας πιέζει ο χρόνος, δεν έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε όλα τα σχόλια και τις παρατηρήσεις ε, που ακούστηκαν από τους συναδέλφους. Βέβαια θα τα λάβω υπόψη όταν ε, θα προσπαθήσουμε να συμπεριλάβουμε τις τροπολογίες στην έκθεση με τους σκιώδεις συζητητές. Και κατόπιν θα παρουσιάσουμε στην Επιτροπή μια αναθεωρημένη έκθεση. Θα ήθελα επίσης να αναφέρω το εξής έχω προετοιμάσει και μία αιτιολογική έκθεση όπου περιλαμβάνονται πολλές ε, πληροφορίες. Στην ε, έκθεση αυτή λέμε ότι το σύστημα έγνος ε, δεν είναι απολύτως ανεξάρτητο. Λαμβάνει και σήματα και από τους άλλους δορυφόρους, από τα υπόλοιπα δορυφορικά συστήματα και σε ό,τι αφορά την στρατιωτική χρήση. Κάτι που ίσως δεν είναι τόσο γνωστό και υπάρχει ευρία εμπειρία εδώ και 30 χρόνια είναι ότι τελικά οποιοδήποτε σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για στρατιωτικούς σκοπούς. Χωρίς αυτό να προσδιορίζεται από τον προτέρων. Έχουμε παραδείγματο χάρη σε δρόμου, ε, εργοστάσια παραγωγή ενέργεια, όλα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για στρατιωτικού ε, σκοπού. Το ίδιο ισχύει και με τα δορυφορικά συστήματα επιλογή. Αν συμφωνήσουν οι κυβερνήσει, δεν εξαιρούνται αυτά. Ευχαριστώ. Να σας ευχαριστήσω και πάλι να σας ε, διευκρινίσω ότι η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών είναι η 10η Μαρτίου 12 το μεσημέρι. Και τώρα θα ήθελα, αν συμφωνείτε, να περάσουμε στο επόμενο θέμα, σε εκ νέου εξέταση του θέματος της πολιτικής για το ραδιοφάσμα. Και έχουμε τον εισηγητή μας, τον συνάδελφο Εκμάρκ. Να του δώσω το λόγο. Γκούνας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω στις μέρες μας όλοι βλέπουμε τον αντίκτυπο του κινητού ίντερνετ και των κινητών συνδέσεων στην καθημερινότητά μας. Το είδαμε στις, στη Λιβύη, στην Αίγυπτο, στην Τινησία. Αυτό είναι ένδειξη των επιπτώσεων που οι καινούργιες ε, τεχνολογίες της πληροφορικής έχουν στις κοινωνίες και στις οικονομίες. Και αυτό είναι κάτι που δεν βρίσκεται στην αρχή του γιατί βλέπουμε όλο και περισσότερο να επεκτείνεται το φαινόμενο. Η το κινητό διαδίκτυο και οι κινητές υπηρεσίες αποτελούν έδαφος για την παροχή νέων υπηρεσιών και για μεταβολές της οικονομίας. Έχουμε δει πόσο έχει αλλάξει και η ευρωπαϊκή και η αμερικανική οικονομία και βλέπουμε ότι αλλάζει η παγκόσμια οικονομία. Κύριε Πρόεδρε, Έχω ένα μάλλον ταπεινό σκοπό ε, για την παρουσία μας εδώ. Θα ήθελα η Ευρώπη να είναι η καλύτερη στη διαδικασία αυτή. Γιατί βλέπουμε πόσο κρίσιμη σημασία είναι να βρίσκεται κανείς στην πρωτοπορία της χρήσης ε, των κινητών ευρυζωνικών υπηρεσιών, του κινητού διαδικτύου και όλων των υπηρεσιών που εφαρμόζουν αυτή τη τεχνολογία. Είναι κρίσιμη σημασία για τους πολίτες της Ευρώπης για την ανάπτυξη του πολιτισμού στην Ευρώπη, για την ανάπτυξη ε, των ειδησιογραφικών ειδήσεων, των νέων μέσων, αλλά και για την οικονομία. Νομίζω ότι λίγα ζητήματα έχουν τόσο μεγάλη σημασία για το να καταστεί η ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά πραγματικότητα. Ε, ε, ε, υπάρχει μια ευκαιρία να έχουμε μια ψηφιακή εσωτερική αγορά και να χρησιμοποιηθεί αυτό ως εφαλτήριο για την πρόοδο της ευρωπαϊκής οικονομίας. Όταν συζητήσαμε το θέμα αυτό, υπογράμμισα το γεγονός ότι ούτε οι Ηνωμένε Πολιτείε ούτε η Κίνα δεν είναι οι μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου, είναι η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά οι Ηνωμένε Πολιτείε και η Κίνα έχουν τις μεγαλύτερες αγορές και προσπαθώντας και διασφαλίζοντας ε, το ότι θα βρεθούμε στην πρωτολογία της χρήσης των σύγχρονων επικοινωνιακών τεχνολογιών, τότε θα μπορέσουμε να καταστήσουμε την αγορά μας τη μεγαλύτερη και την πιο δυναμική. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να είμαστε πολύ φιλόδοξοι. Στο σχέδιο έκθεσης που σας παρουσίασα, αλλά είχα και ευκαιρίες να συζητήσω πολλά θέματα με τους κοιόδης εισηγητές, θέλω να τονίσω κύριε Πρόεδρε ότι οι ευκαιρίες είναι πολύ καλές για να προχωρήσουμε μπροστά. Η κυρία Τράουτμαν υπογράμμισε πόσο σημαντικό είναι να επιτύχουμε υψηλή αποτελεσματικότητα στη χρήση του φάσματος, του ραδιοφάσματος. Ο κύριος Τσίτσεστερ τόνισε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν κάποιες χώρες, όχι μόνο το Ηνωμένο Βασίλειο, όλες οι χώρες που έχουν με τα, 100, με τα 700 θα πρέπει να έχουμε την καλύτερη δυναμικότητα και τις υψηλότερες ταχύτητες. Αυτά τα δύο συνδέονται και γενικώ με το πακέτο των τηλεπικοινωνιών. Πρέπει λοιπόν να εξασφαλίσουμε ότι θα λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα για να είμαστε οι καλύτεροι, γιατί εγώ δεν βλέπω καμία αντίφαση στις τρεις αυτές διαστάσεις, αυτές τις προοπτικές. Έθεσα λοιπόν το στόχο στην έκθεσή μου. Μέχρι το 2015 θα πρέπει να απελευθερώσουμε και να έχουμε 1200 MHz ε, για τη χρήση κινητών υπηρεσιών. Αυτό είναι γενικά αυτό που διεθνεί διεθνοί οργανισμοί τηλεπικοινωνιών λένε, ότι πρέπει να επιτύχουμε μέχρι το 2020. Όταν εμείς προσπαθήσουμε να το κάνουμε μέχρι το 2015, μπορούμε να προλιάνουμε το έδαφος και να είμαστε οι πρώτοι και όχι να έρθουμε δεύτεροι και τρίτοι. Αλλά στην έκθεσή μου τόνισα επίσης την ανάγκη να εντείνουμε την ε, διαδικασία όσο αφορά το πρώτο στάδιο, την απελευθέρωση ε, των 800 MHz. Να το κάνουμε αυτό μέχρι το 2013, έχω προτείνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ξέρω ότι κάποια κράτη-μέλη έχουν μεγαλύτερα προβλήματα, αντιμετωπίζουν μεγαλύτερα προβλήματα από άλλα. Ε, πιστεύω όμως ότι καλό είναι να διατηρήσουμε αυτή την ταχύτητα και να αναπτύξουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα μία συντονισμένη και ευρύτατη χρήση των συχνοτήτων γιατί έχει ζωτική σημασία αυτό για να αρπάξουμε την ευκαιρία και να βρεθούμε πρώτοι στις εξελίξεις. Να τονίσω για άλλη μια φορά κάτι. Όταν λέω να είμαστε στην πρωτοπορία, να είμαστε οι πρώτοι, αυτό δεν είναι και πολύ ε, αντιρεαλιστικός ή εξωπραγματικός ε, στόχος, γιατί η Ευρώπη είναι στην ε, πρωτοπορία, έχει προχωρήσει αρκετά την απορρίθμιση, την απελευθέρωση των τηλεπικοινωνιακών αγορών. Ε, κάπου χάσαμε αυτήν την ε, πρωτιά και νομίζω ότι πρέπει να την ξανακερδίσουμε. Νομίζω ότι αυτό το φάσμα, των, ε, αυτή η ζώνη των 800 MHz είναι ένας καλός στόχος. Νομίζω όμως ότι πρέπει να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα για να απελευθερώσουμε και το 1,5 γιατί αυτό θα μας επιτρέψει να εξασφαλίσουμε και τη δυναμικότητα αλλά και την ευκαιρία υψηλής ταχύτητας για ευρυζωνικές και κινητικές, κινητές υπηρεσίες, υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας και κινητού διαδικτύου. Ε, νομίζω ότι πρέπει να διανύμουμε και να χρησιμοποιήσουμε τις μη αδειοδοτούμενες υπηρεσίες, τις, αυτές που δεν έχουν ακόμη εκχωρηθεί ή παραχωρηθεί. Τα 56 Hz πρέπει επίσης πιστεύω να γίνει και μια καταγραφή από τα 300 στα 60, έτσι ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε στα 70 GHz. Και επίσης προτείνω τώρα να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να, να αναθεωρήσει και να κάνει ό,τι πρέπει να κάνει σε σχέση με τη ζώνη των 700. Γνωρίζω πολύ καλά τα προβλήματα που υπάρχουν, την ευαισθησία αυτού του τμήματος του ραδιοφάσματος και γι' αυτό προτείνω απλώς να έχουμε μια αναθεώρηση και, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει ό,τι είναι απαραίτητο, να λάβει τα πρόσφορα μέτρα. Και έτσι κύριε Πρόεδρε αυξάνουμε τις, επεκτείνουμε τις ε, φιλοδοξίες μας όσο αφορά την ευρωπαϊκή πολιτική για το φάσμα συχνοτήτων αλλά έτσι θα επιτρέψουμε στις ευρωπαϊκές τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες να αναπτυχθούν, αλλά ακόμα πιο σημαντικό, η ευρωπαϊκή βιομηχανία γενικά θα μπορέσει να είναι πρώτη σε όλες αυτές τις νέες εφαρμογές και υπηρεσίες, οι οποίες θα έχουν ζωτική σημασία για τις μελλοντικές αγορές. Και ταυτόχρονα ε, θέτουμε τα θεμέλια να εντάξουμε και πολιτιστικές και εμπορικές ε, εμπορικούς τομείς ε, στις νέες εφαρμογές και με μακροπρόθεσμο σχεδιασμό να διασφαλίσουμε ε, την, ραδιομετάδοση, την ασφαλή ραδιομετάδοση και να έχουμε και πρόσθετο εισόδημα για να καλύψουμε το κόστος των πληστηριασμών τμήματων του φάσματος. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να εντάξουμε, να ενσωματώσουμε στο σχέδιο, στο σώμα της έκθεσης, ε, τις απόψεις των σκιωδών εισηγητών. Σας ευχαριστώ πολύ και σας παρακαλώ τους επόμενους ομιλητές να περιοριστούν σε ένα λεπτό και να δώσω το λόγο στους σκιώδες. Καταρχάς, την κυρία Τράτμαν, ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. για να προσεγγίσουμε αυτό το πρώτο θέμα, νομίζω ότι δεν πρέπει να τα θέτουμε εδώ στο ίδιο καλάθι. Δηλαδή η ποσοτική συζήτηση δεν περιορίζεται μόνο στο θέμα των 700 MHz, αλλά πρέπει να θέσουμε και ένα θέμα ποιοτική διαχείριση του Ευρωπαϊκού Ραδιοφάσματο. Έτσι λοιπόν, θέλω να χαιρετήσω ε, το όραμα του εισηγητή. μερα φτάνουμε και στι πολύ ψηλέ συχνότητε ε, και από ό,τι φαίνεται, το μεγαλύτερο μέρο τη εκθεσή του φαίνεται να επικεντρώνεται στη ζώνη ENSF ε, σε ό,τι αφορά τα κινητά δεδομένα. Ε, Κανείς ε, δεν ε, αμφισβητεί τη διαπίστωση αυτή, αλλά ακόμη και αν θέλουμε να διαθέσουμε όλο το διαθέσιμο φάσμα στις ε, κινητές ζώνες, κάτι τέτοιο απλώς θα καθυστερούσε την κατάρρευση. Έτσι λοιπόν πρέπει να σκεφτούμε περισσότερες βάθος, λαμβάνοντα υπόψη τη συγκεκριμένη αρχιτεκτονική των δικτύων. Επίσης πρέπει να έχουμε μια ισότιμη προσέγγιση για την αποδοτικότητα του φάσματος και αυτός είναι ένας στόχος. Κανείς νομίζω δεν αμφισβητεί το ότι η επίγεια τηλεόραση είναι το πιο ε, κατάλληλο μέσο για να διαδώσουμε ε, από τον ένα στους πολλούς. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να έχουμε ένα καθολικό όραμα για τη συμπεριφορά των ε, χρηστών ε, και πρέπει να δούμε ποιες ανάγκες μπορεί να προκύψουν ακόμη και αν αλλάξουν χρήσεις. Θα πρέπει λοιπόν να καταρτήσουμε ένα κατάλογο, να αναλύσουμε συγκεκριμένα ε, το ε, ευρωπαϊκά, το, μάλλον το κοιτάσμα του ευρωπαϊκού φάσματος, η ζώνη ε, των 700 MHz ε, μέχρι τα 700 MHz ε, χρησιμοποιείται τώρα από τα κινητά, μπορούμε να την εκμεταλλευτούμε περαιτέρω. Θα ήθελα να ζητήσω από την Κομισιόν αν μπορεί να μας διευκρινίσει το θέμα αυτό. Τώρα στα 2 GHz ε, οι φορείς εκμετάλλευση. ήδη έχουν μεγάλη ποσότητα φάσματος, ε, χειρότερης αλλά μπορούν να το ξαναχρησιμοποιήσουν με πιο ε, αποτελεσματικές ε, ε, και νέες τεχνολογίες 3G και 4G αντί να παραμένουν στη 2G. Αν ε, είχε διατηρηθεί η αναλογική προσέγγιση, σήμερα δεν είχαμε περάσει στην ψηφιακή τεχνολογία. σε αυτή την καθολική προσέγγιση δεν μπορούμε να μα απαγορεύσουμε να συζητήσουμε τα 700 MHz, αλλά στο διεθνές πλαίσιο στο οποίο εξελισσόμαστε η παγκόσμια διάσκεψη του φάσματος του 2016 θα είναι αυτή που θα μπορούσε να προσδιορίσει ε, αυτή τη ζώνη για κάτι άλλο πέρα της ε, ε, ραδιοδιάδοσης. Θα πρέπει να μπορέσουμε να επιτρέψουμε στις πόλει να χρησιμοποιήσουμε χρησιμοποιούν τα δίκτυα στις επιχειρήσεις να αναπτύξουν νέες τεχνολογίες ε, για ε, την ε, κάλυψη υψηλού υψηλής χρέωσης και θα πρέπει να είναι δυνατόν να μπορούν να χρησιμοποιηθεί το φάσμα που δεν χρησιμοποιείται τώρα κατάλληλα. Λυπάμαι που ε, το κόστος για τη μετάβαση στο συστήματος ε, δεν ε, παρουσιάζεται με σαφήνεια, λαμβάνοντας υπόψη τις επενδύσεις που έχουν ήδη γίνει, είτε σε ό,τι αφορά την αλλαγή των decoders, των αποκωδικοποιητών ή των συσκευών ραδιομετάδοσης. Αυτή η συζήτηση δεν είναι μικρή. Ε, πρέπει να συζητήσουμε τους τρόπους κατανομής ε, του φάσματος, ε, δηλαδή σε σχέση και με τις άδειες, τις υποχρεώσεις των αδειών κτλ. Θα πρότεινα λοιπόν κάποιες προσαρμογές σε ό,τι αφορά τις άδειες της κινητής τηλεφωνίας, το RSPP, να παραμείνει στο πλαίσιο των γενικών επικοινωνιών και να συζητηθεί αυτό το θέμα με τι ρυθμιστικέ αρχέ. Αυτό σημείο δεν ήταν σαφέ στο κείμενο τη Κομισιόν. Επίση, λυπάμαι που το κείμενο τη Κομισιόν έχει κάποια κενά σε ό,τι αφορά τι πτυχέ εκτό ηλεκτρονική επικοινωνία. Γνωρίζουμε ότι πάρα πολλοί άλλοι τομεί ε, ε, μακρο... Ε, βραχυπρόθεσμα θα χρησιμοποιήσουν τι κινητέ τεχνολογίε ε, και θα πρέπει να διαφυλάξουμε μικρέ ποσότητε του φάσματο και για αυτέ τι καινοτόμε υπηρεσίε. Αυτές ε, τις παρατηρήσεις ήθελα να παρουσιάσω για τη συζήτηση αυτή. Θα προσπαθήσω να τις μεταφράσω και σε τροπολογίες και αύριο σας καλώ να παρευρεθείτε στην ακρόαση που οργανώνεται από την Ομάδα Σοσιαλιστών και Δημοκρατών όπου θα εμβαθύνουμε σε ορισμένα σημεία στα οποία αναφέρθηκα. Ο κύριος Ρούμπιχ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Χοϊκμάρτη γιατί έχω την εντύπωση ότι το θέμα αυτό το προχώρησε και το έθεσε ε, με πιο καταπήγοντα χαρακτήρα στην ευμερησία διάταξη, γιατί μιλάμε για τεχνολογίες τις οποίες μπορούμε να διαθέσουμε προκειμένου και στον τομέα αυτό να υπάρχουν θετικές εξελίξεις. Να προσέξουμε όμως και σε θέματα πληθυριασμών. Ποιοι είναι οι όροι που τίθενται. Και νομίζω ότι εδώ χρειάζεται ο κατάλογος απόδοσης ε, και σε ό,τι αφορά τα 27 κράτη-μέλη και τον υπόλοιπο ε, κόσμο. Να δούμε ποιοι όροι θα πρέπει να πληρώνται σε τέτοιο πληστηριασμό. Για να δούμε ποιες είναι οι θετικέ δυνατότητες και σε ό,τι αφορά τη συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κρατών μελών, η οποία θα πρέπει να είναι δεδομένη. Να σας υπενθυμίσω επίσης σε ό,τι αφορά στην τελική σκέψη 18, σε ό,τι αφορά την βοήθεια σε περίπτωση καταστροφών και ποιες είναι οι επιπρόσθετες συχνότητες ε, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για αυτή την ανακούφιση ε, από καταστροφές και στο άρθρο 7.3 στις, ε, στο έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Νομίζω ότι η διατύπωση είναι κάπως ασαφής. Νομίζω ότι οι υπηρεσίε τέτοιων οργανώσεων θα πρέπει πολύ απλά να έχουν προτεραιότητα. Και επίσης να υπάρχουν συνεργασίες μεταξύ των διαφόρων οργανώσεων σε αφορά θέματα διάσωσης, για παράδειγμα, σε περίπτωση καταστροφής, να υπάρχει δυνατότητα διάθεσης συχνοτήτων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρος, η κυρία Ρόλ. Thank um, Η κυρία Χόλ. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω και τον Ισογητή για το έργο του. Συνεργασία με τον κύριο Ρόντε από το Άλντε. Λείπουν πολλοί συνάδελφοι τη Άλντε γιατί είναι στην Κοπενχάγη. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξή. Να θέσω μάλλον διάφορα στοιχεία προς διευκρίνηση. Καταρχάς, σε ό,τι αφορά το, την προθεσμία για το 2013. Όντω μας προκαλεί ανησυχία σε κάποια κρατημέλη, μεταξύ άλλων και στον Εμένο Βασίλειο. Και το έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής λέει απλά ότι το τμήμα αυτό του φάσματος θα πρέπει να διατεθεί. Αυτό τι σημαίνει, ότι θα έπρεπε να έχει γίνει νέα κατανομή μέσω διαδικασίας πληστηριασμού ή ότι θα πρέπει να έχει ελευθερωθεί τα προηγούμενα χρόνια, γιατί μπορεί να υπάρχει εκ νέου κατανομή σε μετέπειτα χρονικό σημείο και ρωτιόμουν κατά πόσο θα μπορούσατε να μου το διευκρινίσετε αυτό. Δεύτερον, Μου άρεσε και μου προξένησε λίγο το ενδιαφέρον η τροπολογία 43 του εισηγητή. Ένα από τους πιο επικίνδυνους και περίεργους τομεί είναι πώς θα πάει το ευρυζωνικό δίκτυο στις ε, από μακρυμισμένες περιοχές. Αν ε, θα το ρυθμίσει αυτό η αγορά ή μήπως ε, θα πρέπει να υπάρχει πολιτική βούληση γιατί δεν θα αρκούν ε, οι κανόνες της αγοράς σε ό,τι αφορά τις ιεροκατοικημένες περιοχές και πώς μπορούμε να καθορίσουμε τη διάδραση μεταξύ αυτών των στοιχείων σε περίπτωση που θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε για παράδειγμα ότι θα προκύψει στρέβλωση στην αγορά. Θα ήθελα διευκρινήσεις αν θέλετε από τον εισηγητή και από την ε, Επιτροπή για το θέμα αυτό. Η Νίμπλε, ευχαριστώ. Πρόεδρε, θα ήθελα καταρχά να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Χέκμαρ, γιατί νομίζω ότι είναι πάρα πολύ έκθεση που μα υπέβαλε. Θα κάνω και εγώ φυσικά κάποιε τροπολογίε. Αλλά με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και με μεγάλη χαρά διάβασα την έκθεση σας κυρία Χόκμαρκ. Νομίζω ότι είναι ισορροπή η έκθεση. Τέσσερα σημεία θα ήθελα να αναφέρω, Πρόεδρε και κύριε Σιγητά, αγαπητοί συνάδελφοι. Καταρχάς, να συμφωνήσω με αυτά που είπε η συνάδελφο Τράουτμαν. Νομίζω ότι σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή πολιτική για το φάσμα, πολλά έχουμε σκεφτεί στο πακέτο για τις τηλεπικοινωνίες και εκεί προσπαθήσαμε να βρούμε μια ισορροπία μεταξύ πολιτισμικών και οικονομικών πτυχών σε ό,τι αφορά την πολιτική για το φάσμα. Νομίζω ότι κάθε μετέπειτα εξέλιξη της πολιτικής για το φάσμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να διασφαλίζει περαιτέρω αυτή την ισορροπία που ε, εξασφαλίσαμε και στο πακέτο για τις τηλεπικοινωνίες αυτό και σε ό,τι αφορά το πλαίσιο που διατυπώθηκε στο πακέτο για τις τηλεπικοινωνίες. Κατά δεύτερον, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να διασφαλίσουμε πέρα από τις διάφορες δυνατότητες σε ό,τι αφορά την ευρυζωνική ανάπτυξη και τις κινητές υπηρεσίες, να εξασφαλίζεται και το επίγειο φάσμα το οποίο θα πρέπει να διατηρήσει τις λειτουργίες τους. Αυτό θα πρέπει να διασφαλιστεί. Θα πρέπει να διασφαλιστεί η συνέχεια του φάσματος αυτού. Και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά κάτω από τα 790 MHz. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την παροχή των υπηρεσιών αυτό. Πρόκειται για μια σκέψη που διατύπωσε και η συνάδελφο Στράτσμαν. Τρίτο σημείο που θέλω να αναφέρω, κύριε Χόικμαρκ, είναι το θέμα του κόστους ε, μετανάστευσης μετάβασης. Και μιλάμε ήδη για το εύρος ε, κάτω από 800 MHz. Νομίζω ότι το κόστος μετάβασης ε, για τις συχνότητες αυτές θα πρέπει και αυτό να αναλυφθεί. Όσοι δηλαδή ε, ουσιαστικά έχουν τα πλεονεκτήματα από την απελευθέρωση του φάσματος αυτός θα πρέπει να επομιστούν και το κόστος. Και τέλος, αλλά νομίζω ότι αυτό αναφέρεται πάρα πολύ καλά ε, στην έκθεσή σας το θέμα της ε, των παρεμβολών. Νομίζω ότι ε, είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό. Θα πρέπει να κοιτάξουμε. Ενδεχομένω, ίσω να χρειαστεί να προσθέσουμε κάποια ζητήματα. Είναι σημαντικό πάντω και το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Τελκαστήγιο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν ε, να ευχαριστήσω τον κύριο Κόκμακ ε, για την εξαιρετική δουλειά του. Νομίζω ότι εδώ στην έκθεση τίθεται η Ευρωπαϊκή Ένωση σε ηγετική θέση σε σχέση ε, με το πώς μπορεί να καταστεί πρωταγωνιστική παγκοσμίω στα πλαίσια υποδομών. Και μάλιστα μας παρουσιάζεται όλο αυτό το θέμα μακροπρόθεσμα ε, και μεσοπρόθεσμα. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που προσπαθήσατε να λάβετε υπόψη και τα διάφορα συμφέροντα των ε, θυγόμενων τομέων αλλά και όλων των ε, πολιτικών ομάδων. Θα πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια ε, έτσι ώστε βασικά αυτή είναι η θέση του Κοινοβουλίου. Θα προκύψουν προβλήματα πιθανότητα από διαπραγμάτευση με το Συμβούλιο και εκεί είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε μια ισχυρή και ενία θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έτσι λοιπόν εγώ στην παρέμβαση αυτή ε, θέλω να πω τα εξή, υπάρχουν ορισμένα θέματα που μπορούν να θυκθούν. Βέβαια θα προσιάσω κάποιε τροπολογίες για να το πράξω αυτό. Πιστεύω ότι το σημερινό μήνυμα είναι ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να έχει μια θέση ομόφωνη, αν μπορεί να είναι τόσο το καλύτερο, γιατί τα προβλήματα θα προκύψουν στι διαπραγματεύσει με το Συμβούλιο και νομίζω ότι βρισκόμαστε ενώπιον ενό μέσου δηλαδή για το ραδιόφασμα και τη διεύρυνση του ραδιοφάσματος ε, ε, που θίγει ε, πάρα πολλούς τομείς και είναι ζωτική σημασίας. Έτσι λοιπόν το μήνυμά μου σήμερα θα είναι να διατηρήσουμε ως το τέλος, ως την Ολομέλεια, μία ενιαία θέση. Όλες οι πολιτικές ομάδες πρέπει να επιδείξουν ενότητα. Μάλιστα και τώρα να δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για λίγο. Thank you, Mr. Chairman. And very brief. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Με λίγα λόγια θα ήθελα να χαιρετήσω αυτό το σχέδιο έκθεσης εκ μέρους της Επιτροπής. Είναι μια πολύ καλή βάση εργασίας. Νομίζω ότι πολλά σημαντικά θέματα τέθηκαν. Η Ευρωπαϊκή Τροπή είναι πάντοτε διαθέσιμη να εξηγήσει προς τα κράτη-μέλη και τους βουλευτές τα τεχνικά ζητήματα που χρήζουν διευκρινήσεων και διασαφηνήσεων, να διοργανώσει ακροάσεις, ε, συζητήσεις και κοινέ συνεδριάσεις. Εν, εν συντομία τώρα, σε σχέση με τα ζητήματα που απευθύνονται στην Επιτροπή. Ε, καταρχήν τα θέματα που έθεσε η κυρία Τράουτμαν. για τη γεωργία. Θα πρέπει να παραμείνουμε σε ανταγωνιστική θέση και να μην εμποδίζονται, να μην εμποδίζεται η ανάπτυξη αυτών των πολύ σημαντικών ε, υπηρεσιών. Ε, η διαχείριση της ε, ζώνης ε, των MHz είναι πάρα πολύ σημαντική. Εάν μπορέσουμε μέχρι το 2013 να το πετύχουμε, να έχουμε μεγαλύτερο φάσμα και να μπορέσουμε να διεξάγουμε μεγαλύτερες επιχειρήσεις και πιο υψηλότατες ταχύτητες θα ήταν πολύ κακό. Πολύ ορθώς τονίστηκε η σημασία των ε, ραδιοσυχνοτήτων ε, των ε, επίγουσας φύσης, έκτακτης φύσης. Έχουμε χρησιμοποιήσει τη φράση στην οποία αναφέρθηκε όπου αυτό είναι απαραίτητο, γιατί αυτό είναι ένας τομέας που έχουμε από κοινού αρμοδιότητα με τα κράτη-μέλη και προσπαθούμε να συνεργαστούμε με τα κράτη-μέλη να απαντήσουμε στο ζήτημα αυτό. Όσο αφορά το ερώτημα της κυρίας Χόλτς, για την προθεσμία του 2013, αλλά και την τροπολογία 43. Πράγματι, πρέπει να δούμε πολύ προσεκτικά πώς εφαρμόζουμε την τεχνολογία με ουδετερότητα, έτσι ώστε οι υπηρεσίες να παρέχονται και στις αγροτικές υπηρεσίες, ε, να παρέχεται η καλύτερη και η υψηλότερη δυνατή ταχύτητα εκεί όπου δεν πρόκειται να επεκτεθούν τα χερσαία δίκτυα ή δεν θα παρέχονται εναλλακτικέ υπηρεσίες στους πολίτες. Τέλος, πολλοί ομιλητές μίλησαν για ισορροπία. Φυσικά η Επιτροπή ελπίζει ότι επέτυχε την ισορροπία μεταξύ των διαφορετικών συμφερόντων. Ε, ε, αυτό δεν είναι μόνο ε, ραδιοτηλεοπτική μετάδοση έναντι της ευρυζενικότητας. Δεν είναι μόνο αυτό. Προτείνουμε και μια απογραφή. Θέλουμε και άλλοι να χρησιμοποιήσουν αυτή την απογραφή. Θέλουμε μια αντικειμενική ανάλυση και καταγραφή του πού υπάρχει φάσμα, πού χρησιμοποιείται. Και θα πρέπει η Επιτροπή και τα κράτη-μέλη να βρουν την πιο αποδοτική και αποτελεσματική χρήση του φάσματος για όλους αυτούς τους χρήστες και να ενθερρυνθούν τα κράτη-μέλη στην αδειοδότηση και στην, ε, στον επιμερισμό των ραδιοσυχνοτήτων ανάλογα με τις ε, εθνικές ιδιομορφίες. Για μια φορά ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Περότε, ευχαριστώ και τον εισηγητή. Σας ευχαριστώ και να ρωτήσω μήπως θέλει ο Γκούνταρ να πάρει το λόγο, κύριε Σιγητά. Uh, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και όλους ε, τους συναδελφούς για τις ε, διάφορες παρεμβάσεις και τις απόψεις που καταδέχθηκαν εδώ. Δεν βλέπω να υπάρχει κάποιο μεγάλο πρόβλημα ή κάποιο επίμαχο σημείο να προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε μια νέα θέση βάσει όσων ακούστηκαν σήμερα. Και αν ξεκινήσουμε με το πρόβλημα σχετικά με το πώς θα έχουμε τις καλύτερες ευκαιρίες στην Ευρώπη, τότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε διαφορετικού τρόπου και μέσα και να διασφαλίσουμε ότι μπορούμε να εξορροπήσουμε τα διάφορα συμφέροντα. Σω θα θα έπρεπε να προσπαθήσουμε να βοηθήσει ο ένα τον άλλο, δηλαδή να μην δούμε τι κάναμε πριν 5-10 χρόνια, αλλά τι θα γίνει για τα επόμενα 5 έτη. Νομίζω ο κύριο Ρίμπη το είπε ότι είναι πολύ γρήγορη η αλλαγή και νομίζω ότι οι αλλαγέ τα επόμενα πέντε έτη θα είναι πολύ πιο ταχύ από όσα είδαμε τα προηγούμενα πέντε έτη. Και Κατά τη δική μου άποψη, θα έχουμε καλύτερες ευκαιρίες ε, να διασφαλίσουμε ε, τις ε, υπηρεσίες ε, καλύτερα στο μέλλον σε σχέση με σήμερα και αναφέρομαι και στην ψηφιακή επίγεια τηλεόραση και στην ε, ραδιοτηλεοπτική μετάδοση. Θα πρέπει να έχουμε επαρκές φάσμα για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε και τις νέες τεχνολογίες. Γιατί ούτως ή άλλως αυτό θα γίνει, αυτό θα συμβεί. Σε ό,τι αφορά τώρα τα ερωτήματα της κυρίας Χολ. Νομίζω καταρχήν είναι σημαντικό να προσπαθήσουμε να είμαστε κάθετοι σε ό,τι φορά το στόχο του 2013. Ξέρω ότι ορισμένα κρατημέλη έχουν μεγαλύτερα προβλήματα από άλλα, αλλά ενίοτε πιστεύω ότι χρειάζεται να διασφαλίσουμε ότι και όσοι καθυστερούν να ξεκινήσουν το συντομότερο, σε ό,τι φορά την κάλυψη. Προτείνω στην τροπολογία μου στην οποία αναφερθήκατε κυρία Χόλ, ότι θα πρέπει να έχουμε ουδετερότητα από τη σκοπιά της τεχνολογίας, γιατί πρέπει να έχουμε την υποχρέωση και τη συνθήκη για τους ε, ε, operator να έχουν πλήρη κάλυψη. Τώρα όμως το πώς θα λυθεί αυτό το θέμα μπορεί να διαφέρει στις μεγάλες πόλεις ε, από τις λύσεις που θα χρησιμοποιηθούν στις αγροτικές περιοχές. Παραδείγματο χάρη, αν ε, πάρω ένα παράδειγμα από τη δική μου χώρα, ε, μπορεί να έχουμε διαφορετικού τρόπου στο Χόλμη και διαφορετικού τρόπου στο Βορρά, αλλά το θέμα είναι να ξεύρουμε λύσει. Και σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη της αποδοτικότητας, νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε όλες τις ευκαιρίες και όλες τις τεχνολογίες για να διασφαλίσουμε ότι χρησιμοποιούμε όσο το δυνατόν καλύτερα το διαθέσιμο φάσμα αλλά και σε ό,τι αφορά το κόστος ε, της ε, μετάβασης, να προσπαθήσουμε να καλύψουμε αυτό το κόστος από τα χρήματα που θα λαμβάνουμε από τους πληστηριασμούς. Τώρα, το πώς θα γίνει αυτό, καλύτερα είναι να το αναλάβουν αυτό τα κρατη και εθνικές ρυθμιστικές αρχές. Έτσι μπορούμε να διασφαλίσουμε την καλύτερη ισορροπία, γιατί υπάρχουν ε, διάφορες προϋποθέσεις, διαφορετικές προϋποθέσεις σε διάφορες χώρες. Ορισμένα κράτη-μέλη έχουν πολλή τηλεόραση ορισμένα σημεία του φάσματος, ενώ κάποια άλλα όχι και νομίζω ότι καλό να είναι να έχουμε λύσεις ρεαλιστικές σε επίπεδο κράτους μέλους. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ανυπομονώ να λάβω τις τροπολογίες και σας ευχαριστώ για όλα όσα ακούστηκαν εδώ σήμερα. Να σας ευχαριστήσω και εγώ και να υποδείξω το εξής. Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών είναι η 9η Μαρτίου στις 12 η ώρα μεσημέρι. Ωραία λοιπόν και περνάμε τώρα στο 5 6 και 7 στις ψηφοφορίες. Ηλεκτρονικές ψηφοφορίες. Ελπίζω να έχετε όλες τις κάρτες μαζί σας, προκειμένου να ολοκληρώσουμε γρήγορα τις ψηφοφορίες, γιατί έχουμε... Διακοπή πρόεδρος. <laughs> We will, we will see. Hello. So, können wir loslegen? Ξεκινάμε λοιπόν. Είσαστε όλοι έτοιμοι. Also, erster Punkt αυτό το θέμα. Η Ευρώπη είναι ο πρώτο τουριστικό προορισμό στον κόσμο. Με αυτό το θέμα θα ξεκινήσουμε σήμερα. Ένα νέο πλαίσιο πολιτική για τον ευρωπαϊκό τουρισμό. Ο, του συναδέλφου Χατζημαρκάκη. Και ξεκινάμε με τη συμβαστική 1. Υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Στο 5. Περνάμε στην τραπολογία 5. Υπέρ. Κατά. απόχέ. Ε, εγκρίνεται. Συμβαστική 2. Υπέρ. Κατά. άποχέ. Εγκρίνεται. Στην 11. Υπέρ. Κατά. Αποχέ, Εγκρίνεται. 13. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 18. Υπέρ υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 19 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 21 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ, κατά, άποχες, εγκρίνεται. 29 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 31 υπέρ. Αποσύρεται, αποσύρεται 27. Η 31 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται 32 υπέρ. Κατά. Ξανά θα θέλετε για την 32 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Σεμιβαστική 5 με προφορική τροπολογία. Τη γνωρίζετε, χρειάζεται να τη διαβάσουμε. Η κυρία Τράτμαν θέλει να τη διαβάσει. Ε, Θα ήθελα να, με τη συμφωνία του εισηγητή να προτείνει social tourism. Εκεί στη λέξη έρητας να προσθέσουμε το social tourism μετά δηλαδή το θέμα του πολιτισμού να προσταθεί και ο, ο κοινωνικός τουρισμός υπέρ. Για την συμβαστική 5 παρακαλώ. Ξανά. Ξανά. Για τη συμβαστική 5 με την προφορική τροπολογία. Ποιος είναι υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 37 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 38 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 39 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και τώρα περνάμε στις 48 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 49 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Περνάμε λοιπόν στην 50 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 54 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 56 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 58 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 61 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά έναρξη ψηφοφορίας παρακαλώ. And can we close? Noch eine Minute. Άλλο λίγο. Closed. Λήξη. Ωραία. Δεν λειτουργεί κάτι. Εντάξει. Θέλει άλλο ένα να ψηφίσει υπέρ, αλλά εν πάση περιπτώσει ε, νομίζω ότι με στριπτική πλειοψηφία εγκρίνεται η έκθεση, να συγχαρούμε όλους τους εισηγητές. Σχεδόν ομόφωνα εγκρίνεται η έκθεση και περνάμε στο 6 τώρα. Αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα της χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα του παραπλησμού πυρηνικών σταθμών στα νέα κράτη-μέλη. Του κ. Μπαλτσίτης. Έχετε μπροστά σας τα έγγραφα. Περνάμε στην ψηφοφορία κατευθείαν. Στην 5 παρακαλώ υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 7 υπέρ. Να το ελέγξουμε. Ωραία. έχουμε την 6. Παρακαλώ ηλεκτρονικά. Ηλεκτρονικά την 6. Ε- Έναξη ψηφορίας. Για την 6. Number 6. Open. EPP, I uh, want to watch. Έχουμε έναν που περισσεύει από το ΕΛΚ πάντα τα ίδια. Ο κ. Κάλφιν δεν έχει κάρτα, μάλιστα. Πέρα τη ε, ψηφοφορία 16, υπέρ 22 κατά, ο κ. Κάλφιν. Υπέρ 16, 17 λοιπόν και 22. Και πάλι. Απορρίπτεται, 7. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Η 10 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Α, καταπίπτει αλλά και απορρίπτεται. Ωραία, πάμε στην 8. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Στην εννέα. Και αυτό στα δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Στη δώδεκα Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές και αυτό απορρίπτεται. Στη 13 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 11. Ως προσθήκη υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 14 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται 16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται 17 υπέρ. Α, μισό λεπτό. Καταπληκτή, καταπληκτή. Ωραία, πάμε στην 18 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται 20 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται 19 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 21 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 22 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 23 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 1 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η δύο, Η... Α, Οι Η τρία σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται και περνάμε στην τελική ψηφοφορία. Ηλεκτρονικά παρακαλώ. έναξη ψηφοφορίας. One one too much, please. Πάλι περισσεύει ένας από το ΕΛΚ. Okay, and closed. Πέρασε. Κύριε Κάλφιν, εντάξει, ωραία. 39 ψήφοι υπέρ. Συγχαρητήρια, εγκρίνεται η έκθεση και περνάμε τώρα στο επόμενο θέμα, στο 7, μία ενιαία αγορά για τις επιχειρήσεις και την ανάπτυξη. Έχετε τα στοιχεία μπροστά σας και περνάμε στην τροπολογία 1, υπέρ. Κατά αποχές συγκρίνεται. Συμβαστική 1 υπέρ, κατά, απόχέ εγκρίνεται. 5 υπέρ, κατά, Αποχέ. εγκρίνεται. Για την 5 ξανά αν θέλετε παρακαλώ, υπέρ, κατά, απόχέ εγκρίνεται. Η 6 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 2 υπέρ, κατά, Αποχέ εγκρίνεται. Η 7 Υπέρ. Α, συγγνώμη, καταπίπτει. Συγγνώμη, συγγνώμη, συγγνώμη. Στην 9 πάμε, στην 9. Υπέρ. Κατά. Αποχέ, Απορρίπτεται. Στην 10. Υπέρ. Κατά. άποχέ, Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχέ, Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Στην 22 πάμε υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 24 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται. Ναι, να το ελέγξουμε, να ελέγξουμε την 24 παρακαλώ, γιατί είναι λίγο σαφές. Είναι λίγο οριακά. Yeah, Πέρασε. Εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 27 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 28 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 30 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 31 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 32 υπέρ. Κατά. Να το ελέγξουμε παρακαλώ αν θέλετε για την 32 ηλεκτρονικά έναξη ψηφοφορίας. Oh, Closed. Πέρας. Εγκρίνεται. 33 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται και περνάμε τώρα στην τελική ψηφοφορία. Έναρξη ψηφοφορίας παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται λοιπόν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και περνάμε λοιπόν στο επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη στο 8. Έχουμε και άλλους τρεις φυσικά γιατί έχουν τον κύριο Ταγιάννη ο οποίος θα έρθει σύντομα αλλά εν πάση περιπτώσει θα τα ε, προλάβουμε. Όχι, δεν έχουμε στρες που θα έρθει και Γιάννη, έχουμε στρες που έχουν πολλά πράγματα. Έχουμε λοιπόν στο 8 την Ένωση κεντομία μεταμορφώνοντα την Ευρώπη για ένα κόσμο μετά την κρίση. Η συνάδελφο Μέρκη έχει το λόγο και θα είναι και η μοναδική που θα πάρει το λόγο. Αν θα μπορούσαν όμω οι συνάδελφοι να κάνουν ησυχία. Μα τι, τι σα δυσκολεύεται μπορώ να καταλάβω. Βγείτε έξω να συζητήσετε. Κυρίε και κύριοι κυρία Μέρκης έχει το λόγο. Um, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν, θέλω να ευχαριστήσω όλους ε, τους συναδέλφους για την εξαιρετική τους ε, συνεργασία και τη συνεισφορά τους. Είναι σαφές ότι η κοινοτομία αποτελεί μέγιστη προτεραιότητα στο Κοινοβούλιο και για πολλούς από τους ε, συναδέλφους μας και ορθώς γιατί πιστεύω ότι η καινοτομία αποτελεί τη μεγάλη πρόκληση, την μηχανή της Ευρώπης αυτή τη στιγμή. Έτσι λοιπόν, ποια είναι τα κυρία σημεία της έκθεσης αυτής. Ε, πιστεύω ότι το πλέον σημαντικό για την καινοτομία είναι η εστίαση αν μπορώ να το συγκρίνω αυτό με το εξή, αν ε, πείτε ότι έχουμε ε, προκλήσεις στην Ευρώπη, αυτό ισχύει, αλλά έχουμε κοινέ προκλήσεις και θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτές τις κοινέ προκλήσεις. Αν μπορώ να το συγκρίνω αυτό, αν έχουμε ένα σπίτι που καίγεται, παραδείγματο χάρη, ε, δεν θα πάτε να ποτίσετε τα φυτά στο κήπο, αλλά θα χρησιμοποιήσετε το νερό για να σβήσετε τη φωτιά. Και ε, τι γίνεται τώρα με τα σπίτια που έχουν φτιάσει φωτιά αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτά και να τα περιορίσουμε. Βασικά, θα έλεγα ότι έχουμε τρεις ε, κύριες ε, κοινωνικές προκλήσεις, αλλά είναι μόνο τρεις. Η μία είναι η δημογραφική αλλαγή, η γύρανση του πληθυσμού, αστικοποίηση και μεταναστευτικές ροές και... Αυτό αποτελεί την ε, κύρια πρόκληση την κοινωνική. Αν δείτε όλα αυτά τα θέματα έχουμε ένα κοινό παρανομαστή. Αυτό είναι το πρώτο λοιπόν. Το δεύτερο είναι η βιώσιμη διαχείριση των πόρων προκειμένου να μειώσουμε την εξάρτησή μας ε, για την εισρωή ε, νέων ε, πρώτων υλών. Πρέπει να επικεντρωθούμε στην λειψιδρία, στην φοδιασμό των υδάτων, στι πλημμύρε και στην ξηρεσία στην Ευρώπη και πώς θα έχουμε πρώτες ύλες στην Ευρώπη και τρίτον μία ισότιμη και σταθερή οικονομική βάση για το πώς να εξέλθουμε από την οικονομική κρίση, πώς να έχουμε μία κοινωνία που θα βασίζεται στη γνώση και θα προωθεί την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτές είναι οι κυρίες ε, Τρει κυρίε κοινωνικέ προκλήσεις που βλέπω και καλώ στην έκθεση για μια καθολική ολιστική προσέγγιση. Δηλαδή αν αυτά είναι τα τρία κεγόμενα, φλεγόμενα σπίτια θα πρέπει να σβήσουμε τη φωτιά σε όλους τους τομείς πολιτικής ε, μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν μπορούμε να επικεντρωθούμε στις μικρότερες προκλήσει αν έχουμε αυτέ τι ε, τρει. Ε, κύριες ε, κοινωνικές προκλήσεις ενωπιών μας. Πώς θα το πράξουμε λοιπόν αυτό. Νομίζω ότι το κλειδί για να προωθήσουμε την καινοτομία έγκυται σε μια καλή συνεργασία. Και νομίζουμε ότι μέχρι τώρα έχουμε ξεχάσει ένα πολύ σημαντικό παράγοντα, δηλαδή τον πολίτη. Συνήθως ε, χρησιμοποιούμε για το μιλάμε για το τρίγωνο κυβερνήσεις, ε, ερευνητικοί οργανισμοί και επιχειρήσεις. Αλλά νομίζω ότι ο πολίτης με την κατανάλωσή του ή με τη συμπεριφορά του είναι αυτός που αποτελεί τον παράγοντα που κινεί ε, την καινοτομία και η δημιουργικότητα του πολίτη θα φέρει την αλλαγή. Αν επικεντρωθούμε στον πολίτη προκύπτει ένα διαφορετικό μοντέλο γιατί οι ίδιοι οι πολίτες ε, είναι καινοτόμοι και περιγράφω κάτι τέτοιο στην έκθεση. Είδαμε ότι μέχρι σήμερα έχουμε επικεντρωθεί τα μάλα στην τεχνολογία και στα προϊόντα. Αλλά η καινοτομία μπορεί να ε, αποτελεί κάτι πολύ περισσότερο. Μπορεί να μιλάμε και για μια διαδικασία κοινωνική καινοτομία. Ένα προϊόν μπορεί να είναι ένα προϊόν, μπορεί να είναι μια υπηρεσία, αλλά και ένα κίνημα. Τι είναι, τι είναι αυτό το κίνημα, ακριβώ αυτό δηλαδή. Θα βλέπουμε τον πολίτη ω ε, παράγοντα καινοτομία. Αν δείτε το Facebook, παραδείγματο χάρη, αυτό αποτελεί ένα κίνημα και δεν μπορεί να περιγραφεί με κανέναν άλλο τρόπο. Πού επικεντρώνομαι λοιπόν εγώ σε αυτή την έκθεση στους ε, πολίτες, δίνεται στήσεις αυτές τις ε, τρεις κοινωνικές προκλήσεις και στην πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Η πρόσβαση στη χρηματοδότηση είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για όλες τις επιχειρήσεις και για τα επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα, αλλά και για τι μικρέ και μεσέ επιχειρήσεις. Και νομίζω ότι πρέπει να επεκτείνουμε το επίπεδο υπηρεσιών μας, δηλαδή από την ενία θηρίδα, ε, να προχωρήσουμε γιατί οι, επιχειρή... μικρές και μεσέ επιχειρήσεις δεν έχουν χρόνο τη νύχτα να μελετήσουν όλους τους κανονισμού που θα ζητήσουν χρηματοδότηση, εγγύσει και πρέπει να παρέχονται κάποιε υπηρεσίε. Αν θέλουμε να διευκολύνουμε λοιπόν την καινοτομία, πρέπει να διευκολύνουμε την πρόσβαση στη χρηματοδότηση και πρέπει να παράσχουμε και υπηρεσίε στην Ένωση τη Καινοτομία. Έτσι λοιπόν, ένα θέμα είναι ότι έχουμε πάρα πολλά νομοθετήματα και πρέπει να επικεντρωθούμε στη χρηματοδότηση, ε, δηλαδή στην χορήγηση ε, επιδοτήσεων ε, αντί κεφαλαίων κεφαλαίου επιχειρηματικού κινδύνου. Ε, έτσι λοιπόν πρέπει να επικεντρωθούμε και στη χρηματοδότηση. Πρέπει να προσπαθήσουμε να συγχωνεύσουμε πολλά από αυτά τα νομοθετήματα ή τα προγράμματα ή τα επιδοτήσει όπως θέλετε να τα αποκαλέσετε όλα αυτά. Να υπάρχει εμπειρογνωμοσύνη, να παράσχεται στήριξη είτε μέσω ε, ενός νομοθετήματος ή ενός, ε, μιας επιδότησης για να προωθήσουμε την κοινοτομία. Νομίζω ότι συνήθως οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν είναι αυτοί ε, που έχουν την πλήρη κατανόηση όλης αυτής της διαδικασίας. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να βρούμε έναν καλύτερο τρόπο που να βασίζεται στην εμπειρογνωμοσύνη για να παράσχουμε αυτή τη στήριξη. και για να εμπλέξουμε κυρίως τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Κάτι τελευταίο, νομίζω ότι η κοινωνική καινοτομία είναι πάρα πολύ σημαντική. Απλώς έχουμε το ερώτημα σε τι συνίσταται η κοινωνική καινοτομία. Δεν αποτελεί τίποτα περισσότερο, ούτε τίποτα λιγότερο η κοινωνική καινοτομία ε, στο να ανοίξει η δυνατότητα για όλους να αλλάξουν το περιβάλλον τους. Και όταν λέω περιβάλλον δεν το εννοώ με την οικολογική έννοια και μόνο δηλαδή οι εργαζόμενοι να επηρεάσουν στο χώρο εργασία. οι πολίτες να επηρεάσουν στην κοινωνία, οι επιχειρήσεις να επηρεάσουν ε, το επιχειρησιακό τους περιβάλλον. Δηλαδή επικεντρωνόμαστε ε, στους ανθρώπους να μπορέσουν να επηρεάσουν το χώρο που εργάζονται. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να προσπαθήσουμε να προωθήσουμε την καινοτομία. Αυτό αποτελεί αποτέλεσμα εστίασης και αναρωτιέμαι αν χρειάζεται να συστήσουμε πολλά διαφορετικά προγράμματα για να προωθήσουμε την καινοτομία, γιατί αυτή η προώθηση μπορεί να γίνει ήδη μέσω της εστίασης. Υπάρχει και ένα θέμα για τα πρότυπα, για την τυποποίηση. Ευχαρίστω να το συζητήσω. Και φυσικά μιλάμε και για την ενιαία αγορά. Μόλις ε, ολοκληρώθηκε η ψηφορία για το θέμα αυτό, γιατί το άνοιγμα τη ενιαία αγορά δημιουργεί αυτή τη μεγάλη αγορά για τα καινοτόμα προϊόντα και τις υπηρεσίε. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω ότι πολλά πρέπει να γίνουν ακόμη. Εγώ στην εκθεσή μου έχω αναφερθεί και στο άνοιγμα αυτών των αγορών, ε, τις οποίες δεν συζητήσαμε για τα προϊόντα υγείας, παραδείγματος χάρη, γιατί σχετίζεται πάρα πολύ στενά και φυσικά οι δημόσιες προμήθειες είναι ένας τρόπος να προωθήσουμε την καινοτομία και να έχουμε έναν υπεύθυνο ρόλο ως κυβέρνηση και φυσικά και οι περιφέρειες είναι πολύ σημαντικός εταίρος σε επίπεδο διακυβέρνησης γιατί βρίσκονται πάρα πολύ κοντά στις μικρές και μεσές επιχειρήσεις, ε, στον πολίτη και στα ερευνητικά ιδρύματα. Σας ευχαριστώ και σας ευχαριστώ ήδη για όλες σας τις συνεισφορές. Ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί σας για την εκθέση αυτή στο μέλλον. Σας ευχαριστώ, συνάδελφος Σατούρη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν, ευχαριστώ τη συνάδελφο Μέρκης, η οποία πραγματικά κάνει πολύ καλή δουλειά ε, στην σύνταξη αυτής της έκθεσης. Θέλω να τονίσω επίσης την τεράστια σημασία της, αν και αυτή τη στιγμή είναι πολύ γενική φύσεως. Νομίζω ότι η πρόταση της κυρίας Μέρκη καλύπτει εν μέρη το κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπή. Εν μέρη όμως ε, προσφέρει καινούργιε προσογγίσεις, ιδίως όσο αφορά την πρόσβαση στα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά μέσα, ένα ζήτημα εξαιρετικής σημασίας, αλλά δίδει και έμφαση στο θέμα τη κοινωνική καινοτομία. Εξάλλου, με μεγάλη προσοχή ε, επαναλαμβάνει μια αντίληψη που είναι πάρα πολύ σημαντική, την, την εγκάρσια φύση αυτών των πραγμάτων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό όταν μιλάμε για καινοτομία. Η καινοτομία πρέπει να διασχίζει εγκάρσια όλους τους τομείς ε, ε, εργασίας και δραστηριότητας. Σημερίζομαι επίσης την προσοχή που έχει αποδώσει η κυρία Μέρκης στην κεντρική θέση που πρέπει να καταλαμβάνει ο άνθρωπος, το άτομο. Ε, βέβαια, εδώ επισέρχονται μια σειρά παράγοντες. Πάνω ε, παράγοντες οι οποίοι χρήζουν, θεωρώ, κάποιων προσθήκων. Πρέπει να προσθέσουμε πράγματα δηλαδή. Νομίζω ότι ο ρόλος των επιχειρήσεων πρέπει να προσεχθεί περισσότερο και εξηγούμε. Ε, μέχρι στιγμής σίγουρα η επιχείρηση εμφανιζόταν στο προσκήνιο όταν μιλούσαμε για καινοτομία. Ωστόσο, ε, χωρίς να θέλω να αφαιρέσω ε, ισχύ από το επιχείρημα που τοποθετεί το άτομο στο κέντρο της προσέγγισης μας, δεν μπορώ παρά να επαναλάβω πόσο σημαντική είναι η κεντρική θέση της επιχείρησης. Δεύτερον, υπάρχει το θέμα της επικοινωνίας. Και εδώ, σε αυτόν τον τομέα, όπως σε τόσους άλλους τομείς, η επικοινωνία είναι βασική, θεμελιώδης, γιατί όπως ξέρουμε όλοι υπάρχει δυσκολία κοινωνίας της δουλειάς που κάνουμε προς τα έξω. Όταν γίνεται λόγος για καινοτομία, είναι σημαντικό όσο το δυνατόν περισσότεροι να, να μάθουν ποιες καινοτόμες διαδικασίες και διεργασίες υπάρχουν. Και νομίζω ότι εδώ είμαστε προβληματικοί στο θέμα της επικοινωνίας. Για μένα έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό το θέμα. Ωστόσο, δίπλα σε αυτό θέτω και το ζήτημα όλων των διοικητικών διαδικασιών. Ναι, είναι σημαντική η επικοινωνία προς, το έξω, προς τα έξω, αλλά σημαντικό είναι να, αναθεωρούν, να αναθεωρηθούν οι διοικητικές διαδικασίες για να απελευθερωθούν πόροι. Άλλο ζήτημα. Συμφωνώ απόλυτα ε, για τη σημασία της συνεργασίας με τις περιφέρειες και τα κράτη-μέλη. Υπάρχει αυτή η συνεργασία, πρέπει όμως να ενταθεί. Όμως σήμαση, ε, προσοχή, έχουμε υπερβολικά πολλά σημεία εξυπηρέτησης, θηρίδες. Ε, όταν φανταζόμαστε τη συνεργασία μας, πρέπει να ε, να το φανταστούμε, να περνάει η συνεργασία αυτή μέσα από τα υπάρχοντα κανάλια ή θα πρέπει να σκεφτούμε πώς θα υποκαταστήσουμε αυτά τα κανάλια. Κύριε Πρόεδρε, επίσης θέλω να πω τα εξής. Θα ήθελα να συμπεριληφθούν στον προβληματισμό κάποια θέματα τα οποία, για τα οποία έχει πρωτοστατήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρώτον είναι η υιοθέτηση το 2011 ένα ευρωπαϊκό πιλωτικό ε, πρόγραμμα για την κοινωνική καινοτομία από τη μία πλευρά και να ενεργοποιηθεί ένα νέο ερευνητικό πρόγραμμα στον τομέα της κοινωνικής καινοτομίας. Θεωρώ ότι η πρόταση αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανταποκρίνεται στις προσδοκίες που εξέφρασε η κυρία Μέρκης με την πρότασή της. Δηλαδή αυτό δείχνει τη στήριξη που θα δοθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο ζήτημα αυτό. Τέλος, το ερευνητικό πρόγραμμα για την καινοτομία θα πρέπει να εφαρμοστεί στη δημόσια διοίκηση. Αυτό το ζήτημα έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί βρίσκεται στη βάση πολλών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η διοίκηση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Πέντε άτομα έχουν στήσει το λόγο, αλλά να σας ε, πω ότι δεν μπορείτε να μιλήσετε πάνω από δύο λεπτά. Δεν θα καταφέρουμε άλλος ή άλλος να μιλήσουν όλοι. Ο Πολ ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να χαρώ την ε, εισηγήτρια σε ό,τι αφορά την καινοτομία, γιατί αυτή αποτελεί τη βάση για τις νέες θέσεις εργασίας και μάλιστα τις πιο καλοπληρωμένες. Και θα πρέπει να κοιτάξουμε λοιπόν πώς ε, οι υποδομές στο μέλλον μπορούν να αναπτυχθούν με καλύτερο τρόπο. Και νομίζω ότι με, την, με τον προπολογισμό για τη γεωργία και την ε, περιφερειακή ανάπτυξη θα καταφέρουμε να βελτιώσουμε τους τομείς και τις υποδομές σε θέματα τροφίμων κτλ. Για να λάβει σε ευρωπαϊκό επίπεδο μια ευρωπαϊκή διάσταση, αν θέλετε, η περιφερειακή ανάπτυξη και να εφαρμοστεί αντίστοιχα να εφαρμοστούν όλα τα προγράμματα σε υπηρεσίες και υποδομής. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος ο συνάδελφος um, Ευχαριστώ. Η έκθεση αυτή για την ε, Ένωση καινοτομία. έχει μία στερεά βάση και ορθώς εντοπίζει ότι η καινοτομία είναι απαραίτητη όχι μόνο για μία εφορ οικονομία, και για τη δημιουργία θέσεων εργασία, αλλά σήμερα είναι και μια απαραίτητη απάντηση για τις νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, όπως ε, δημοκρατικές ελέγχες, ε, η μετάβαση σε εφόρο διαχείριση των πόρων. Καλωσορίζω λοιπόν αυτές τις προοπτικές που θέτει η συγκήτρια, που είναι από κάτω προς τα πάνω. Νομίζω ότι είναι ορθή η προσέγγιση αυτή γιατί αυτή η προσέγγιση μας επιτρέπει να λάβουμε υπόψη καλύτερα τα μοντέλα του καταναλωτή και αυτό είναι πολύ σημαντικό για την επιτυχία της καινοτομία. Επίσης, συμφωνώ με την ανάγκη να προωθήσουμε την ε, ατομική καινοτομία, πρόσβαση στην αγορά, εξάλληψη των εμποδίων, πρόθεση ιδεών την ε, διατομεακή, διαπολιτική προσέγγιση και προθυμένη συνεργασία μεταξύ όλων των φορέων, κυβερνήσεων, πολιτών, οργανώσεων, συμπράξεων για την καινοτομία κτλ. Γενικά, η έκθεση λοιπόν είναι σωστή. Μια μικρή λεπτομέρεια μόνο ότι, εντάξει, γνωρίζετε ότι ο καθένα έχει και τι δικέ του θέσει. Ιδεολογικά υπάρχουν κάποιε έννοιε που χρησιμοποιούνται από την εισηγήτρια που μπορεί να δημιουργήσουν κάποιε αμφιβολίε, όπω ε, αυτή η έννοια social innovation, κοινωνική κοινοτομία. Νομίζω πρέπει όλοι να συμφωνήσουμε από αυτού. Και η αποσύνδεση τη οικονομική ανάπτυξη από τη χρήση των πόρων πολύ ωραία ακούγεται. Αλλά πρέπει και αυτό να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί διαφορετικά θα μπορούσαμε να είμαστε και στη σφαίρα της ουτοπία. Αλλά πέραν αυτού, καλωσορίζουμε ε, θετικά την έκθεση αυτή. Καβάλιο. Ευχαριστώ κύριε Καβάλιο. Uh, Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια. Θα ήθελα απλά να προσθέσω κάτι το οποίο για μένα χαρακτηρίζει όλες τις πρωτοβουλίες που λαμβάνει η Ευρώπη για την καινοτομία επειδή αναλαμβάνουμε μεγάλες πρωτοβουλίες ή έχουμε μεγάλα προγράμματα για την καινοτομία, αυτό δεν σημαίνει ότι η καινοτομία θα υπάρξει. Η καινοτομία είναι ένα πολύ περίπλοκο σύστημα. Πρέπει να υπάρχει καλή και οργανωμένη έρευνα, σωστή ανώτατη εκπαίδευση με σωστή χρηματοδότηση, όλα αυτά. Χρειάζεται να υπάρχει κοινωνική δεξιότητα στον ε, πληθυσμό και αυτό έχει να κάνει με το γενικό εκπαιδευτικό επίπεδο. Έχει να κάνει με σύγχρονες υποδομές, σωστέ συνθήκες εργασίας, ευέλικτες και δημοκρατικές κοινωνίες, λειτουργούσες αγορές και πέρα από όλα αυτά χρειάζεται να υπάρχει και κουλτούρα καινοτομία και η δυσκολία ε, συνίσταται στο ότι αν λείπει μία από αυτές τις διαστάσεις που προανέφερα δεν θα υπάρξει καινοτομία μπορεί να δημιουργηθεί βαθιά, ε, βαθιά απογοήτευση στην Ευρώπη. Ε, να ληφθεί αυτή η τεράστια πρωτοβουλία, για την καινοτομία και στη συνέχεια να αποτύχουμε γιατί μια από αυτές τις συνιστώσεις δεν θα υπάρχει, δεν θα λειτουργεί. Ε, αν δηλαδή κομμάτι ε, αυτής της πολιτικής δεν υλοποιηθεί και δεν λειτουργήσει σωστά από τα κράτη-μέλη, θα αποτύχει αυτό το εγχείρημα. Νομίζω λοιπόν ότι είναι σωστό να δούμε ότι πρέπει να διασφαλίσουμε την ύπαρξη όλων ε, εκείνων των συνιστοσών που απαρτίζουν την ε, καινοτομία. Δεν αρκεί να έχουμε ένα μεγάλο και ωραίο ευρωπαϊκό πρόγραμμα για να επιτύχουμε την ε, καινοτομία. Αλλά όπως και να έχει είναι μια πολύ καλή έκθεση και σας ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Λάμπερτς θα επειδή δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο, στις κοινωνικές προκλήσεις. Μπορείτε να θεωρήσετε ότι ο καθένας έχει τη δική του άποψη. Είναι σημαντικό όμως αυτό, γιατί αυτό θα πρέπει να καθορίσει την πολιτική για την καινοτομία. Θα ήθελα να διαμορφώσω κάπως αυτά που προτείνει η κυρία Μερκής. Ξεκινώντας με το δεύτερο στοιχείο για την μετάβαση στην βιώσιμη διαχείριση των πόρων, συμφωνώ ουσιαστικά με αυτά οτιδήποτε έχει να κάνει με τους φυσικούς περιορισμούς του πλανήτη. Νομίζω ότι πρόκειται για ένα από τα βασικά ζητήματα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Και αν μπορούμε να πετύχουμε την καινοτομία, θα μπορέσουμε να είμαστε και ηγετικοί σε παγκόσμιο επίπεδο. Έχουμε το δυναμικό. Τα άλλα δύο στοιχεία όμως. Να αντιμετωπίσουμε όσα άπτονται της κοινωνικής συνοχής αναφέρεστε σε θέματα αστικοποίησης μετανάστευσης που θα μπορούσαν να υπάγονται στο γενικότερο αυτό το τομέα. Όντως, πρόκειται για μια μεγάλη πρόκληση για την Ευρώπη, γιατί βλέπουμε ότι αυξάνονται διαφορές και στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό μεταξύ των χωρών, των κοινωνιών. Αυτό αποτελεί μια πρόκληση για την σταθερότητα της Ευρώπης στο μέλλον. Αυτό θα το ήθελα ως δεύτερο στοιχείο. Και τρίτο στοιχείο, σε ό,τι αφορά την υγεία. Το να υπάρχει μια αξιοπρεπής ζωή, ακόμα και σε μια γυράσκουσα κοινωνία, αντιμετωπίζοντας όλα τα θέματα υγείας. Νομίζω ότι αυτό θα το έβαζα ως τρίτο στοιχείο. Μία ερώτηση. Κατά πόσο θα πρέπει στόχος μας να είναι η ανταγωνιστικότητα ή η οικονομική βάση. Αφε αυτή. Θεωρώ ότι θα πρέπει φυσικά να υπάρχει μια βιώσιμη οικονομία που να υποστηρίζει τους στόχους αυτούς, αλλά αν η οικονομία δεν εξυπηρετεί την ευημερία, τα πράγματα δυσκολεύουν. Γι' αυτό λοιπόν δεν είναι η οικονομία αυτή στόχος. Θα καταθέσουμε κάποιες τροπολογίες που σκοπό θα έχουν να διευκρινίσουν αν θέλετε κάποια άρθρα, αλλά ξέρω ότι πάντα είναι ευπρόσδεκτα τα σχόλια αυτά γι' αυτό λοιπόν ελπίζω να εκτιμήσετε τις τροπολογίες που θα θέσω. Ευχαριστώ. όλη Εγώ εδώ συμφωνώ στην αναγνώριση του έργου της ε, εισηγήτριας. Είναι πολύ καινοτόμος ε, η εργασία της. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο κατάλληλο κομπλιμέντο για μια έκθεση που ασχολείται με την καινοτομία. Συμφωνώ με όσα έχουν γραφτεί. Θα κάνω μόνο μία πρόταση και θα ζητήσω κάτι για το οποίο θα παρουσιάσω και μια τροπολογία. Νομίζω ότι στο πλαίσιο αυτής της εργασίας, που είναι μια ολοκληρωμένη και διατομεϊκή προσέγγιση, θα μπορούσαμε να τονίσουμε στον τομέα της ε, καινοτομίας για τις υπηρεσίες και τη βιομηχανία. Θα μπορούσε να αποτελέσει αυτό μεγάλη συνεισφορά για να υλοποιήσουμε την αντιμετώπιση των προκλήσεων ε, που έχουν προσδιοριστεί εδώ. Ε, ήμουν στην, παρευρέθησα στη Ρώμη ε, ένα, σε μια συζήτηση που έγινε από σε ένα πάνελ που οργάνωσε η Κομισιόν και εκεί ακριβώς αναφερόταν πώς αυτές οι νέες υπηρεσίες μπορούν να προωθήσουν την καινοτομία. Έτσι λοιπόν θα ζητήσω από την συγκήτρια αν είναι δυνατόν να τροποποιήσει αυτό το είδος μεθοδολογίας που έχει χρησιμοποιήσει ε, στην εκθεσή της και να βρει έναν τρόπο να δώσει έμφαση και σε αυτό το τμήμα ε, και που μπορεί να αναφέρεται σε αυτό το συγκεκριμένο νέο τομέα γιατί εκεί μπορούν να απασχοληθούν πολλοί και οι νέοι και οι γυναίκες για να δημιουργήσουν αυτές τις καινοτόμες υπηρεσίες. Νομίζω ότι είναι σημαντικό στοιχείο που πρέπει να υπογραμμιστεί σε μια τέτοια έκθεση. Έτσι λοιπόν πολλά συγχαρητήρια και από μένα. Kollegin Herzog. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική έκθεση και συμφωνώ απόλυτα με όσα ελέγχθησαν. Θέλω να τονίσω μόνο ένα ζήτημα, το οποίο πρέπει νομίζω ε, να τύχει μεγαλύτερης προσοχής. Και αυτό είναι ο ρόλος των κρατών μελών. Δεν, θα δημιουργούμε την ένωση της κοινοτομίας στη θέση των ε, κρατών μελών, αλλά το, το κάνουμε από πάνω και υπάρχει ένας κίνδυνος τώρα τα κράτη-μέλη να πούν «Α, το ανέλαβε η Ευρωπαϊκή Ένωση και εμείς δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτε». Να σας δώσω το παράδειγμα της δικής μου χώρας, τη χώρα που γνωρίζω καλύτερα. Ο προϋπολογισμός... Είχε... 70 της... Υπόθηκε φέτος ε, ότι η Ουγγαρία εξοικονόμησε το 70% της χρηματοδότησης που θα πήγαινε στην καινοτομία επειδή έλαβε χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωραία συγχαρητήρια, αλλά δεν είναι αυτός ο δρόμος. Τα κράτη-μέλη και η κοινωνία των ε, κρατών μελών πρέπει να ε, διαδραματίσουν στρατηγικό ρόλο. Είμαι και το γεγονός ότι συμμετέχω και στον προϋπολογισμό ε, με βοηθάει να βλέπω ότι η καινοτομία αναφέρεται όταν περισσεύουν τίποτα λεφτουδάκια από εδώ και από εκεί. Όχι, δεν γίνεται έτσι. Πρέπει να είναι στρατηγική, πρέπει να είναι προτεραιότητα. Ε, εγώ θα υποβάλω και σχετικές ε, τροπολογίες. Απλά ήθελα να τονίσω ότι δεν, δεν κάνουμε αυτά τα πράγματα στη θέση των κρατών μελών, αλλά τα κάνουμε από πάνω, υπό την έννοια μιας επίβλεψης. Η κυρία Μέρκε, θέλει να μιλήσει λίγο για να απαντήσει σε αυτά που είπε ο συνάδελφος Κούτσε θα ήθελα να παρουσιάσει κάτι που ήθελα να παρουσιάσει ο συνάδελφο, αλλά δεν μπόρεσε να είναι εδώ. Μάλιστα, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Μέρκη για την συνδέση τη, αλλά και για την συνεργασία. Ε, το σχέδιο γνωμοδότηση για την Επιτροπή Πολιτισμού θα ψηφιστεί την επόμενη Πέμπτη και να πω ότι υπήρξε ήδη ευρεία ομοφωνία μεταξύ των κρατών μελών για τις προτεραιότητες της Ευρώπης, αν και πολλές ιδέες αποτυπώνονται ήδη στην έκθεση της κυρίας Μέρκης από την ε, ε, Επιτροπή Πολιτισμού τονίσαμε ότι αν θέλουμε να πετύχουμε τους στόχους μας για τις γενοτομίες θα πρέπει να επισπεύσουμε τις ε, προσπάθειές μας, θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη πρόσβαση στην ε, παιδεία, ιδιαίτερα στην τριτοβάθμια, να υπάρχει μεγαλύτερη σύνδεση μεταξύ της εκπαίδευσης της παιδείας και των επαγγελματικών τριεντοτήτων, να υπάρχει και επαγγελματική κατάρτιση και να υπάρχει επίσης μεγαλύτερη δέσμευση σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λοιπόν, λέει ο Πρόεδρος, να δώσω τον λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Thank you very much, Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω την κυρία Μερκής για την πολύ καλή έκθεση και για τα σχόλια. Θα ήθελα να τονίσω όσα υπόθηκαν από την κυρία Χέρτσανγκ ε, δηλαδή ότι θα ήταν καλό να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση ακριβώς στο ρόλο και στη σημασία της στρατηγικής προσέγγισης για την καινοτομία. Δηλαδή η καινοτομία δεν είναι κάτι που γίνεται από μόνη της, αλλά αποτελεί τμήμα των περισσότερων από τις υπόλοιπες πολιτικές και συμφωνώ εδώ με την κυρία Καρβάλιο που είπε ότι δεν ε, θα πετύχουμε την καινοτομία με ένα μέτρο ή με ένα πρόγραμμα αλλά είναι κάτι ε, το οποίο είναι οριζόντιο. Επίσης ε, θέλουμε επίσης να μιλήσουμε για ενοποίηση. Εδώ βρισκόμαστε ξέρετε σε περίοδο οικονομικής κρίσης αλλά θα ήταν έξυπνο να μην ε, μειώσουμε τον προπολογισμό που έχουμε για την έρευνα, για την παιδεία και την καινοτομία στο μέλλον. Είναι πάρα πολύ σημαντική και πρόσβαση στη χρηματοδότηση για τις ΜΜΕ. Θέλω να τονίσω πόσο σημαντικό σημαντικό είναι ε, ο διαφορετικό τρόπο χρηματοδότησης ανάλογα με το είδο τη μικρή και μεσαίας επιχειρήσης και ανάλογα με το βαθμό ανάπτυξης αυτών των ε, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Χρειαζόμαστε λοιπόν δάνεια, επιδοτήσεις, κεφάλαιο, Ε, και κάθε ένα από αυτά έχει το δικό του σκοπό. Τα πανεπιστήμια ελπίσεις ε, έχουν ανάγκη για πρόσβαση στη χρηματοδότηση, αλλά η πρόσβαση στη χρηματοδότηση είναι πολύ περιορισμένη από το βαθμό της αυτονομίας. Έτσι λοιπόν ε, χρειάζεται σε ορισμένους τομείς και μεταρρύθμιση στα πανεπιστήμια. Η κυρία Σαρτόρη αναφέρθηκε σε κάτι πολύ σημαντικό που έχει να κάνει με τη διάδοση και κοινοποίηση των αποτελεσμάτων. Τίποτα θα συμβεί αν δεν έχουμε μια καλή στρατηγική για την χρήση και τη διάδοση των αποτελεσμάτων. Τώρα για το κέντρο ενιαία εξυπηρέτηση, πράγματι είναι κάτι πολύ σημαντικό. Ο Επιτροπ... Επιτροπό μα ε, το έχει αναφέρει σε πάρα πολλά σημεία. Πρέπει να βρούμε έναν ευφύ τρόπο ε, να το πράξουμε αυτό, ίσω μέσω διαδικτύωση, ε, γιατί είναι πολύπλοκο ο κόσμο στον οποίο ζούμε και το κέντρο Ινέα εξυπηρέτηση εξυπηρέτησης ε, θα έπρεπε να μπορεί να αντικατοπτρίζει την πολυπλοκότητα του κόσμου στον οποίο ζούμε. Θα σταματήσω εδώ και σας ευχαριστώ πολύ όλους και την εισηγήτρια. Σα ευχαριστώ πολύ, κυρία Μέρκη. Θέλετε να κάνετε κάποιε καταληκτικέ παρατηρήσει. Ευχαριστώ, συνάδελφοι, για τι παρατηρήσει σα, πολύ πολύτιμε. Συμφωνώ Συμφωνώ μαζί σα ότι είναι κάπω ε, ε, λακωνική η έκθεση σε ό,τι αφορά του ορισμού. Θα πρέπει ίσω να το διορθώσουμε αυτό. Θα πρέπει να ξέρουμε τι σημαίνει η κοινωνική καινοτομία και ασφαλώ. να σας ε, μιλήσω ώρες ολόκληρε, άμα θέλετε για θέματα τη χρήση των πόρων και το καθεξής. Φυσικά έχουμε και την ανακοίνωση και την δημοσίευση ιδιαίτερα των επιτυχιών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό προκειμένου τώρα να αναφερθώ. Και ναι, θα πρέπει να είμαστε πιο συγκεκριμένοι. Αν υπομονώ να λάβω όλες τις προτάσεις για βελτίωση που θα μου στείλετε, ποτέ δεν θεωρούσα ότι αυτή η καινοτομία της Ένωσης θα αντικαταστήσει οτιδήποτε. Ίσως, κοιτάξτε, διστάζω να πω ότι θα έρθει από πάνω, ότι θα καπελώσει την καινοτομία των κρατών μελών. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και καλά θα κάνουμε να το επαναλαμβάνουμε όποτε μπορούμε, ότι η εστίαση στην καινοτομία θα λειτουργήσει μόνο αν όλοι οι φορείς συνταχθούν και να αρμονιστούν. Ο καθένας έχει να διαρματίσει το ρόλο του και τα κρατημέλη. Αλλά βασικά θα πρέπει όλοι να υποστηρίζουμε τους ίδιους στόχους. Ιδάλλως, έχουμε πολλές ιδέες, οι οποίες όμως ποτέ δεν θα συνενωθούν για να πετύχουν ένα στόχο. Μάλιστα, ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών είναι η 3η Μαρτίου στις 12. Στενά τα περιθώρια, όλοι να κάνουμε μία προσπάθεια και να περάσουμε τώρα στο 9 μια νέα εμπορική πολιτική για την Ευρώπη στα πλαίσια της στρατηγικής Europe 2020. Ο κύριος Κτσουπ. Αχ, ποτέ δεν θα μάθω πώς να λέω το όνομά σας, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Επιτροφή Περιφερειών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Επιτροπή έχουν αυτό το έγγραφο που αναφέρεται στο ε, εμπόριο. Παρόλο που έχει γίνει έρευνα, ε, είναι το θέμα ποια θέση θα πάρει η Επιτροπή πάνω σε αυτό το θέμα. Το εμπόριο είναι ένα από τα πιο σημαντικά θέματα στην ευρωπαϊκή πολιτική. Αυτή εδώ η πολιτική θα πρέπει να συνδεθεί με άλλες πολιτικές ε, περιοχές έχουν στρατηγική σημασία όλα αυτά εν ώψη του 2020. Ε, έχουμε να κάνουμε την καλύτερη οικονομική ανάπτυξη, την απασχόληση και το πώς ακριβώς θα ξεπεράσουμε την υπάρχουσα κρίση. Πάρα πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται ακόμα σε, κρίση. Ελπίζουμε λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορέσει να δράσει σε αυτό εδώ τομέα. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό όλα όσα γίνονται εξωτερικά και εσωτερικά, εσωτερικό και εσωτερικό εμπόριο δηλαδή, θα πρέπει να αποτελούν σημαντικά μέρη αυτής εδώ της στρατηγικής. Αυτό εδώ το πρόγραμμα, ε, όπως ξέρετε, θα αναπτυχθεί, θα συνεχώς θα και θα πρέπει να εξασφαλιστούν οι σωστές, οι σωστές προϋποθέσεις στην Επιτροπή, στην Επιτροπή Εμπορίου, ο συνάδελφός μας ο Κασπάρη που δούλευσε εκεί, μας είπε ότι στην έκθεσή του κοιτάει να κάνει με θέματα τα οποία εμείς ε, ε, μας ενδιαφέρουν στην Επιτροπή μας, είναι προσφυλή σε μας, φέρει πίνει το θέμα της ενέργειας. Στο έγγραφο της Επιτροπής αναφέρεται το θέμα τα που έχουν να κάνουν με την ε, ε, πρόσβαση στην ενέργεια και αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι θα υπάρχει μια αμοιβαιότητα όταν συζητάμε για ενεργειακές αγορές. Θα πρέπει να δούμε ε, πόση σημασία έχει να έχουμε μια σωστή ενεργειακή αγορά, μια βελτιωμένη θα έλεγα ενεργειακή αγορά, η οποία να μπορέσει να συμβάλλει στην ανάπτυξη. Επίσης πρέπει να δούμε ότι τα θέματα που έχουν να κάνουν με την ενέργεια έχουν να κάνουν και με άλλες πολιτικές που αφορούν φέρει τη βιομηχανία. Και αυτό θα πρέπει να το υπογραμμίσουμε. Και εδώ θα πρέπει να δώσουμε έμφαση. Επίσης, έχουμε την έκθεση του Μπίτικ ε, και οποία, την οποία θα έχουμε αμέσω μετά, όπου και εκεί θίγονται θέματα που αφορούν το έγγραφο της Επιτροπής. Μετά έχουμε το θέμα της ε, ε παγκοσμιοποίησης και θα πρέπει να δούμε από τη βιομηχανική σκοπιά Ε, για το πώς ακριβώς θα έχουμε και εμείς κάποιο όφελος από αυτήν εδώ την ανάπτυξη. Έχουμε να κάνουμε με μέσα δηλαδή τα... Μπορούν να, μέσα τα οποία μπορούν να βοηθήσουν χώρες οι οποίες έχουν πληγεί από την ε, μετεγκατάσταση επιχειρησιών. Απ' την άλλη όμως όταν κοιτάμε αυτό το θέμα βλέπουμε ότι δεν είναι και πάρα πολλές. Είναι μια σειρά χωρών μελών θα πρέπει λοιπόν πάνω σε αυτό να σκεφτούμε, δηλαδή πώς να ενισχύσουμε τον ανταγωνισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και εδώ η στρατηγική της Ευρώπης για το 2020 είναι πολύ σημαντική. Δηλαδή αποτελεί ακρογωνίο λίθο όσον αφορά την ανάπτυξη των μεγάλων επιχειρήσεων. Θα πρέπει δηλαδή να πάρουμε μια ιδιαίτερη θέση πάνω σε αυτό εδώ το θέμα. Και εδώ έχουμε να κάνουμε με κάποιες προκλήσεις. Από τη μία θα πρέπει να δούμε πώς μπορούν οι επιχειρήσεις στο εμπόριο να βγει στην διεθνή αγορά και εδώ υπάρχει κάποιο ε, ε, δυναμικό ε, και αυτό σημαίνει ότι ίσως σήμερα δεν βρίσκονται στην καλύτερη διεθνή κατάσταση. Απ' την άλλη έχουμε την παγκοσμιοποίηση η οποία θα πρέπει να συμβάλλει στην ενίσχυση της ανάπτυξης, θα λέγαμε της πνευματικής και να μπορέσουν στο τέλος και οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να μπορέσουν να αναπτυχθούν και να βγουν ε, στον διεθνή στίβο. Όσον αφορά την ενέργεια, είχαμε μια κρόαση στην Επιτροπή μας και είδαμε ότι υπάρχει ένα μεγάλη δυναμική σε αυτόν τον χώρο. Τώρα, θα ήθελα επίσης να υπογραμμίσω ότι το, έχουμε και να κάνουμε και με το ρόλο της γεωργίας, του γεωργικού κλάδου. Υπάρχει άμεση σχέση με, την, ε, με τις τιμές, με το κόστος όσον αφορά την ενέργεια. Εδώ έχουμε να κάνουμε αποφάσεις, πολιτικές αποφάσεις. Διότι πλέον ε, έχουμε να δούμε μια κατάσταση όπου η έχουμε αυξήσει με τις τιμές των τροφίμων και εισαγωγές, ε, ε, καθαρά εισφορείς, θα λέγαμε ε, εισαγωγής όσον αφορά το τρόφιμα. Επίσης θα μπορούσαμε εμείς να δούμε το θέμα των επενδύσεων και πώς ε, ε, αυτό το θέμα έχει να κάνει με την παραγωγικότητα και τις τιμές σε αυτό εδώ το σχέδιο έκθεση. εγώ δεν, ελα... δεν να συμπεριλάβω όλες τις πτυχές αλλά παρόλα αυτά να πω ότι είχα πρόσβαση σε έγγραφα αυτό είναι σημαντικό και θα πρέπει να συμπληρώσω επιπλέον ε, όλα τα δυνατά σχέδια που έχω. Φυσικά σε αυτήν εδώ την πρόταση που σας κάνω, την παρουσίαση δεν έχω την, ε, τον κατάλληλο χώρο σας. Επίσης υπάρχει το θέμα των ε, συμφωνιών ε, με τρίτους, εμπορικές συμφωνίες, όλα αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ πολύ. Να σας παρακαλέσω Συνάδελφοι, να προσπαθήσετε και πάλι να είστε λακωνικοί. Ο συνάδελφο Ρούμπιχ έχει πρώτο το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το πρώτο και το πιο ουσιώδε είναι ότι θα πρέπει να κάτσουμε να σκεφτούμε σε περίπτωση που ολοκληρωθεί ο γύρος του ΠΟΕ ποιοι θα είναι οι βασικοί πυλώνες που θέλουμε να κρατήσουμε για τον επόμενο γύρο. Έχουμε τα θέματα της Σιγκαπούρης, σε ό,τι αφορά τις ε, θέματα ανταγωνισμού, προστασίας της ιδιοκτησίας, ε, δημοσίων συμβάσεων. Θα πρέπει όλα αυτά να αποτελούν βασικά θέματα για το 2020. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε και την συνεργασία με τον κόλπο. Θα πρέπει να υπάρχει διμερή συμφωνία ε, μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρετε, επί 20 χρόνια προσπαθούμε και διαπραγματευόμαστε με τα κρατή του κόλπου. Ακόμα όμως δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή. Δεν είναι δυνατόν μετά από 20 χρόνια να μην έχει ολοκληρωθεί μια τέτοια διαπραγμάτευση με μια τόσο σημαντική ομάδα. Θα πρέπει να το εξετάσουμε αυτό και οι περιφερειακές συμφωνίες που θα ενταχθούν στα πλαίσια και διμερών ε, συμφωνιών θεωρώ ότι θα μπορούν να εισαχθούν οι στρατηγικοί αυτοί. Θα πρέπει να ίσως και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει ε, μια ανακοίνωση για να μας πει ποιες είναι οι συμφωνίες που βρίσκονται σε εξέλιξη. Ο κ. Συνόρφος Μπαλσίτης, ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την εκτενή του έκθεση όπου παρουσιάζει με σαφή τρόπο τα προβλήματα. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αναφέρθηκε το θέμα των ενεργειακών πόρων, αλλά και άλλα ζητήματα. Ωστόσο, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι όλοι δεν ε, μπορούμε να αναφέρουμε όλα τα ζητήματα στην έκθεση αυτή. Το πρόβλημα είναι ότι είναι διαφορετική η νομική κατάσταση σε κάθε κρατος μέλος. Άρα θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα εμπόδια αυτά ουσιαστικά θα απαλληφθούν και σε ό,τι αφορά τις δημόσιες προμήθειες. Και εδώ θεωρώ ότι υπάρχει σημαντικό πρόβλημα, γιατί σε κάποιους τομείς, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τους πόρους και την πρόσβαση για κάποιες χώρες, ε, δυσκολεύεται σημαντικά. Υποστηρίζω λοιπόν το έγγραφο αυτό και ελπίζω να οδηγήσει σε μια καλύτερη κατανόηση της κατάστασης στα κράτη-μέλη, αλλά και της κατάστασης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, ο συνάδελφος μου Τικόφερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Απόλυτα δίκαιο και με λακωνικό τρόπο αναφέρει ότι το εμπόριο θα πρέπει να είναι τμήμα της εμπορικής μας πολιτικής και όχι όπως το παρελθόν κάποιες φορές όπου μας ε, δίνονταν η εντύπωση ότι η πολιτική, η εμπορική δεν είχε τη σημασία που της άρμοζε. Κατά δεύτερον, θα ήθελα ε, να εστιαστώ σε τρία σημεία, εν συντομία. Τρία σημεία τα οποία θα ήθελα να υπογραμμιστούν πιο έντονα. Θα ήθελα να υπογραμμιστεί ότι η φιλόδοξη πολιτική για την καινοτομία πρέπει να συνδεθεί με την προσέγγιση αυτή. Επίσης, να υπογραμμίσουμε ότι η παραγωγική συνεργασία μεταξύ ανταγωνιστικότητας και ανταγωνιστικότητα για το μέλλον και βιωσιμότητας πρέπει να επιτευχθεί. Τρίτον, θεωρώ ότι είναι επίσης σημαντικό να καταστεί σαφές ότι μιλάμε αν θέλουμε να προασπίσουμε μακροπρόθεσμα τα συμφέροντά μας, θα πρέπει να υπάρχουν αμοιβαία συμφέροντα στις εμπορικές σχέσεις με τις άλλες χώρες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λίγο, έχουν ε, οριακά τα πράγματα, είναι λέει ο Πρόεδρος για με το χρόνο, αλλά να δώσω το λόγο στην ε, συνάδελφο γιατί δεν μπορούσε να έρθει ω χειόδηση συζήτηση ο κ. Καμπάν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο συνάδελφος Ντεκάμπος ε, θα ήθελε να ευχαριστήσει την εισηγήτρια, τον εισηγητή για την εξαιρετική του δουλειά. Μεταξύ Δεν, θέλουμε όμως να τονίσουμε μόνο τα θετικά στοιχεία, αλλά και τα στοιχεία που μας προξενούν ε, αλησυχίες. Πρώτον, θα χρειαστεί χρόνος για όλα αυτά. Κερδίζονται μερίδια αγορά στις αναδυόμενες αγορές και αυτό είναι θετικό. Όσο αφορά την Κίνα, επιτακτική ανάγκη είναι να αυξηθεί η πρόσβαση σε αυτές τις αναπτυσσόμενες αγορές και να μειωθεί το ελληματικό ισοζύγιο το εμπορικό με αυτή τη χώρα. Δεύτερον, έμφαση δίδεται στην πρόσβαση στην αγορά, αλλά αυτό δεν πρέπει να είναι σε βάρος των βιομηχανικών αγαθών. Είναι ζωτική σημασίας να προστατεύσουμε τις ευκαιρίες ε, των ευρωπαϊκών βιομηχανιών να έχουν πρόσβαση στις διεθνείς αγορές για να αντισταθούν στον έντονο ανταγωνισμό και στις πιέσεις για μεταφορά της ε, παραγωγικής του δραστηριότητας αλλού. Πρέπει επίσης να εκμεταλλευτούμε τομείς εντάσεως ε, τεχνολογίας και καινοτομίας. Επίσης υπάρχει και η ρυθμιστική σύγκληση με τρίτες χώρες και ενίσχυση του κρίκου μεταξύ των ρυθμίσεων για τις εξωτερικές και εσωτερικές αγορές. Αυτό μπορεί να αποβεί σε βάρος της υγιεινής και της ασφάλειας, καθώς και της προστατείας των καταναλωτών. Εγώ νομίζω ότι τα πρότυπα της ζωής μας πρέπει να προστατευθούν και να επιβληθούν στην πράξη ε, και για, τα, για την εμπορία τόσο των υπηρεσιών όσο και των αγαθών. Προβλέπετε Επίσης, προβλέπονται επίσης σε περίπτωση φυσικών θεομηνιών όπως αυτή που έγινε στο Πακιστάν, ε, να επιτραπούν κάποια έκτακτα μέτρα. Τα μέτρα αυτά είναι ανθρωπιστικής φύσης, αλλά μπορεί να έχουν σημαντικές επιπτώσεις για ορισμένες ευρωπαϊκές περιφέρειες, χώρες ή τομείς που ήδη βρίσκονται σε ευαίσθητη οικονομική θέση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να εξετάσει και να αξιολογήσει προσεκτικά τον αντίκτυπο αυτών των μέτρων. Και τέλος, Υπάρχει το Ταμείο της ε, Παγκοσμιοποίησης. Αυτό αναφέρεται λίγο περιθωριακά στην ε, έκθεση. Πρέπει να χρησιμοποιηθούν όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας για την επιτάχυση και την προσαρμογή ε, στις διεθνείς πιέσεις. Πάνω σε αυτά τα σημεία ο συνάδελφος κ. Ντεκάμπος θα θα καταθέσει τροπολογίε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ στον Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η σχέση ανάμεσα στην πολυμπορική πολιτική και τι οικονομικέ ε, και βιωματικέ δράσει είναι ένα θέμα το οποίο μα ε, φέρει πολύ κακές μνήμε. Θυμάμαι τον Επίτροπο Μέντελσον, ο οποίο έκανε έλαβε μέτρα κατά του ντάμπινγκ με τον τρόπο του. Είχαμε χάσει θέσει εργασίες και σήμερα μιλάμε για στρατηγική. Στα πλαίσια τη στρατηγικής της Σαββόνα, εμείς είχαμε αντιμετωπίσει και είχαμε κάνει κάτι ανάλογο πρώτη φορά για την Κορέα. Τώρα όμως θα ήθελα να πω ότι αυτή η έκθεση αποτελεί ένα θέμα το οποίο θα δείξει ποια είναι η θέλησή μας Δηλαδή αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε το τι ακριβώ γίνεται. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει πολυμερεί ε, συμφωνίες ε, με μια μεγάλη διαδικασία και ποτέ δεν υπήρξε διάλογος. Πότε είχαμε συζήτηση για την ανάπτυξη της εμπορικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να δοθεί μια επιτάχυνση σε όλες αυτές τις συμφωνίες. Δίνεται επιτάχυνση στο Mercosur, σε όλε τι δραστηριότητε και αποτυχαίνουμε όσον αφορά το θέμα της, ε, των ε, ανταλλαγών με την ε, ευρωμεσογειακή ζώνη. Θα πρέπει να δούμε εδώ πέρα κάποιους κανόνες που έχουν να κάνουν με την κοινωνική διάσταση. Στην ανακοίνωση της Επιτροπής, για παράδειγμα, μια μικρή αναφορά. Μια απέτηση ώστε να οι κοινωνικοί εταίροι να εφαρμόζουν κάποιες αρχές. Τα ίδια βλέπουμε για τα θέματα που αφορούν το περιβάλλον, και εδώ δεν υπάρχουν σαφείς περιορισμοί. Επίσης έχουμε το θέμα του διοξιδίου του ανθράκου και εδώ χρειάζεται μια συζήτηση και να προσθέσουμε να μην χάσουμε και εδώ θέση εργασίας. Ε, στα, πρέπει να γίνει σαφές εδώ πέρα το τι ακριβώς ζητάμε. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε απαιτητικοί όσον αφορά την αμοιβαιότητα. Ε, αυτό είναι κάτι στο οποίο πρέπει να επιμένουμε σε μια κατάσταση στο, που όπως έχει στο πλανήτη μας. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Ε, thank you, Mr. Ευχαριστώ. Η κυρία Όλσκο. Ευχαριστώ. Ως και να πω ότι Πραγματικά με καθυσχάζει η εισαγωγή του κυρίου Μπουδικόφερ και θα προσθέσω κάτι στα σουηδικά. Το θέμα αφορά πολλά θέματα, δηλαδή το εμπόριο, βιομηχανική πολιτική, εξωτερική πολιτική. Εγώ συμφωνώ με τον Μπίτι ότι αυτή η στρατηγική θα πρέπει να δώσει έμφαση σε μια βιώσιμη και ε, σωστή διαχείριση των ε, πόρων που έχουμε στη διάθεσή μας. Αυτό είναι σημαντικό. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να υπογραμμίσουμε, να δώσουμε δηλαδή μια έμφαση σε αυτό εδώ το σημείο όσον αφορά τη στρατηγική μας. Αυτό δεν έρχεται σε αντιπαράθεση με θέματα όπως έχουν να κάνουν με την ανταγωνισμό, την ανάπτυξη της θέσης Η βιομηχανική πολιτική είναι μέρος αυτού. Για παράδειγμα, θα πρέπει να γίνουμε καλύτεροι ούτως ώστε να κάνουμε καλύτερη χρήση των πρώτων υλών μας. Ξέρουμε ότι υπάρχουν ε, διαθέσιμοι πόροι στην Ευρώπη που, τους οποίους δεν εκμεταλλευόμαστε. Έχουμε την Εστονία, στις σκανδιναβικές χώρες και σε άλλες περιοχές. Υπάρχουν διάφορα μεταλλεύματα, αλλά υπάρχουν πάρα πολλές άλλες πρώτες ύλε οι οποίες ε, δεν, έχουν, ε, δεν τις έχουμε εκμεταλλευτεί καταλήλως ακόμα στην Ευρώπη. Είχαμε μια ενδιαφέρουσα ακρόαση πριν από μερικές εβδομάδες εδώ στην Επιτροπή μας. Την Πέμπτη εδώ θα έχουμε την, ε, μια άλλη ακρόαση όπου θα θίξουμε το θέμα με, για τις πρώτες ύλε και όλοι σας είσαστε ευπρόζεκτοι στην ακρόαση της Πέμπτης. Να σας δώσω κάποια παραδέγματα όσον αφορά τα θέματα που θα συζητήσουμε. Η πρόσβαση στις ε, πρώτες ύλε, ε, η παγκόσμια αναζήτηση για τις πρώτες ένα ε, έναντι του ανταγωνισμού της Κίνας και των ΗΠΑ, ποιος θα είναι ο ρόλος της διπλωματίας, αναθεώρηση ε, της πολιτικής, της ρυθμιστικής Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΕΠΑ, ε, πρόθεση αποτελεσματικής ε, παραγωγής κτλ. Όλοι είστε ευπρόσδεκτοι. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ. Oh, Ωραία, λοιπόν. Αν και περάσαμε στο επόμενο θέμα τη σημερινή διάταξη, επισήμω να κλείσουμε το 9. Ή μήπω θέλετε να κάνετε κάποιε παρατηρήσει συνάδελφε. Ε, ευχαριστώ όλου που σχολιάσανε και όλα αυτά τα βλέπω θετικά. Επίσης, θα ήθελα να πω ότι υπάρχουν τέσσερα βασικά θέματα όπως προκύπτει από αυτή τη συζήτηση. Πρώτον, θα έχουμε μια φιλόδοξη στρατηγική ε, για την καινοτομία. Επίσης το θέμα που έχει να κάνει με τον ανταγωνισμό και την βιώσιμη ανάπτυξη, το θέμα των πρώτων υλών. Επίσης έχουμε να κάνουμε το θέμα με τις διαπραγματεύσεις όσον αφορά τις εμπορικές συμφωνίες. για τους περιορισμούς στη βιομηχανία. Επίσης να πω ότι οι εμπορικές αυτές συμφωνίες σίγουρα επηρεάζουν ε, την σύγκληση όσον αφορά το κοινωνικό πακέτο που λέμε. Φυσικά έχουμε και το κόστος και όλες αυτές τις πτυχές. Αυτά είναι βασικά, θεμελιώδη θα έλεγα, μέρη σημεία τα οποία θα πρέπει να στα συμπληρώσουμε. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. 3 Μαρτίου στις 12 η ώρα το μεσημέρι, η προθεσμία κατάθεση τροπολογιών, όπως και για την άλλη έκθεση. Και περνάμε στο 10 τώρα, μια αποτελεσματική στρατηγική για τις πρώτες ύλες στην Ευρώπη. Και ξεκινάμε εδώ τη συζήτηση, θα είναι η πρώτη συζήτηση. Σίγουρα θα εμβαθύνουμε και στη συζήτηση με τον ε, συνάδελφο Ταγιάννη, με τον κύριο Ταγιάννη. Ο συνάδελφος Ποντικόφερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να σας ομολογήσω ότι στην παρούσα φάση θεωρώ ότι το θέμα αυτό είναι εξαιρετικά συναρπαστικό και χαίρομαι που θα υπάρξει και περαιτέρω συνεργασία. Το 2010 για το θέμα των πρώτων υλών και της σχετικής πολιτικής έγινε, αν θέλετε, μία έκκληση από πλευράς ε, του κοινού. Οι συγκρούσεις που προέκυψαν για τα σπάνια ορυκτά που κατάφεραν ε, να θέσουν το θέμα αυτό με ιδιαίτερο τρόπο στην καθημερινή ε, στην ημερήσια διάταξη. Το θέμα αυτό θα πρέπει να μείνει στην ημερήσια διάταξη και υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι, τους οποίους δεν πρόκειται να παριθμίσω, για τους οποίους θα πρέπει να υπολογίζουμε ότι ή ο ανταγωνισμό για την πρόσβαση στις πρώτε ύλε, αλλά και οι τιμέ των πρώτων υλών δεν θα διαμορφωθούν με σημαντικά πιο ευνοϊκό τρόπο στο μέλλον από ό,τι συμβαίνει σήμερα. Μάλλον θα υπάρξει αύξηση των τιμών και αύξηση του ανταγωνισμού. Άρα χρειάζεται μια ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική. Χρειάζεται μια βιομηχανική πολιτική η οποία όπως είπαμε θα πρέπει να συνδυάσει την βιωσιμότητα με τον ανταγωνισμό και την ανταγωνιστικότητα, θα πρέπει να είμαστε και ρεαλιστές αλλά και ρομαντιστές παράλληλα. Στην έκθεσή μου επικεντρώνομαι στην εντολή μας, όπως την κατανοώ, σε ό,τι αφορά τα ορυκτά καύσιμα. Τις πρώτες ύλες, φυσικά, για την υγειοργία είναι σημαντικό ζήτημα. Τα καύσιμα επίσης αποτελούν σημαντικό θέμα, αλλά εδώ δεν κοιτάμε τις πτυχές αυτές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρούμε ότι είναι σε θέση να κατανοήσει και μάλιστα κατανόησε τη σημασία του θέματος αυτού πριν από πολλούς άλλους και δραστηριοποιήθηκε εγκαίρως. Συμφωνώ με τους τρεις πυλώνες που έχει θέσει στη στρατηγική της. Ένας πυλώνας αφορά την ε, αποδοτικότητα των πρώτων υλών και την ανακύκλωση κτλ. Ένας άλλος στην ε, ενίσχυση, αλλά και ο τρίτος πυλώνας στην πρόσβαση στις διεθνείς αγορές. Αυτό που θεωρώ ότι είναι σημαντικό και ελπίζω να το πετύχουμε ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να ευαισθητοποιήσουμε το ευρύ κοινό. Να εξηγήσουμε πόσο λίγος είναι ο χρόνος που έχουμε στη διάθεσή μας για να δημορφώσουμε μια κατάλληλη, μια δέουσα πολιτική για τις πρώτες σύλλες και για να την πραγματοποιήσουμε. Δεν είναι μόνο η Κίνα που μας ακολουθεί, αν θέλετε, με φιλόδοξο και πολύ οργανισμένο τρόπο, οργανωμένο τρόπο τα τελευταία χρόνια, που ακολουθεί δηλαδή μια εμπορική πολιτική πολύ φιλόδοξη σε ό,τι αφορά τις πρώτες και η Ιαπωνία μετά από τις ε, άσχημες εντυπώσεις του περασμένου έτους, έχει δείξει μεγάλη δέσμευση. Ένα δισεκατομμύρια δολάρια δαπανώνται στην Ιαπωνία και θα δαπανηθούν τα επόμενα χρόνια στον τομέα της ε, πολιτικής για τις πρώτες ύλες. Άρα, θέτει φιλόδοξους στόχους ε, η Ιαπωνία σε ό,τι αφορά την κατανάλωση τέτοιων σπάνιων ορεικτών παρά το γεγονός ότι θέλει να το περιορίσει μάλλον την κατανάλωση στο 1 τρίτο της σε σχέση με την τρέχουσα κατάσταση. Οι ΙΠΑ μας έχουν ξεπεράσει αρκετά σε ό,τι αφορά την δικτύωση των διαφόρων φορέων, τη διασύνδεση των διαφόρων φορέων. Άρα πρέπει και εμείς, θεωρώ, να καταβάλουμε μεγάλες προσπάθειες χωρίς να επισέλθω σε λεπτομέρειε για τα μεμονωμένα μέσα, γιατί θεωρώ ότι αυτό θα πρέπει να γίνει σε μια μετέπειτα συζήτηση, να πω δύο λόγια για τους τρεις πυλώνες της στρατηγικής. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό το ζήτημα κατά πόσον θα ακολουθήσουμε τους Ιάπωνες. για να αξιοποιήσουμε αυτή την πρόκληση και να την καταστήσουμε μια ευκαιρία, μια ευκαιρία για μια στρατηγική για την καινοτομία που θα μας επιτρέψει να κάνουμε ένα άλμα προς τα εμπρός. από τις επαφές μου με τις επιχειρήσεις έχω ακούσει πολλές ε, διαφορετικές ε, τοποθετήσεις. Κάποιες ε, κλαίγονται, κάποιες είναι φιλόδοξες και διατυπώνουν φιλόδοξους στόχους, τέτοιων φιλόδοξους στόχους. Λένε λοιπόν ότι θα πρέπει να ακολουθήσουμε και να κάνουμε αυτά που κάνουν οι Κινέζοι. Γιατί να περιμένουμε να μας ξεπεράσουν, γιατί να μην είμαστε εξίσου φιλόδοξοι. Αποτελεσματικότητα των ε, πρώτων υλών, αλλά και ανακύκλωση. Ανακύκλωση, αλλά και σε τομεί που δεν είχαμε φανταστεί μέχρι πρόσφατα. Ανακύκλωση σπάνιων ορεκτών. Κάποιων από τα οποία δεν, είχαμε το το είχαμε καν σκεφτεί πριν από τρει μήνες. Ύστερα, το θέμα του domestic mining. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ θετικό ότι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στη Γενική Διεύθυνση Βιομηχανίας και Περιβάλλοντος ε, υπήρξε μια συνεργασία προκειμένου να συζητήσουν θέματα για την Natura 2000 και να αποτραπούν ενδεχόμενες αποκλήσεις. Νομίζω ότι ακριβώς αυτή τη γραμμή της ε, σωστής συνεργασίας πρέπει να ακολουθήσουμε αν θέλουμε να κοιτάξουμε και την άμεση γειτονία. Εντάξει, η Γρυλανδία μπορεί να μην είναι εγχώριο, να μην είναι domestic ε, τομέας, αλλά τέλος πάντων νομίζω ότι θα πρέπει εξ αρχής ε, να είμαστε ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι και τρίτον και τελευταίων και σίγουρα είναι ο πιο δύσκολος τομέας αυτός σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στη διεθνή αγορά. Εδώ σαφώς και ζητώ μία, όχι μάλλον μία, πολλές στρατηγικές συνεργασίας. Φυσικά, φυσικά μπορούμε σε κάποιους τομείς να επιχειρήσουμε και το έχει επιχειρήσει άλλωστε η Ευρωπαϊκή Ένωση και σε ό,τι αφορά το Μεξικό αλλά και τη ΣΥΠΑ. Μπορούμε να προσπαθήσουμε να τα βρούμε στον ΠΟΕ, αλλά το να πιστεύουμε ότι μέσω τέτοιων μηχανισμών ε, σύγκρουσης μπορούμε να ρυθμίσουμε θέματα πρόσβασης, νομίζω ότι είναι μεγάλη αυταπάτη. Θα πρέπει να καταρτήσουμε σχετικές στρατηγικές με τον ΩΣΑ, με, με την Ιαπωνία και τη ΣΥΠΑ, αλλά και στρατηγικές σε ό,τι αφορά την Κίνα και με άλλες χώρες ε, που είναι πλούσιες σε πρώτες ύλες. Τελευταίο τώρα σημείο. Στην παρούσα φάση δεν είναι ακόμα σαφές κατά πόσο στην Ευρώπη η ανάγκη αυτή για την αποδοτική πολιτική για τις πρώτες ύλες γίνεται αντιληπτή από όλους. Και μήπως ε, θα διαμορφωθεί μια νέα, ένα νέο είδος, αν εθνικού εγωισμού ή αν θα υπάρξει όντως μια ευρωπαϊκή συνεργασία. Ελπίζω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μπορέσει να συμβάλλει προκειμένου να επιλεχθεί αυτός ο κοινό δρόμος παρά τα μεγάλα κράτη-μέλη και τα ενδεχόμενα συμφέροντά τους. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα 6-7 άτομα έχουν ζητήσει λόγο, 8 ομιλητές. Ο Επίτροπος θα έρθει στις 5.30. Αν περιοριστείτε σε ένα-ενάμιση λεπτό, θα μιλήσετε όλοι. Ιδάλλως θα πρέπει να διακόψουμε. Ο συνάδελφος Σιμάνσκι έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το θέμα. Γιατί δεν υπάρχει νομοθετική κατηγοριοποίηση, αλλά η δική μας επιλογή σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στις ε, πρώτες ύλες, ε, ε, καθορίζει και τη θέση των πιο προηγμένων ευρωπαϊκών βιομηχανιών στην παγκόσμια οικονομία. εμείς θα μπορούσαμε <laughs> ίσως να διαλύσουμε όλες αυτές τις βιομηχανίες στην Ευρώπη και να τις στείλουμε όλες στην Κίνα, αν δεν είμαστε προσεκτικοί. Έχουμε τρία εργαλεία. Ε, έχουμε την εμπορική πολιτική, πρέπει να τη χρησιμοποιήσουμε αποτελεσματικά για να μπορέσουμε να έχουμε πρόσβαση στις πρώτες ύλες. Για να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Βιομηχανία να έχει πρόσβαση στις πρώτες ύλες. Και έχουμε και ίδιους πόρους η Ευρώπη διαθέτει πόρους, δεν είναι στερημένη πόρων. Ε, ορισμένες φορές τις ε, είχαμε, τους είχαμε χρησιμοποιήσει τους πόρους αυτούς και πρέπει να θεωρήσουμε αυτή την πολιτική γιατί έχουμε πάρα πολλές πρωτεσίλες στο υπέδαφος και δεν χρησιμοποιούνται λόγω ορισμένων ε, ευαισθησιών. Και έχουμε και το θέμα της ανακύκλωσης και της αποτελεσματικής χρήσης. Πάρα πολύ σημαντική και αυτή η πτυχή, όχι λιγότερο σημαντική από τις άλλες δύο πτυχίες, αλλά ας θυμόμαστε ότι η ανακύκλωση και η αύξηση ε, των προτύπων κοστίζουν πάρα πολύ για τις επιχειρήσεις. Όμως, ε, αν υπάρξει μία νομοθετική παρέμβαση, τότε θα μπορούσαμε, αν δεν υπάρξει μια νομοθετική παρέμβαση, τότε θα μπορούσαμε να ε, οφήσουμε αυτές τις επιχειρήσεις σε άλλα σημεία του κόσμου. Πιστεύω ότι αυτές τις τρεις πτυχές πρέπει να τις δούμε με ισορροπημένο τρόπο. Ο συνάδελφος Ρούμπεχ, ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να συμφωνήσω με τον συνάδελφο Μπουτικόφερ. Είναι πολύ σημαντική η στρατηγική αυτή, ιδιαίτερα για τη βιομηχανία μας, γιατί από αυτό εξαρτώνται πάρα πολλές θέσεις εργασίας και στην βιομηχανία μεταποίηση, αλλά και στην ε, βιομηχανία την χρηματοοικονομική. Χρειαζόμαστε λοιπόν σωστή ρύθμιση για να ρυθμιστούν σωστά οι τομεί αυτοί. Σίγουρα δεν μπορεί να ισχύει το one fits all, μία λύση για όλου. Θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένε, μεμονωμένε λύσει. Και σίγουρα θα υποβάλει συγκεκριμένε προτάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ληφθούν υπόψη οι ξεχωριστέ ανάγκε και στους εμπορικούς όρους, ιδιαίτερα στο διεθνές προσκήνιο, ανεξάρτητα αν μιλάμε σε διμερές επίπεδο ή σε επίπεδο ΠΟΕ, το θέμα είναι να υπάρχει και στρατηγική ε, συνεπειών. Και τα ζητήματα της Σιγκαπούρης είναι σημαντικά, το είπα και προηγουμένω αν θέλουμε να έχουμε επενδυτική ασφάλεια. Πολύ απλά θα πρέπει να γίνονται σεβαστά τα απαραίτητα κριτήρια. Θα πρέπει να υπάρχουν θα πρέπει να λειτουργούμε και βάσει των κανόνων των ισχύοντων. Υπάρχουν πολλές βασικές προϋποθέσεις σε θέματα έρευνας. Θα πρέπει να βρεθούν και προϊόντα υποκατάσταση. Συμφωνώ με τον συνάδελφο Μπουτικόφερ σε ό,τι αφορά ε, θέματα έγκρισης και σε ό,τι αφορά το Natura 2000. Και τέλος, σε ό,τι αφορά την ανακύκλωση, θα πρέπει να την ε, θεωρήσουμε συνολικά. Νομίζω ότι μπορούν να δημορφωθούν ευέλικτοι κανόνες για να ανταποκριθούμε και στις ανάγκες του μέλλοντος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. εδώ και καιρό είναι προφανές ότι υπάρχει το πρόβλημα ανισορροπίας μεταξύ ζήτησης και προσφοράς ε, σε παγκόσμιο επίπεδο στις πρώτες ύλε. Ε, το υφίσταται το πρόβλημα αυτό και Ευρώπη και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Και αυτή η πολύ ισχυρή ζήτηση που προέρχεται από αναδυόμενες ασιατικές οικονομίες μας υποχρεώνει να αναζητήσουμε ένα είδος κοινή ε, στρατηγικής Αυτό που μας προτείνει η Επιτροπή βασίζεται σε τρεις πυλώνες, όπως εξήγησε και ο κ. Μποτικόφερ, φυσικά συμφωνούμε. Πρέπει να προωθήσουμε την ε, αϊφόρο ε, εξόρυξη στην ε, ίδια την Ένωση. Προτείνονται μια σειρά μεθόδων πολυλογικών και μια σειρά εργαλείων. Εδώ θέλω να τονίσω την αρχή της επικουρικότητας, γιατί οι ανισότητες μεταξύ κρατών μελών είναι τεράστιες. Στη δική μου χώρα, ε, στο 30% της επικρατειάς της ε, είναι προστατευόμενες ε, περιοχές από Ιρλανδική Σκοπιά. Ενώ όλες χώρες έχουν πολύ μικρότερο ποσοστό. Έτσι λοιπόν, όταν μιλάμε για εκμετάλλευση πόρων, δεν έχουμε ίδια μεταχείριση μεταξύ των χωρών. Τώρα, πρόθεση της ανακύκλωσης ε, και αποδοτική χρήση των πόρων. Πρέπει να το προωθήσουμε και αυτό. Υπάρχουν υπερβολικά πολλά κρατημέλη, όπου η κύρια διαδικασία της επεξεργασίας ε, είναι να τα ρίχνουν στη χωματερή και τελικά στο τέλος έρχεται ένα σύστημα ανακύκλωσης. Έτσι λοιπόν εδώ πρέπει να αναλάβουμε δράση από κοινού για να αποφεύγουμε τέτοιες καταστάσεις. Και τέλος... Έχουμε και τον πυλώνα της δίκαιης εκμετάλλευσης και η φόρο εκμετάλλευσης των πρώτων υλών σε παγκοσμίο Βλέπετε τι γίνεται στον αραβικό κόσμο και η Ευρώπη πρέπει να σκεφτεί για το αν θα πρέπει να υποστηρίξουμε αδίστακτους και διεφθαρμένους δικτάτορες απλώς γιατί ε, μας βολεύει τη στιγμή που θα βοδιαστούμε με πρώτες ύλες ή αν θα πρέπει να λειτουργήσουμε με έναν έξυπνο πολιτικό τρόπο και ηθικά σωστό γιατί ε, τελικά μακροπρόθεσμα ε, αν ακόμη και στηρίζουμε αυτά τα καθεστώτα, τι στην ε, καταλήγουμε στο να έχουμε ένα πάρα πολύ ένα χειρότερο ε, καθεστώς που είναι και εχθρικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι λοιπόν καλύτερο είναι να υποστηρίζουμε δημοκρατικά καθεστώτα και έτσι θα έχουμε και λιγότερες δυσκολίες σε γεωπολιτικό επίπεδο. Ασφαλώς, ε, συμφωνώ με τους συναδέλφους οι οποίοι θεωρούν ότι είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό και σίγουρα θα μας απασχολήσει στους επόμενους μήνες. Στην παρούσα φάση, επειδή δεν έχουμε και πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, θα ήθελα να περιοριστώ σε δύο ζητήματα. Πρώτον, καταρχάς, η βιώσιμη διαχείριση των πρώτων υλών, το αναφέρει αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ωστόσο, να μην μείνουμε στον τομέα των ευγενών προθέσεων και να μην μείνουμε στα ωραία λόγια. Πρόσφατα στα διεθνή μέσα ενημέρωσης αναφέρθηκε ότι μεγάλες μεταλλουργικές εταιρείες κοιτούν την κάθετη ενσωμάτωση, δηλαδή όλο και πιο συχνά αποκτούν πλέον ε, ε σε χώρες του τρίτου κόσμου. Είναι θετική αυτή η εξέλιξη άραγε. Και κυρίως πώς θα φροντίσουμε να είναι βιώσιμη η εξόρυξη αυτών των ε, πρώτων υλών. Δεύτερο ζήτημα σε ό,τι αφορά την αποδοτική χρήση και την ανακύκλωση. Ε, ασχολούμαι εδώ και χρόνια με θέματα που αφορούν το περιβάλλον και βλέπουμε ότι στην όλη συζήτηση για τις πρώτες ύλες πάντα επικρατεί ένα οικονομικό επιχείρημα για την ανακύκλωση, υπέρ της ανακύκλωσης. Πώς γίνεται αυτό και πάλι βλέπω στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πάρα πολύ όμορφα λόγια αλλά πολύ λίγες συγκεκριμένες δράσεις. Ποτού δεν βλέπω την ε, αναφορά για παράδειγμα στην πρωτοβουλία Cradle to Cradle το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να φροντίσουμε τα προϊόντα να παράγονται με τρόπο που να, μπορούν, να επιτρέπουν την ανακύκλωσή τους. Και όχι να παράγονται γρήγορα γρήγορα για να διατεθούν στην αγορά. Και κάτι άλλο, το οποίο πάντα αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά στην πράξη δεν μας ε, πετυχαίνει, είναι σε ό,τι αφορά τη διαρροή από τον τρίτο κόσμο κατά όχι κατά τύχη, αλλά εν πάση περιπτώσει βρέθηκα στο λιμάνι της Αμβέρσας της πόλης μου για να δω πώς γίνεται η εφαρμογή του κανονισμού για τα ηλεκτρονικά απόβλητα. Ό,τι θέλουμε μπορούμε να λέμε, αλλά αν περνούν τόνοι κάθε χρόνο από τα λιμάνια μας, ό,τι και να λέμε, όσο όμορφα και αν το λένε, δεν θα πετύχουμε τίποτα. Θα πρέπει να φροντίσουμε οι υπολογιστές, τα κινητά τηλέφωνα και του καθεξής να μένουν στο δικό μας έδαφος, στην δική μας επικράτη και να ανακυκλώνονται με βιώσιμο τρόπο. Η κυρία Δελκαθήγιο λέει ο Πρόεδρος. Πρόεδρε, πολύ σύντομα για να μην επαναλάβω όσα υπόθηκαν. Ο συνάδελφος ε, Βιταλκό Συμφωνώ απόλυτα. Θέλω να επιμείνω σε δύο σημεία όμως. Πρώτον, στις διαφορές που υπάρχουν σε ό,τι αφορά στην προστασία των εδαφών σε ορισμένα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είπαμε ότι στην Ισπανία προστατεύεται το 30% της επικρατειάς μας το δίκτυο Natura ε, καλύπτει το 30% της δικής μας επικράτειας, ενώ σε άλλες χώρες μιλάμε για το 14-15%. Και ε, όπως ε, προκύπτει σε αυτές τις προστατευόμενες περιοχές ακριβώς υπάρχουν μια σειρά ορεικτών πόρων που δεν μπορούμε να τους εκμεταλλευτούμε λόγω της περιβαλλοντικής προστασίας. Έτσι λοιπόν χρειάζεται αυτό που μέχρι τώρα η ε, Επιτροπή δεν ήθελε να το λάβει υπόψη, ε, να το λάβει υπόψη, γιατί πολύ δύσκολο θα είναι να πάμε σε μεγαλύτερη αυτόχθον παραγωγή και σε μεγαλύτερη βιωσιμότητα, αν δεν λάβουμε υπόψη αυτές τις πηγές παραγωγής που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τι υπάρχουν αυτοί οι περιβαλλοντικοί περιορισμοί. Φυσικά πρέπει να έχουμε υπόψη και τον περιβαλλοντικό στόχο, αλλά θα πρέπει να δούμε και πώς θα το συνδυάσουμε με αυτή την αναγκαιότητα. Και η δεύτερη πτυχή είναι η εξή, αναφέρθηκε και από τον κύριο Ρούμπικ. Είναι θεμελιώδη σημασία να αναζητήσουμε πέρα από την ανακύκλωση, να αναζητήσουμε ε, κάποια στοιχεία, κάποια υλικά, κάποιες ύλες υποκατάστασης. Αυτές οι ύλε υποκατάστασης δεν μπορούν παρά να έρθουν από την έρευνα στους τομείς αυτούς. Ε, στο μέλλον θα έχουμε το 8ο πρόγραμμα πλαίσιο και νομίζω ότι θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον να εξετάσουμε και αυτό το πεδίο έρευνας σε σχέση με αυτή τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω από το πρόγραμμα πλαίσιο και να επιμείνουμε στον τομέα αυτό ο ρόλος της έρευνας για την απόκτηση τέτοιων υλών υποκατάστασης είναι πάρα πολύ σημαντικός καθώς θα μείωνε τις αναγκαιότητες που έχουμε σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ τον κύριο Μπουτικόφερ, τον συγχαίρω και αυτά από μένα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι σημαντικό το θέμα και όλοι συμφωνούμε ότι η ανάγκη για πρώτες ύλες στο μέλλον θα αυξηθεί. Βλέπουμε λοιπόν ε, τι προβλήματα υπάρχουν σήμερα σε ό,τι αφορά το φυσικό αέριο. Κάποια κρατημέλη πληρώνουν 30% παραπάνω για το φυσικό αέριο από ότι κάποια άλλα. Φυσικά υπάρχουν γεωγραφικές ε, διαφορές και διαφορές ως προς την περιβαλλοντική πολιτική. Αντιλαμβανόμαστε τα προβλήματα που οθούν στα ύψη της τιμές των τροφίμων. Βλέπουμε και τι συμβαίνει στην Βόρεια Αφρική. Όπου οι υψηλές τιμές των τροφίμων προκάλεσαν μέχρι και την κατάρρευση καθεστώτων. Βλέπουμε και ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί στη διεθνή αγορά πρώτων υλών, όπου είναι έντονη η κερδοσκοπία. Αναφέρθηκαν οι τρεις ε, πυλώνες. Συμφωνώ με το μοντέλο αυτό και θεωρώ ότι ο σημαντικότερος ρόλος πρέπει να τον διαδραματίσει μάλλον σημαντικότερο ρόλο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι σημαντικό αυτό να αποτυπωθεί ανάλογα και στο έγγραφό μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Μερικής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αναζητάμε κάποια στοιχεία. Έχουμε και τις πρώτες ύλε και σχετική ανακοίνωση και την αποδοτικότητα των ε, πόρων. Μοιάζει μια ανακοίνωση με την άλλη, αλλά δεν είναι το ίδιο. Να σας πω ότι θα ήθελα να υπάρχει λίγο πιο σαφή δομή. Όπως είπε ο κ. Μπιλικόφερ, υπάρχουν ε, τρεις πυλώνες. Στην αποβατικότητα των πόρων είναι λίγο πιο έντονη οι δύο πρώτες ε, οι δύο πρώτοι πυλώνε και θεωρώ ότι κάποια θέματα θα ταιριάζαν καλύτερα στην άλλη ανακοίνωση. Γιατί σε τελική ανάλυση το θέμα είναι τι θα κάνουμε με, τους, με τις πρώτες ύλες. Άρα θεωρώ ότι θα πρέπει να συνενωθούν τα δύο θέματα και θεωρώ ότι έχουμε χάσει μια ευκαιρία εδώ. Και γι' αυτό επικεντρωνόμαστε στο πώς θα μπορέσουμε να έχει η Ευρώπη πρόσβαση στις πρώτες ύλες. Σαφώς και είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα αυτό. Υπάρχει επίσης εστίαση στην, στο εμπόριο, στις πρώτες ύλες, αλλά δεν υπάρχει επαρκής επικέντρωση στην αποδοτικότητα. Πώς μπορούμε, με πιο ευθύ τρόπο να καταναλώνουμε τις πηγές αυτές. Άρα τελικά το θέμα των πρώτων ύλων είναι λίγο άσχετο με το θέμα της αποδοτικότητας. Ε, των πόρων. Και είναι κρίμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ασφαλώς και το επιδιώκω και εγώ. Αλλά τελικά έχουμε καταλήξει σε μια φιλοσοφική ανάλυση παρά σε συγκεκριμένα μέτρα, τα οποία πραγματικά θα ήθελα να υπάρχουν. Ύστερα, να πω ότι με ικανοποιεί το γεγονός ότι η ανακοίνωση δεν επικεντρώνεται μόνο στις πρώτες αλλά και σε άλλα σπάνια ορυκτά και ίσως ε, κάποια ε, υλικά. Να μην, φαίνεται ότι, να μην φαίνεται σήμερα ότι μπορούν να καταστούν σπάνια, όπως το ξύλο για παράδειγμα, η ξυλία, αλλά δεν ξέρουμε τι θα γίνει στο μέλλον. Άρα να μην περιοριστούμε στα ορυκτά, στις ορυκτές πρωτοσύλλες, αλλά και σε άλλα είδη σπάνιων υλών, πρώτων υλών. Δεν θεωρώ ότι θέματα περιβαλλοντική προστασία και αποδοτικότητα των πόρων είναι αντίθετα και θεωρώ ότι θα πρέπει να έχουμε πιο πολύ χρόνο για τη συζήτηση αυτή. Ευχαριστώ, κυρία Νίμπλερ. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Είδα ότι κοιτάτε το ρολόι σας. Τρεις παρατηρήσει. Καταρχάς θεωρώ κύριε Μπουτικόφερ ότι η έκθεση αυτή είναι σε πολύ καλά χέρια και αυτό το επιβεβαίωσαν ε, οι σημερινές σας ε, επεξήγησεις. Θα ήθελα να σας υποστηρίξω. Είναι σημαντικό στην Επιτροπή ε, Βιομηχανίας να επικεντρωνόμαστε σε θέματα βιομηχανικής πολιτικής. Αν περιληφθούν και άλλα γεωργικά προϊόντα, νομίζω δεν θα βγάλουμε κάποια άκρη θεωρώ ότι καλό είναι που επικεντρωθήκατε στην έκθεσή σας αυτά που αφορούν εμάς, την ε, πολιτική, την Επιτροπή ε, Βιομηχανίας. Κατά δεύτερον, το είπαν και άλλοι συνάδελφοι, συμφωνώ ότι το πιο σημαντικό είναι να κοιτάξουμε κατά πόσον μπορούμε να δημορφώσουμε μια ευρωπαϊκή προσέγγιση σε ό,τι αφορά την πολιτική για τις πρώτες ύλες και Θεωρώ ότι αποτελεί ένα από τα βασικά ζητήματα που θα απασχολήσουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τους επόμενους μήνες και καθημερινά διαβάζουμε στις εφημερίδες και διαπιστώνουμε και η ότι υπάρχουν και εθνικά συμφέροντα. Νομίζω όμως ότι σε ό,τι αφορά το φάκελο αυτό θα πρέπει αγαπητέ συνάδελφοι Μπουτικόφερ να αποσταλεί ένα σαφέ μήνυμα ότι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα επικεντρωθούμε σε μέτρα και πολιτικές που θα έχουν την υποστήριξη των κρατών μελών. Τρίτο θέμα το οποίο έθιξαν και συνάδελφοι. Θέλουμε να βρούμε σωστές λύσεις και από πλευρά περιβαλλοντικής προστασίας. Νομίζω ότι έχουμε ε, ηγετική θέση ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι ίσως θα έπρεπε να επιτραπούν ε, σε σχέση με την σχετική οδηγία και κάποιες εξαιρέσεις. Θα πρέπει κάπως να διαμορφωθεί με πιο ευέλικτο τρόπο η νομοθεσία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ ο συνάδελφος podział... όσον αφορά το θέμα των πρώτων υλών και ο τρόπος προσέγγισης του θέματος. Θα πρέπει εδώ να δούμε ότι υπάρχουν νέες τεχνολογίες όσον αφορά την ε, εκμετάλλευση, την χρησιμοποίηση πρώτων υλών. Ε, υπάρχουν τρόποι φερπή να ε, κάνει κανείς χρήση φυσικού αερίου, να μπορέσει να το εκμεταλλευτεί όταν υπάρχουν κοιτάσματα. Αυτό είναι σημαντικό. Επίσης, ε, και είναι ένα θέμα που θα το θίξω στην Ολομέλεια, η πολιτική για τις πρώτες ύλε. Είναι κάτι για το οποίο ε, υπάρχουν αντιδράσεις από τις χώρες μέλη Υπάρχει μια ομάδα χωρών μελών η οποία δείχνει ενδιαφέρον όσον αφορά αυτό το θέμα. Εδώ έχουμε να κάνουμε μία, θα λέγαμε, πολιτική ε, αιμονής, καταναγκαστική. Ε, και εδώ έχουμε ένα πρόβλημα, δηλαδή, όταν κανείς ε, σκέφτεται ή νιώθει ότι πρέπει οπωσδήποτε να ακολουθήσει κάποιους κανόνες. Ε, είχαμε, όπως ξέρετε, ε, εκλογές στο Σουδάν ε, και άλλες περιοχές. Ξέρουμε ότι εκεί πέρα υπάρχει θέμα κοιτασμάτων πετρελαίου. Ε, υπάρχει ενδιαφέρον από άλλες περιοχές του κόσμου. Από την Κίνα, Φερπίν. Υπάρχει το θέμα της εξέλιξης όσον αφορά την ε, εκμετάλλευση πόρων, το κόστος και όλα αυτά συσχετίζονται με το διεθνές εμπόριο. Υπάρχει αυτή η διάσταση. Ευχαριστώ. Μάλιστα, σας ευχαριστώ. Προλάβα να μιλήσουν όλοι. Συνάδελφε Μπιουτικόφερ, θέλετε να μιλήσετε τώρα. Τέσσερις προτάσεις, θα τα μετρήσουμε. Θα τις μετρήσουμε όμως. <laughs> ναι, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τις ιδέες και τις προτάσεις τους. Υπόσχομαι ιδιαίτερα στην κυρία Μερκής ε, τα συγκεκριμένα μέτρα να συμπεριληφθούν στην έκθεση και συμφωνώ με αυτά που μόλις είπε ο συνάδελφος Τσίπ σε ό,τι αφορά τις νέες τεχνολογίες και την πρόσβαση στις ε, πρώτες ύλες σε τομείς που δεν το είχαμε σκεφτεί στο παρελθόν. Και να πω ότι θεωρώ ότι είναι θετικό το γεγονός ότι ως τώρα και ελπίζω έτσι να μείνει δεν υπήρξε κράχ μεταξύ, δεν υπήρχε συγγνώμη, σύγκρουση μεταξύ ε, περιβαλλοντικής πολιτικής και εμπορικής πολιτικής και βιομηχανικής πολιτικής. Μεταξύ των προτάσεων της Γενικών Διευθύνσεων α, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν υπάρχει κριτική από καμία από τις δύο Γενικές ε, Διευθύνσεις Τρίτων. Συμφωνώ με αυτά που είπαν η ε, κυρία Φανμπρέμπτ, ε, Δελκαστήγιο και Βιδελκουάντρας ότι θα πρέπει να προσέξουμε τι γίνεται στην πράξη, να μην μείνουμε στην διατύπωση γενικών ε, αρχών. Αυτό ισχύει και για το, την οδηγία WEEE, αλλά και θέματα πρόσβασης σε πρώτες ύλες, αλλά και για άλλα ζητήματα. Τέλος, τελευταία πρόταση προς τον κύριο Τσιμάνσκι ήμουνα πριν από... Μα τέταρτη πρόταση, πρόεδρε. Πριν από μία εβδομάδα παραβρέθηκα στην 10η ε, ε, σε 11ο συνέδριο ανακύκλωση αλουμινίου. Και είπαν, υπόθηκε το εξής, ότι αν 95% μάλλον αν υπάρχει ανακύκλωση αλουμινίου, θα μπορούσαμε να γλιτήσουμε 95% της ενέργειας που χρησιμοποιείται για την παραγωγή νέων προϊόντων και νομίζω ότι αυτό αποτελεί το ύψιστο επιχείρημα ότι μπορεί να είναι και οικονομικά ένα ανακύκλωση. Μάλιστα, λέει ο Πρόεδρο, σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Κλείνει το θέμα αυτό τη ημερήσια διάταξη και ανακαλωσορίζει τον Επιτρόπο Ταγιάννη για πολλαπλή φορά εδώ στην Επιτροπή μα. Βρίσκεται μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε δύο θέματα κατά σε ό,τι αφορά την ε, πράξη για τις μικρές επιχειρήσεις και για θέματα πρώτων υλών. Μπορεί δηλαδή να ξαναδείξουμε θέματα για τις πρώτες ύλες. Καταρχάς να σας καλωσορίσω και κατά δεύτερον σας δίνω το λόγο. Επίτροπε για κάποιες εισαγωγικές παρατηρήσεις και μετά θα κάνουν ερωτήσεις οι συνάδελφοι. Τάγκεσεν κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σε όλους. Πριν να σας αναπτύξω τις δύο πρωτοβουλίες εφαρμογή του εγγράφου μας για τη βιομηχανική πολιτική. Θα ήθελα να συγχαρώ την Επιτροπή σας για την στήριξή σας, για τη στήριξη που προσέφερε γιατί η έκθεση του κυρίου Λάνκε ερμηνεύει τέλεια το πνεύμα της δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία άλλωστε εκέρδισε και τη στήριξη του Συμβουλίου γεγονός που μας ικανοποιεί βαθύτατα. Ελπίζουμε λοιπόν να κερδίσουμε και τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο όπως ξέρετε αγαπώ πάρα πολύ. 14 χρόνια δεν πέρασαν εις Μάρτιν βεβαίως. Όπως ξέρετε, την περασμένη Τετάρτη ε, υποβάλαμε μια πρόταση να υιοθετήσουμε την ε, πράξη για τις μικρές επιχειρήσεις, ε, στρατηγικό κείμενο, σημαντικό, όχι μόνο για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και για να επαναφέρουμε στο κέντρο της οικονομικής πολιτικής της Ένωσης την πραγματική οικονομία ο λόγος, αφορά, ο λόγος για ένα θέμα που αφορά πολύ υψηλό ποσοστό των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, αφορά σχεδόν το 70% της απασχόλησης και επομένως το να εργαζόμαστε για την επιτυχία των μικρομεσαίων επιχειρήσεών μας σημαίνει ότι εργαζόμαστε όχι μόνο ότι εργαζόμαστε για έναν κρίσιμο τομέα, αλλά ότι εργαζόμαστε για εκατομμύρια Ευρωπαίων εργαζομένων. Το 2008 υιοθετήθηκε, ήδη ήταν ένα φιλόδοξο σχέδιο, ε, σημαντικό. Ε, καταφέραμε χάρη στη στήριξη του Κοινοβουλίου να επιβάλλουμε έναν βασικό κανόνα. Ε, σκέφτομαι την οδηγία για, την καθυστέρηση, για τις καθυστερούμενες οφειλές και την καθυστέρηση των πληρωμών, διατάξεις που ήδη έχουν τεθεί σε λειτουργία. Και το τελευταίο στοιχείο ε, στο οποίο είμαστε λίγο αδρανείς είναι το καθεστώς της Ευρωπαϊκής Ιδιωτικής Εταιρείας. Ελπίζω η πρόταση αυτή να εγκριθεί εν τέλει και από το Συμβούλιο. Έχουμε εγκρίνει λοιπόν ένα κείμενο το οποίο θέλει να δώσει όθηση ξανά ε, σε αυτήν την πράξη των μικρών επιχειρήσεων γιατί η κρίση έχει πλήξει και τις μικρές επιχειρήσεις και χρειάζεται μια ανανέωση της συνεργασίας ε, των ε, θεσμών, τόσο των ευρωπαϊκών όσο και των ε, εθνικών. Η στρατηγική που θα σας παρουσιάσω σήμερα λοιπόν ε, διέρχεται μια καινούρια φάση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να στηρίξει αυτόν τον τομέα, τον τόσο σημαντικό της οικονομίας μας. Βεβαίως η πραγματικότητα έχει αλλάξει σε σχέση με το 2008. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν απολέσει πολλές θέσεις εργασίας, σχεδόν 3 εκατομμύρια 325.000 θέσεις εργασίας έχουν χαθεί. Ε, καθόλου αμεληταίος αριθμός. Τι συγκεκριμένο λοιπόν υπάρχει σε αυτό το έγγραφο ενημέρωσης, επικαιροποίησης της πράξης ε, για τις μικρές επιχειρήσεις. Καταρχήν, δώσαμε μία όθηση στον στην, ε, στον κύριο, τον υπεύθυνο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τον πρέσβη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Όπως θα ξέρετε, ο καινούριο υπεύθυνο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ο κύριος Ντανιέλ Καγέχα, ο οποίος βρίσκεται και εδώ. Σας παρακαλώ να έρθετε και εδώ, παρακαλώ. Ντανιέλ, έλα εδώ. Σε χαιρετώ και θα ήθελα πολύ να έρθει εδώ, λέει στα Ισπανικά ο κύριος Ταγιάννη. Ο κύριος Ντανιέλ Καγιέχα είναι ο νέος γενικός διευθυντής, ε, αναπληρωτής γενικός διευθυντής ε, της Γενικής Διεύθυνσης ε, για τις επιχειρήσεις. Εκείνος τώρα θα πρέπει να αγρυπνεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την υλοποίηση και εφαρμογή της πράξη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επειδή όμως θέλουμε ακριβώς ε, μάλλον επιλέξαμε ένα πρόσωπο που θα αγρυπνά πραγματικά για την εφαρμογή αυτής της πράξης στα κράτη-μέλη. Θέλουμε το άτομο αυτό να είναι σημείο αναφοράς για όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να είναι κάποιος που θα μπορεί να τις παρακολουθεί συστηματικά από τη θέση του, από το αξίωμά του, να μπορεί να παρακολουθεί όλες τις δράσεις υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ε, ζητήσαμε από όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ορίσουν και εκείνα έναν πρέσβη ε, ε, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επίσης, ζητήσαμε από την τοπική αυτοδιοίκηση τις Ιταλικές περιφέρειες, τις, τις Ισπανικές περιφέρειες, ε, τα κρατήδια της Γερμανίας, γενικά όλες οι αρχές της τοπικής αυτοδιοίκησης που έχουν τη σχετική αρμοδιότητα να ορίσουν και αυτές έναν υπεύθυνο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για την εφαρμογή της πράξης ε, των μικρών επιχειρήσεων στην επικράτειά τους. Όλοι αυτοί οι εκπρόσωποι των εθνικών τοπικών θεσμών θα έρθουν εδώ στις Βρυξέλλες να συμμετέχουν σε μια ημερίδα εργασίας για να δουν πώς πρέπει να υλοποιηθεί, πώς πρέπει να εφαρμοστεί η πράξη για τις μικρές επιχειρήσεις. Ένα είδος οργάνωσης που θα ε, αντιπροσωπεύει όλο το μηχανισμό που θα υπάρχει για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ελπίζουμε ότι έτσι θα δημιουργήσουμε ένα συμπίλημα καλών ιδεών ε, για δράσεις υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ε, με συμβουλευτική δράση. Ο, ο, ο ρόλος αυτής της οργάνωσης θα είναι να παρακολουθεί όλες τις σχετικές πολιτικές, τις δημόσιες διοικήσεις των κρατών μελών, αλλά και τους συλλόγους και τις ενώσεις των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η ομάδα αυτή θα ορίσει κριτήρια παρακολούθησης των δράσεων που θα αναλαμβάνουν τα διάφορα κράτη-μέλη, γιατί διακυβέρνηση πρέπει να σημαίνει και συνεχή έλεγχο των αποτελεσμάτων, αλλά και στενή συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης και κρατών μελών. Αποφάσισα να παρουσιάσω αυτή την ενημέρωση της πράξης για τις μικρές επιχειρήσεις, όχι μόνο στο Κοινοβούλιο, αλλά και στις διάφορες ε, χώρες μέλη. Το, το παρουσίασα ήδη την περασμένη εβδομάδα στη Ρώμη Μεθαύριο θα το παρουσιάσω στο Ηνωμένο Βασίλειο και στο Παρίσι την ίδια εβδομάδα, στη συνέχεια στη Γερμανία και στη Βουλγαρία. Πρέπει να ομολογήσω ότι η Βουλγαρία ήδη ανήγγειλε, ανακοίνωσε ότι θα διορίσει κάποιον υπεύθυνο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σύμφωνα με την υπόδειξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ήδη λοιπόν θετικές ενδείξεις έρχονται και θετικά σήματα από πολλές χώρες και από πολλές αρχές της τοπικής αυτοδιοίκησης. Μία άλλη ιδέα την οποία ξεκινήσαμε και ανακοινώσαμε στα κράτη-μέλη Μία φορά το χρόνο να οργανώνεται ένα συμβούλιο άτυπης ανταγωνισμού, ένα άτυπο συμβούλιο ανταγωνισμού στο πλαίσιο λοιπόν της διακυβέρνησης, μια σειρά συγκεκριμένες πρωτοβουλίες δρομολογούνται για, την, ε, για τον έλεγχο της υλοποίησης της πράξης για τις μικρές επιχειρήσεις, αλλά και για να δοθεί όθηση και παρένεση στα κράτη-μέλη και αυτά να φροντίσουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Υπάρχουν και άλλα πράγματα στην ανακοίνωση αυτή. Καταρχήν επιμένω πάνω στο θέμα της απλούστευσης, της απλοποίησης, γιατί το να, το να επιχειρηματίας θα πρέπει να είναι πιο απλό και λιγότερο ακριβό από ότι είναι σήμερα. Σίγουρα έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος, αλλά αυτό πρέπει να συνεχιστεί. Ο στόχος που προτείνουμε είναι να μπορέσουμε να συστήσουμε, να μπορεί να συστήνεται μια εταιρεία μέσα σε τρεις ημέρες με ένα μέγιστο κόστος 100 ευρώ. Θέλουμε επίσης να είναι δυνατόν να εκδοθούν όλες οι απαιτούμενες άδειε ε, σε μικρότερο χρονικό διάστημα από ό,τι απαιτείται σήμερα. Θέλουμε να φτάσουμε σε ένα μέγιστο αριθμό 30 ημερών. Δηλαδή, όποιος θέλει να συστήσει μια επιχειρήση, ε, να μην χρειάζεται να υπερβαίνει και να υπερσκελίζει ανυπέρβλητα εμπόδια και χρόνους. Ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι η πρόσβαση στι πιστώσει στην πίστονη. Απαιτούνται περισσότερες πιστώσει για τις επιχειρήσεις μας. Έχουμε σκεφτεί νέα συστήματα εγγυήσεων για τα δάνεια, μεγαλύτερων εγγυήσεων, επίσης ε, επενδύσεις και στο πλαίσιο του επόμενου οικονομικού προγραμματισμού. Επίσης, στις αγορές του επιχειρηματικού κεφαλαίου στην Ευρώπη, να τις ενεργοποιήσουμε και αυτές. Ξέρετε πόσο σημαντικό σημαντικό είναι το επιχειρηματικό κεφάλαιο, το, το venture capital. Συνεργαζόμαστε με τον συνάδελφο Μισελ Μπαγνιέ για να εκπληρώσουμε αυτό το στόχο και θα θέλαμε μέχρι το 2012 η εσωτερική αγορά να αποτελέσει μια πραγματικότητα και για τις εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου. Επίσης, προγράμματα ή εργαλεία, τα, τα προγράμματα ή τα οικονομικά εργαλεία, τα χρηματοδοτικά, τα ευρωπαϊκά πρέπει να απλοποιηθούν. Θέλουμε να αφαιρέσουμε τα ανώφελα διοικητικά προσκόμματα και τους ε, ελέγχους και θέλουμε να εντάξουμε ε, και τις ε, τράπεζες μικρότερης κεφαλαιοποίησης. Όλες οι επιχειρήσεις θα πρέπει να μπορούν να βρουν στο διαδίκτυο πληροφορίες ε, για να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα χρηματοδοτικά μέσα και όχι μόνο στην αγγλική γλώσσα, στα γαλλικά ή στα γερμανικά, αλλά και στη δική τους γλώσσα. Γιατί δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι μια μικρούλα επιχείρηση θα έχει κάποιον που θα μιλάει και ξένες γλώσσες τόσο καλά όσο απαιτείται για τους τεχνικούς αυτούς όρους. Άλλο ζήτημα είναι η πρόσβαση στις αγορές. Πρέπει να επικεντρώσουμε την εργασία μας στο θέμα των δημόσιων προκηρύξεων και διαγωνισμών. Υπάρχουν πολλά να γίνουν ακόμη. Χρειάζεται ένα κώδικα ε, καλών πρακτικών που έχει προταθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2008. Πολλά κράτη-μέλη δεν το έχουν ακόμα θέσει σε εφαρμογή αυτό τον κώδικα καλής πρακτικής. 16 11 το έχουν εφαρμόσει. Είναι μια αγορά που αξίζει το 17% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ και πρέπει πραγματικά να έρθει στην εμβέλεια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ε, ηλεκτρονική δημόσιοι διαγωνισμοί, απλοποίηση, εργαλεία τα οποία πρέπει να χρησιμοποιηθούν από τις διάφορες αρχές που προκυρήσουν διαγωνισμούς και πρέπει ήδη να σκεφτούμε την αναθεώρηση της οδηγίας για τους δημόσιους διαγωνισμούς που προβλέπεται για το 2012. Ασφαλώς σημαντικό είναι να, να δίδονται στους καταναλωτές οι απαραίτητες πληροφορίες. Πρέπει λοιπόν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να πληροφορούν τους ε, καταναλωτές για την προέλευση των ε, προϊόντων, για όλα αυτά που άπτονται της υγείας και της ασφάλειας, για την τήρηση της νομοθεσίας. Είναι κάτι η ανάγκη για το οποίο έχει γίνει αισθητή και πολλά κράτη-μέλη έχουν πάρει μέτρα για να σημειώσουν πρόοδο. Πρέπει λοιπόν τα προϊόντα και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να, γίνονται, να είναι αναγνωρίσιμα και να επικοινωνούνται ε, στο καταναλωτικό κοινό. Όταν μιλούμε για αγορές δεν μπορούμε να λησμονήσουμε ε, την ανάγκη για βέβαιους κανόνες. Λοιπόν, καταπολέμηση των καταχρηστικών εμπορικών ρητρών. Έχει να κάνει αυτό με την ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που συχνά παραπονιούνται για, αυτά τα, για αυτούς τους περιορισμούς. Υποχρεώνονται να συνάπτουν συμβάσεις με δυσβάσταχτους όρους. Αυτό δεν πρέπει να συνεχιστεί. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει ενδεχομένως να υιοθετήσει σχετική νομοθεσία. Το άλλο θέμα μεγάλης σημασίας είναι η διεθνοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ε, προετοιμάζουμε μία πρωτοβουλία για να καταστήσουμε την ε, ανάκτηση των διασυνοριακών χρεών πιο εύκολη ε, παγώνοντας τους τραπεζικούς λογαριασμούς των οφειλετών. Η σημερινή κατάσταση είναι απαράδεκτη. Δεν είναι δυνατόν μια επιχείρηση να ανταπεξέλθει σε αυτές τις συνθήκες, εάν θέλει να έχει διασυνοριακές δραστηριότητες και συναλλαγές. Στο δεύτερο ήμιση του 2011 θα παρουσιάσω επίσης και την καινούργια στρατηγική για την διεθνοποίηση. Εργαλεία όπως τα Market Access Teams ήδη παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες στις επιχειρήσεις που θέλουν να έχουν πρόσβαση σε συγκεκριμένες αγορές Απλώς χρειάζεται η βελτίωση της χρήσης αυτών των market access teams και να γίνουν αυτές γνωστές στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτά εν ολίγης περιλαμβάνει το έγγραφό μας για την πράξη περί των μικρών επιχειρήσεων. Και τώρα θα περάσω στο θέμα των πρώτων υλών. Και αυτό είναι στρατηγική σημασία ε, για την ανάπτυξη της οικονομίας μας, ε, γιατί σχετίζεται με την ανταγωνιστικότητα των επιχειρησιών μας. Ε, μέχρι προλίγου συζητήθηκε γιατί έχουμε το έγγραφο του κ. Μπουτικόφερ, αλλά θέλω να σας επαναλάβω ότι η δική μας ανακοίνωση για τις πρώτες ύλε ε, αφορά και το τμήμα της δικής μου στενής αρμοδιότητας αλλά και της αρμοδιότητας των συναδέλφων Μπαρνιέ και που αφορά τα βασικά προϊόντα και τι χρηματοοικονομικές αγορέ. Ο στόχο είναι να ρυθμίσουμε με πιο αποτελεσματικό τρόπο τη λειτουργία των χρηματοοικονομικών και φυσικών αγορών των πρώτων υλών για να έχουμε μεγαλύτερη διαφάνεια και να μειώσουμε την υπερβολική αστάθεια. Το έγγραφο φυσικά θα είναι μία συνεισφορά για την G20 και για την G8. Όμως εγώ θα ήθελα να σταθώ στα θέματα που είναι δικές μου αρμοδιότητας. Όπως ε, γνωρίζετε, εγώ ε, έχω βασιστεί σε τρεις πυλώνες. Ο πρώτος αφορά την ε, προμήθεια πρώτων υλών ε, στο εξωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεύτερον την ενίσχυση του βιώσιμου φοδιασμού στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτον την ανακύκλωση και την αποτελεσματική χρήση των πόρων η εφαρμογή της στρατηγικής του 2008 μας επέτρεψε ήδη να έχουμε κάποια σημαντικά αποτελέσματα όπως ε, η σύσταση ενός καταλόγου 14 ε, ε, σημαντικών πρώτων υλών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ανάπτυξη μιας εμπορικής στρατηγικής πρόθεση μέσω της αναπτυξικής μας πολιτικής και νέες ευκαιρίες έρευνα στο πλαίσιο του 7ου προγράμματος πλαίσιο και οι νέες κατευθυντήριες γραμμές εξηγούν ε, τους ε, κανόνες που εφαρμόζονται για τις εξορυκτικές βιομηχανίες που λειτουργούν ε, στις περιοχές Natura 2000. Κατά τη διάρκεια της Ισπανικής Προεδρίας παρουσιάσαμε αυτές τις 14 πρώτες ύλες που βρίσκονται σε κίνδυνο. Εμείς θεωρούμε ότι ορισμένες ότι ο κατάλογος θα μπορούσε να αυξηθεί Επίσης, το επίπεδο της ζήτησης το 2030 θα μπορούσε να τριπλασιαστεί σε σχέση με το 2006 για ορισμένες πρωτεσίλες. Εμείς ε, θα δούμε τι γίνεται με τις ε, σημαντικές πρωτεσίλες ε, προκειμένου να δούμε ποιες δράσεις προτεραιότητας θα αναλάβουμε. Η δική μου δέσμευση είναι να αναθωρείται τακτικά ο κατάλογος και να τον ολοκληρώσουμε. Θα ήθελα να μειώσω τον αριθμό, αλλά νομίζω ότι δυστυχώ δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Θα υπάρχει συνεχής παρακολούθηση και όπως ε, ξέρετε ε, στην ε, Ένωση παρόλο που δεν παράγουμε πολλές πρωτεσίλες δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει τέτοια δυναμική. Εμεί θέλουμε να δούμε πώ μπορούμε να ενισχύσουμε αυτή τη δυναμική τη Ευρώπη. Με το σχέδιο προ Mine. Όπως ξέρετε, ε, έχω δεσμευτεί για να συμπεριλάβω στο έγγραφο, στο σχέδιο δράσης Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αφρικανικής Ένωσης, ένα κεφάλαιο που να αφορά ακριβώς τον εφοδιασμό σε πρώτες ύλες, ένα είδος ε, συμφωνίας με την Αφρικανική Ένωση για τη στρατηγική αυτή. κατόρθωσα να συμπεριλάβω στις διαπραγματεύσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, Ρωσίας το θέμα των πρώτων υλών ε, κατά τη διάρκεια της συνάντησης ε, που είχαμε το περασμένο φθινόπωρο στη Ρώμη. Ξανασυζητήθηκε το θέμα αυτό στη συνάντηση που είχαμε την περασμένη εβδομάδα με τη Ρωσική Ομοσπονδία και θα το ξανασυζητήσω το θέμα αυτό στην επόμενη συνάντηση στην Αγία Πετρούπολη με τον Υπουργό Βιομηχανίας της Ρωσίας. Έτσι λοιπόν και από τη σκοπιά αυτή εργαζόμαστε πιστεύω για να υπερασπίσουμε το ευρωπαϊκό επιχειρηματικό σύστημα. Πριν ε, από τις διακοπές, ε, κατά τη διάρκεια του Μαΐου νομίζω, θα μεταβώ στη Λατινική Αμερική έχει 15 χρόνια να πάει ο αρμόδιο επίτροπο για τη βιομηχανία στη Λατινική Αμερική, έτσι ώστε με την ε, Βραζιλία και την Χιλή και την Αργεντινή να συζητήσω τα θέματα των πρώτων υλών. Και άλλα θέματα, αλλά κυρίω ε, θέματα πρώτων υλών. Και πρέπει να πω ότι σε όσο αφορά τον πυλώνα αυτό των πρώτων υλών, ε, εμείς θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και το ότι συζητάτε στι διμερεί και πολυσμερείς διαπραγματεύσει και να θέσουμε ω προτεραιότητα του νομικούς περιορισμούς στην εξαγωγή και σε άλλε στις και σε άλλες επενδύσεις. Σε ό,τι αφορά τώρα το δεύτερο πυλώνα, τι μπορεί να γίνει στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, να σας πω ότι έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας. Έχουμε ακόμη πολλά κοιτάσματα στην Ευρώπη. Πρέπει να συνεχίσουμε να ε, βελτιώνουμε το θεσμικό πλαίσιο που ρυθμίζει τις εξορρυκτικές δραστηριότητες στην Ευρώπη. Εμείς θέλουμε να υπάρχει, βελτί... Ε, να υπάρχει ανταλλαγή βελτιστών πρακτικών μεταξύ των αρμοδίων αρχών των κρατών μελών. Ε, ήδη έχουν εκδοθεί κάποιες ερμηνευτικές γραμμές για το, για το Natura 2000 ε, ε, σύμφωνα με τις οποίες ε, λέγεται ότι δεν υπάρχει εξόριξη κοντά σε τέτοιες περιοχές. Ο τρίτος πυλώνας αφορά το τι μπορούμε να κάνουμε εμείς στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας. Ε, είμαι επιβισμένος ότι έχουμε εμείς πραγματικά αστικά ορυχία. Γιατί πράγμα μιλάω, πρόκειται για όλα τα ορυκτά που υπάρχουν στα αποβλήτα που παραμένουν αχρησιμοποιητά αν δεν ανακυκλωθούν. Η Κομισιόν προτείνει στοχευμένα μέτρα για να προωθηθεί η ανακύκλωση και η συλλογή διασφαλίζοντα την ε, εφαρμογή της νομοθεσίας ε, για το ε, ηλεκτρονικές συσκευέ, λοχάρι ή για τα οχήματα που δεν χρησιμοποιούνται. Όπω ξέρετε, ένα από τα έγγραφα για την καινοτομία ε, προβλέπεται να υπάρχει μία σύμπραξη για την καινοτομία που θα επικεντρώνεται στην ανακύκλωση των πρώτων υλών και ε, πιστεύω ότι και το Κοινοβούλιο θα θέλει να εμπλακεί σε αυτή τη σύμπραξη για την καινοτομία και για να κλείσω. Ε, πρέπει να διασφελίσουμε την παραγωγική ικανότητα, την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση της Ευρώπης. Ε, έτσι λοιπόν ε, και σήμερα αλλά και στο μέλλον θα πρέπει να θέσουμε σε εφαρμογή. Αυτή τη δράση αποτελεί προϋπόθεση για να ικανοποιήσουμε όλες τις απαιτήσει. Για μένα πρόκειται για προτεραιότητα, το επαναλαμβάνω και θα καταβάλω κάθε προσπάθεια Ε, γιατί μπορεί να υπάρχει αποτελεσματική στρατηγική για τις πρώτες ύλες ε, με συγκεκριμένες απαντήσεις που θα βοηθήσουν ε, το επιχειρηματικό μας σύστημα. Δηλαδή δεν θα έχουμε αύξηση στο τιμών, αλλά και ταυτόχρονα θα αναλαμβάνονται δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος. Θα συνδυάσουμε δηλαδή την προστασία των επιχειρήσεων και την προστασία του περιβάλλοντος με μια συντονισμένη δράση και με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν πάρα πολλέ ερωτήσει. Έτσι λοιπόν, σταματώ εδώ και περιμένω να ακούσω τι δικέ σα παρατηρήσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Επίτροπε, για τι ε, εκτενεί αυτέ πληροφορίε για τα δύο αυτά θέματα. Πάνω από δέκα συνάδελφοι έχουν ζητήσει το λόγο. Ένα λεπτό για τον καθένα, λοιπόν. Ένα λεπτό αναλογή στον καθένα. Να τηρήσετε παρακαλώ το όριο αυτό. ή Ιδάλω δεν θα μπορούσαν να μιλήσουν οι τελευταίοι. Συνάδελφο Χέρτσοκ ξεκινάει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τον Επίτροπο που βρίσκεται μαζί μας σήμερα και που συζητάει τα σημαντικά αυτά θέματα. Δεν θα σας προκαλέσει έκπληξη αν σας θέσω το ερώτημα για την αναθεώρηση της πράξης για τις μικρές επιχειρήσεις. Θα προσπαθήσω να είμαι πάρα πολύ σύντομη. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την αντίδρασή σας και για την απάντησή σας στην προφορική ερώτηση που τέθηκε την προηγούμενη εβδομάδα από, την, από τους συναδέλφους στην ομάδα SME. Τι μπορεί να κάνει το Κοινοβούλιο για να υποστηρίξει τις προσπάθειές σας, τη δέσμευσή σας για να υπάρχουν πραγματικά αποτελέσματα από την ε, πράξη αυτή για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Γιατί αποτελέσματα θέλουν οι μικρές επιχειρήσεις, όχι ανακοινώσεις. Τέλεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο συνάδελφος Ρίμπη έχει το λόγο. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο γιατί η πράξη για τις μικρές επιχειρήσεις πάντα θα πρέπει να τίθεται στην ημερήσια διάταξη και το θέμα της μελέτης αντικτύπου. Θα πρέπει να συζητήσουμε τη μείωση, την αύξηση μάλιστα, μάλλον της ε, μείωσης της εκπομπής ε, διοξιδίου του άνθρακα. Τι σημαίνει αυτό για τις επιχειρήσεις ε, υψηλή και βιομηχανικής έντασης. Εδώ θα πρέπει να μου στείλει μία απάντηση και γενική διεύθυνση βιομηχανίας για το ποιος θα είναι ο αντίκτυπος της αύξησης ε, της μείωσης των εκπομπών σε 30% και τι θα σημαίνει αυτό για την, ε, με την επιχειρήσεων. Επίσης, σε ό,τι αφορά τις μικρές επιχειρήσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει τον όρο του 20% για το κεφάλαιο κινδύνου για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέχρι το 2020. Θα πρέπει να είναι 20% το ποσοστό αυτό για την φερεγγιότητα, για την ε, ε διασφάλιση της φερεγγιότητας και της ε, Ρευστότητα. Η κυρία Νίμπλερ, ευχαριστώ. Κυρία Επιτρόπη, σας ευχαριστώ και για την παρουσίαση και την επεξήγηση των θέσεών σας ε, για, την πράξη για τις μικρές επιχειρήσεις και συμφωνώ φυσικά γιατί πρόκειται για τον κατεξοχή κλάδο καινοτομία και την κινητήριο ε, μηχανή της οικονομίας μας. Έχουμε δύο θέματα καταρχάς. Το πρώτο θέμα που ακούω συνέχεια είναι η γραφειοκρατία και πάλι γραφειοκρατία και το δεύτερο είναι η πρόσβαση στα μέσα χρηματοδότησης. Δύο συγκεκριμένες ερωτήσεις σε ό,τι αφορά την γραφειοκρατία και να αναφέρω και αυτό που είπε και η κυρία Έρτσοκ ότι οι μικρέ επιχειρήσει αποτελέσματα θέλουν να δουν. Πριν από δύο χρόνια έγινε η συζήτηση για την υποχρέωση για τους ταχογράφους. Δεν ξέρω αν θυμάστε. Εσύ, αυτή η υποχρέωση πριν από δύο χρόνια. Και είχαν γίνει και διάφορες προτάσεις από την ε, ομάδα καθοδήγησης. Το είχαμε συζητήσει και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είχε αναφερθεί ότι δεν θα πρέπει αυτή η υποχρέωση να αφορά τι μικρές επιχειρήσεις. Τότε είχαμε θέσει ω όριο τα 50 χιλιόμετρα και τώρα λέμε ότι θα θέλουμε να επεκταθεί αυτό το όριο σε 150 χιλιόμετρα. Τι γίνεται λοιπόν με το θέμα αυτό. Ένα άλλο θέμα που συζητιέται πάρα πολύ στο Κοινοβούλιο και ψηφίστηκε, αλλά δεν ξέρετε δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα, είναι οι απλοποιημένοι κανόνες για τους ε, κανόνες ε, υπολογισμού σε ό,τι αφορά τον ισολογισμό μικρών επιχειρήσεων. Τι πρόοδο έχουμε σημειώσει. Θα ήταν καλό να μπορέσω να πω δύο λόγια στι μικρές επιχειρήσεις της περιφερειάς μου. Ευχαριστώ πολύ. Συνάδελφος Καβάλια, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Συγχαρητήρια στην Επιτροπή και στον Επίτροπο. Έχω μια ερώτηση για την ε, πράξη περί μικρών επιχειρήσεων. Όπως είπατε, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, ιδρύουν τις περισσότερες θέσεις εργασίας. Ήθελα να ρωτήσω τον Επίτροπο κατά πόσο θα μπορούσαν να δημιουργηθούν περισσότερες νέες θέσεις εργασίας για τους νέους στον τομέα αυτό και οι καινοτόμε μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι πολύ σημαντικές δυνητικά για τη δημιουργία θέσεων εργασίας για τους νέους. Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες υπάρχει σοβαρό πρόβλημα ανεργίας για τους νέους. Ξέρω ότι το, πρόβλημα αυτό σας απασχολεί όλους ιδιαίτερος, αλλά στην ανακοίνωσή σας δεν είστε πολύ δεν υπήρξατε πολύ φιλόδοξο. Λέτε να δημιουργηθούν συστήματα παρακολούθηση, να εντοπιστούν βέλτιστε πρακτικέ, να υιοθετηθούν μελλοντικά πρωτοβουλίε, αλλά δεν βλέπω να είστε πολύ φιλόδοξο ω προ αυτό. Έχετε καμία ιδέα, υπάρχουν κράτη-μέλη τα οποία έχουν να επιδείξουν κάποιε βέλτιστε πρακτικέ για του νεαρού επιχειρηματίε. Μπορούμε αυτό να το προωθήσουμε κι άλλο. Ευχαριστώ. Κυρία Καστίγιο, ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε που περιβρίσκεστε σήμερα εδώ και μας παρουσιάσετε με διαφορετικές διαστάσεις ε, δύο θέματα πολύ σημαντικά. Εγώ θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Καταρχήν, σε ό,τι αφορά τι μικρέ και μεσαίε επιχειρήσει, δεν υπήρχε αμφιβολία ότι υπάρχει πρόβλημα ανταγωνιστικότητα που θίγει κάθε είδου επιχείρηση, αλλά εδώ μιλάμε καταρχήν για τι μικρέ και μεσαίε επιχειρήσεις. Εγώ θέλω να επισημάνω ορισμένα στοιχεία που νομίζω ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη και ε, είναι τόσο σημαντικά όπω αυτά που αναφέρατε. Δεν έχει κανένα νόημα ε, να συστήνεται ταχαίω μια υπηρεσία και να υπάρχει πρόσβαση στη χρηματοδότηση κτλ. Αν έχουμε αυστηρέ και μη ευέλικτε αγορέ εργασίε. Εδώ έχουμε ένα βασικό πρόβλημα που έχουν πολλέ χώρε και πραγματικά ουσιαστικά ε, καταπνίγει τις πιθανότητες ε, όλων των ε, ε, επιχειρήσεων, κυρίως των ΜΜΕ για ανάπτυξη. Ε, ε, τώρα, το δεύτερο, νομίζω ότι ένα ζωτικό θέμα είναι αυτό που έχει να κάνει με την εσωτερική ψηφιακή αγορά. και φυσικά υπάρχουν παρόμοια προβλήματα για την ανάπτυξη αυτής της αγοράς, όπως έχουμε και για την ανάπτυξη της ενίας αγοράς. Ο κατακαιρματισμός που υπάρχει στις νομοθεσίες που αναφέρονται στα δικαιώματα θέματα των καταναλωτών, τα θέματα της διανοητικής ιδιοκτησίας. Όλα αυτά είναι σημαντικά θέματα και οι ΜΜΕ έχουν ένα διάβλο ανάπτυξη ε, σημαντικό ε, μέσω της ψηφιοποίησης, ε, γιατί βλέπουμε εδώ μία σχέση μεταξύ επενδύσεων και κόστους ωφέλου. Και τέλος, ένα θέμα που σχετίζεται με όσο είπε η συνάδελφος κυρία Καρβάλιο, κάτι που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ε, δηλαδή, να ε, μιλάμε ουσιαστικά ε, για ένα σύστημα ε, που θα μπορεί να χρησιμοποιήσει ο νέος επιχειρηματίας για τη φορολόγηση. Δηλαδή, ε, να έχουμε, παραδείγματο χάρη, έναν αριθμό φορολογικού μητρώου για το νέο επιχειρηματία. Εγώ νομίζω ότι κάτι τέτοιο θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ο συνάδελφο Μπένσον και να σα προειδοποιήσω ότι δεν πρόκειται να μιλήσουν όλοι. Ε, ευχαριστώ Πρόεδρε, να ευχαριστήσω τον Επιτροπό που ξεκίνησε αυτό το καυγά για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Όσον αφορά τις μικροψές επιχειρήσεις υπάρχουν δύο ε, θέματα. Υπάρχει το θέμα της χρηματοδότησης όπως είπε και ο Επίτροπος και ε, όπως είπατε υπάρχει το θέμα της αναθεώρησης της οδηγίας. Εδώ τώρα φυσικά εγώ δεν θα ήθελα να μακρηγορήσω αλλά το θέμα της χρηματοδότησης είναι πολύ σημαντικό για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ξέρουμε ότι είναι δύσκολα για αυτές τις επιχειρήσεις να μπουν στις ε, δημόσιες προσφορές. Ξέρουμε ότι όταν θα γίνει αναθεώρηση της οδηγίας θα πρέπει να προσπαθήσουμε ούτως ώστε να διευκολυνθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να κάνουμε τα πράγματα πιο απλά. Θα πρέπει λοιπόν αυτές οι επιχειρήσεις να έχουν καλύτερες δυνατότητες. Επίσης να πω ότι το θέμα που έχει να κάνει με το διοικητικό άχθος. Προσπαθεί κανείς να, ε, να διευκολύνει τις ε, επιχειρήσεις αυτές όσον αφορά το διοικητικό άχθος. Αλλά διαπιστώνουμε και εδώ στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή όλες οι, όλοι οι περιορισμοί, όλοι οι κανόνες που δεσπίζονται οδηγούν σε επιπλέον επιβάνηση. Θα πρέπει να το προσέξουμε αυτό. Θα πρέπει να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι για να ξεπερασεί αυτό το πρόβλημα. Κάποιο να μου εξηγήσει όμως πώς να γίνει να τελειώσουμε στην ώρα μας. Έχουμε και τους συντονιστέ μετά χωρίς να σας περιορίσω χρονικά δηλαδή. Ο κύριο Μπαλσίτη, εγώ δεν μπορώ να το καταφέρω τι να κάνω, θα πρέπει να σταματήσουμε σε λίγο. Κύριε Μπαλσίτη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αξιότιμη κύριε Επίτροπε. Ήδη σα έκαναν οι συνάδελφοι κάποια ερωτήματα. Εμένα με ανησυχεί ιδιαίτερα το γεγονό. το ότι Θέλετε η οδηγία για τις δημόσιες συμβάσεις να αναφερθεί το 2012. Θα πρέπει να σκεφτείτε τι εμπειρίες έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση όταν το 2002 15 δισεκατομμύρια ευρώ τελικά κάπου βρέθηκαν στις τράπεζες και δεν έφτασαν στα χέρια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Μιλήσατε λοιπόν για τις μικρομεσαίες αυτές επιχειρήσεις. Να σας ρωτήσω πόσο θα συνεχίσει αυτή η συζήτηση και πότε θα κατατεθούν συγκεκριμένες προτάσεις σε ό,τι αφορά τις ε, μικρόμεσαίες επιχειρήσεις προκειμένου να τους δοθούν οι σωστοί οικονομικοί όρες. Ο κύριος Ντεάντζελης. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον κύριο Επίτροπο. Πολύ γρήγορα για να μην ε, κλέψω πολύ χρόνο. Καταρχήν καθυστερήσεις πληρωμών. Εμείς συγκρίναμε την οδηγία. Εγώ θα έβλεπα χρήσιμη μια πρωτοβουλία ενεργοποίηση εφαρμογή τη οδηγία αυτή, Γιατί είναι αλήθεια ότι έχουμε 24 μήνε καιρό, αλλά καθώ υπάρχει σοβαρή δυσκολία για τι ΜΜΕ που έχουν προβλήματα ε, υποκεφαλοποίηση, πρόσβαση στη χρηματοδότηση, ε, οι 24 ε, μήνες είναι πάρα πολύ γιατί υπάρχει κίνδυνο χεροκοπία. Έτσι λοιπόν από τη σκοπιά αυτή θα ήθελα να καλέσω για την εφαρμογή αυτής της οδηγίας. Τώρα, ποια μέσα για την ε, άρση ε, των προβλημάτων, κυρίως της δημόσιας διοίκησης. Κοιτάξτε, οι θεσμοί λειτουργούν με διαφορετικό χρόνο σε σχέση με το χρόνο των επιχειρήσεων. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Τρίτο θέμα πολύ σημαντικό να ευνοήσουμε την ε, επιχειρηματικότητα των νέων. Ε, τι σημαίνει κυρίως να έχουμε εναλλαγή στις γενναίες αλλά και συνέχεια στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Γιατί κυρίως για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις δεν υπάρχει συνέχεια. Όταν ε, το χαρή σταματά ο επιχειρηματίας να ασκεί τη δραστηριότητά του πεθαίνει η επιχείρηση. Έτσι λοιπόν πρέπει να ευνοήσουμε την είσοδο των νέων και πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο, με ποια κίνητρα. Ο συνάδελφο Μπιτικόφερ, Πρόεδρε, επειδή δεν έχουμε και χρόνο, να παρακαλέσω μόνο το εξή και δεν θα μιλήσω. Αν έχουμε στο μέλλον τόσο λίγο χρόνο, ίσω θα μπορούσατε να φροντίσετε στην αρχή τη συζήτηση να, μιλήσει ένας από, να μιλάει ένα από κάθε ομάδα για να είναι λίγο πιο δίκαιη η κατανομή. Μάλιστα, λέει ο πρόεδρο. Το θέμα είναι αν εγώ πρέπει να επιβάλλω δίκαιου όρου ή μήπω θα πρέπει από μόνοι σα να ε, επιβάλλεται κάποια δικαιοσύνη. Δίκιο έχετε, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι δύσκολα τα πράγματα. Θέλετε να φέσετε ερώτηση πάντω. Δύο θέματα ήθελα να θίξω. Καταρχά, ε, επί τη ουσία, από ό,τι φαίνεται το πρόβλημα είναι στο επίπεδο των κρατών μελών σε ό,τι αφορά αυτή την πράξη για τι μικρέ επιχειρήσει. Θα πρέπει να σκεφτούμε πώ λοιπόν μπορούμε να ασκήσουμε πίεση στα κράτη-μέλη για να τα πάρουν στα σοβαρά. Δεύτερον, υπάρχουν πάρα πολλά σημεία για τα οποία θεωρώ ότι πολλές καλές ιδέες υπάρχουν και τις έχετε υποβάλει κύριε Επίτροπε, αλλά πολλά λείπουν. Για παράδειγμα στο Seed Money λείπει η ιδέα του Angel Investment για το θέμα των δημόσιων συμβάσεων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα πρέπει να το υπογραμμίσουμε πιο έντονα. Η αξιοποίηση ε, επιστημόνων που έχουν φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ο ρόλος των προτύπων. Πολλές φορές το έχουμε συζητήσει με φιλόδοξο τρόπο εδώ πέρα στο Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Ο πρόεδρος, η συνάδελφος Σαρτόρη. Πρόεδρε, σε 30 δευτερόλεπτα ένα πράγμα μπορώ να ρωτήσω μόνο θα καταφέρουμε να ξαναβάλουμε στο κέντρο και της συζήτησης ε, την επιχείρηση, ε, στο επίκεντρο και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο επίκεντρο και της δικής μας Επιτροπής. Γιατί δυστυχώς το ενδιαφέρον του Κοινοβουλίου στρέφεται πάντοτε προσανατολίζεται σε άλλα θέματα. Στην πρότασή σας για την πράξη των μικρών επιχειρήσεων βλέπω αυτή τη δυνατότητα. Ε, θα πρέπει πράγματι οι κανόνες μας να προσανατολιστούν σε μια μεγαλύτερη απλοποίηση. Ευχαριστώ. <clears throat> Eh, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Επίτροπο που παρουσίασε τόσο ενδιαφέρουσες πρωτοβουλίες στη δική μας Επιτροπή και ευχαριστώ και τον κύριο Καγέχα. Είμαι σίγουρος ε, ότι ε, θα λειτουργήσει τόσο εξαιρετικά στο ένα του καθήκοντα όπως και η προκατοχή του. Τώρα, η επιτυχία μιας πολύ μικρής επιχείρησης ή μιας μικρής επιχείρησης πολλές φορές είναι να μεταμορφωθεί σε μεσαία επιχείρηση, να κερδίσει μέγεθος δηλαδή. Ε, αυτή είναι η επιτυχία της. Υπάρχουν κράτη-μέλη στα οποία τιμωρείται η μεγέθυνση μιας μικρής επιχείρησης, τιμωρείται, ποινικοποιείται με ε, νομοθεσίες εργασιακές, ε, γιατί ε, κάτι τέτοιο έχει ως αποτέλεσμα να ζημιώσει η αλλαγή του μεγέθους στην επιχείρηση, όταν η επιχείρηση δηλαδή αποκτήσει συγκεκριμένο μέγεθος, να ζημιωθεί λόγω συνδικάτων ή παραδείγματος χάρη και σε άλλες περιπτώσεις πάλι τιμωρείται η επιχείρηση επιχείρηση μέσω της φορολογίας. Και μπορούν να υπάρξουν και άλλα πολλά που θα ε, ανέφερα εδώ, αλλά δεν θέλω να χρονοτριβώ. Τώρα, η ερώτησή μου είναι, κύριε Επίτροπε, τι έχει σκεφτεί η Κομισιόν ε, έτσι ώστε μία επιχείρηση ε, που από μικρή μετατρέπεται σε μεσαία να μην τιμωρείται από τις δράσεις ορισμένων κρατών μελών και από τις νομοθεσίες ορισμένων κρατών μελών. Γιατί τελικά κανείς δεν μπορεί να ε, καινοτομήσει ούτε ε, να αναπτυχθεί αν δεν έχει και ένα συγκεκριμένο μέγεθος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και κύριε Επίτροπε. Χάρηκα στην εισαγωγή σας που είπατε ότι δεν υπάρχουν διενέξεις όσον αφορά να προσέχει κανείς το περιβάλλον, αλλά να βοηθήσει και τη χώρα της βιομηχανία. Εγώ θα ήθελα να πω, παρόλο που είπατε ότι δείξατε που θα πρέπει να πέσει το βάρος, παρόλα αυτά όμως είναι κατανοητό ότι θα πρέπει να αλλάξουμε τους κανόνες. Έχουμε το Natura 2000. Εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε κλασικές ε, αντιπαραθέσεις που μας εμποδίσαν να έχουμε από τη μια ε, βιωσιμότητα, ε, το θέμα της αρχής της ε, πρόληψης και από την άλλη το να, δώσουμε, ε, να βοηθήσουμε τις ανταγωνιστικές χώρες. Τι εννοείτε δηλαδή, για πείτε μας, εννοείτε ότι θα πρέπει να το δεχτούμε αυτή την πρόκληση αντί να δουλεύουμε και να συνεργαστούμε μαζί. Um, η κυρία Μερκή, ευχαριστώ Πρόεδρε. Υπάρχει αυτό το φλάξιο για την αποδοτικότητα των πόρων και αργότερα θα έχει περαιτέρω επεξεργασία σε αυτό στον οδικό χάρτη. Θα προπταθούν διάφορα μέσα στον οδικό χάρτη. Και αυτή η ανακοίνωση για τις πρώτες ύλες, πώς σχετίζεται με τον οδικό χάρτη. Καλωσορίζω την πρωτοβουλία σας για τις πρώτες ύλες, όπως γνωρίζετε. Θεωρώ ότι είναι πολύ καλή ιδέα να υπάρχει ένα δικό μας μοντέλο για την αντιμετώπιση πρώτων υλών σε διεθνές επίπεδο. Αλλά τι μέσα προτείνετε ιδιαίτερα για τον τρίτο πυλώνα, είναι μέσα για την αποτελεσματικότητα των πόρων, τα οποία θα αναφέρονται στον οδικό χάρτη. Νομίζω ότι αυτό που τελικά λείπει στην πρωτοβουλία για τις πρώτες ύλες είναι η πτυχή της αποδοτικότητας και καλωσορίζω το γεγονός ότι συμπεριλάβατε τα υλικά με βιολογική βάση. Αν οδεύουμε προς την υποκατάσταση των σπάνιων αυτών υλών, χρειαζόμαστε αυτά τα προϊόντα. Μπορείτε να μας εξηγήσετε γιατί προσθέσατε και τα δύο αυτά στοιχεία, το οποίο και υποστηρίζω. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ. Τώρα πώς να σας ζητήσω να απαντήσετε τις ερωτήσεις, όλες τις ερωτήσεις. Α, θα μπορούσατε να προσπαθήσετε σε πέντε, άντε έξι λεπτά. Να πείτε λίγο τα πιο σημαντικά και τα υπόλοιπα τα γραπτά. Θα είσαστε πραγματικά ήρωας. Ευχαριστώ Πρόεδρε για την πρόσκληση. Ε, με όλες αυτές τις ερωτήσεις θα μπορούσαμε να μείνουμε εδώ μέχρι τις μία και να συζητούμε. Χαίρομαι πάρα πολύ για όλες τις ερωτήσεις ε, και θα προσπαθήσω να προσανατολιστώ σε αυτά που υπογράμμισα κατά την παρουσίασή μου. Καταρχήν προς την κυρία Σαρτόρη. Πραγματικά είναι προτεραιότητα για μένα να ξαναθέσω στο επίκεντρο της οικονομικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης μια ισχυρή δράση υπέρ της πραγματικής οικονομίας. Να ξαναθέσω στο επίκεντρο μετά από χρόνια πολιτικής που βασιζόταν στα χρηματοοικονομικά, στις υπηρεσίες και τα λοιπά, να ξαναθέσω στο επίκεντρο την πραγματική οικονομία. Και επομένως τη βιομηχανία και την επιχείρηση με όλες τις δυνατές δράσεις έτσι ώστε πάντοτε υπάρχει ένα καινούριο μοντέλο βιομηχανίας ή επιχείρησης. Αλλά είμαι πεπισμένος ότι μόνο ξαναθέτοντας τα αυτά στο επίκεντρο θα μπορέσουμε να τηρήσουμε και να εφαρμόσουμε τη συνθήκη της Λισαβόνας και να βασιστούμε στην κοινωνική οικονομία της αγοράς. Η αγορά λειτουργεί μέσω της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων και της βιομηχανίας και ο στόχος είναι πάντοτε η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για τους νέους μας Εκινώντας ε, λοιπόν και από ένα σύστημα επιχειρηματικών που να ανοίγει προοπτικές για τους ε, νέους. Γιατί οι νέοι δεν πρέπει να επιθυμούν να πάνε να γίνουν μόνο δημόσιοι υπάλληλοι, αλλά θα πρέπει να γίνονται και νέοι επιχειρηματίες, να ρισκάρουν. Υπάρχει το πρόγραμμα Έρασμος για τους νεαρούς επιχειρηματίες, το οποίο σκοπεύω να εφαρμόσω στην πράξη. Τώρα πώς θα βοηθήσουμε την δημιουργία ή την επιβίωση των εθνικών επιχειρήσεων. Αυτό είναι ένα ερώτημα το, με το οποίο μας απασχολεί, το οποίο απασχολεί πολλούς από εμάς. Ε, η κυρία Καρβάλιο το έθεσε πολύ σωστά. Το ζήτημα αυτό το βάλαμε επίσης στο επίκεντρο των δράσεων ακόμα και πριν από την παρουσίαση της επικαιροποίηση της πράξης για τις μικρές επιχειρήσεις. Υπάρχει ένα κείμενο εμβάθυνση, το οποίο μάλιστα εγκρίθηκε την περασμένη εβδομάδα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είμαστε πολύ ευτυχεί γι' αυτό, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το λεγόμενο Οικονομικό Φόρουμ για τις ΜΜΕ, όπου διάφοροι ομιλητές, ε, μεταξύ των οποίων πολλοί ευρωβουλευτές, ο κύριος Ντεάντζελης νομίζω είχε συμμετάσχει σε αυτό το φόρουμ, πολλοί ομιλητές λοιπόν ε, εξατομίκευσαν τα προβλήματα και πρότειναν λύσεις για την πρόσβαση στην χρηματοδότηση. και τη χρησιμοποίηση του τραπεζικού συστήματος για να χορηγήσουμε πιστώσεις και χρηματοδοτήσεις στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ζήτημα κλειδί το οποίο πρέπει πραγματικά να αντιμετωπιστεί. Γιατί ακόμα και τώρα η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων πρέπει να διευκολύνει τη χορήγηση χρηματοδοτήσεων στις... και πιστώσεων στις τράπεζες για να μπορούν να στηρίξουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το χρηματιστήριο του Λονδίνου εκδήλωσε, ε, δήλωσε ότι είναι διαθέσιμο ε, να επενδύσει υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Εμφανίστηκε διαθέσιμο να επενδύσει. Εν ώψη αυτή τη διαθεσιμότητα, ζήτησα από τον εντεταλμένο αντιπρόσωπο του χρηματιστηρίου του Λονδίνου να συμμετέχει στο Οικονομικό Φόρουμ για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και εκείνος δέχθηκε την πρόσκληση. Ε, το φόρουμ θα διεξαχθεί σε μερικές μέρες και το χρηματιστήριο του Λονδίνου λοιπόν, αφού διακήρυξαν αυτόν διαθέσιμο να χρηματοδοτήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, θα συμμετέχει σε αυτό το φόρουμ το οποίο είναι ανοιχτό και το οποίο σίγουρα θα δώσει απαντήσεις, κάποιες απαντήσεις στους πολίτες που είναι και επιχειρηματίες. Τώρα, για να απαντήσω και στην κυρία Καρβάλιο. Μιλάμε για ευκολότερη πρόσβαση σε εγγυήσει, ε, με ένα ενισχυμένο σύστημα εγγυήσεων, με δράσεις βελτίωσης της πρόσβασης ε, στην ε, πίστοση, ακόμα και για, ακόμα και για τις επιχειρήσεις κινδύνου. Όπως είπαμε πρέπει να υπάρχουν και εννέα κέντρα εξυπηρέτησης στα κράτη-μέλη για την διευκόλυνση της πρόσβασης στις πιστώσεις. Ένα άλλο θέμα που θύχτηκε για την στήριξη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και που θέλει να δώσει μια συγκεκριμένη απάντηση στον επιχειρηματία, να διευκολύνει αυτόν που θέλει να ασκήσει επιχειρηματική δραστηριότητα και ο οποίο λόγω της κρίσης ε, ίσω αντιμετωπίζει προβλήματα, ίσω μπροστά στο ενδεχόμενο τη πτώχευση να βρίσκεται. Ε, ξεκινούμε, μάλλον ε, θελήσαμε να δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία στου επιχειρηματίε, μειώνοντα στα τρία χρόνια το πολύ μέχρι το 2013 τους όρους αποκατάστασης και ρευστοποίησης των χρεών, των οφειλών. Αυτό φυσικά για εκείνους τους ε, ε επιχειρηματίες που δεν πτωχεύουν δόλια βέβαια. Που δεν μηχανεύονται την πτώχευση. και μάλιστα ασκούμε πίεση στα κράτη-μέλη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει κανονιστική αρμοδιότητα άμεση. όπως συνέβη με την οδηγία για, την, για τις καθυστερούμενες ε, πληρωμές. Ο κύριος Ντε Άντζελης ε, όταν κατά την παρουσίαση της επικαιροποίηση της πράξης για τις μικρές επιχειρήσεις στην Ρώμη έθεσε και ερωτήσεις εκεί στους εκπροσώπους του, του Ιταλικού κράτους. Ε, ίσως το ίδιο γίνει και με την γαλλική κυβέρνηση, με την αγγλική κυβέρνηση αυτή την εβδομάδα, την επόμενη εβδομάδα με την Ουγγαρία και τη Γερμανία και πάλι θα μπορέσουμε να απευθυνθούμε, να αποτανθούμε στις κρατικές αρχές για τη διευκόλυνση των επιχειρηματιών που βρίσκονται, που αντιμετωπίζουν προβλήματα. Τώρα, για το όσο αφορά το ερώτημα για την ε, πρόοδο και την πιο μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει πολλά πάνω στο θέμα αυτό. Έχει κάνει πολλά για τα θερμοκοιτίδες των επιχειρήσεων, τις δεσμίδες των επιχειρήσεων. στήριξη στις καινοτόμες δράσεις, ε, στις συμπράξεις μεγάλων και μικρών επιχειρήσεων, στις συμπράξεις επιχειρήσεων και πανεπιστημίων και σε διεθνές επίπεδο ακόμη. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έτσι εντάσσονται σε ένα τέτοιο σχήμα, πιο καινοτόμο, πιο αρθρωμένο, πιο διαρθρωμένο, λαμβάνουν βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η καινοτομία είναι ένα άλλο στοιχείο. Υπάρχει ένα πρόβλημα με την εκπαίδευση. Ήδη μίλησα με τον, κύριο, με τον Επίτροπο Βασίλειο για να οργανώσουμε κάτι και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη σχέση που υπάρχει μεταξύ της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της εισόδου στον κόσμο της εργασίας. Τώρα για τη μείωση των ε, διοικητικών εμποδίων και βαρών. Ε, και ο κύριος Λίμπεν το έθεσε αλλά και άλλοι βουλευτές στη διάρκεια της συζήτησης. Εμείς θέλουμε να βελτιώσουμε όλο το κανονιστικό πλαίσιο το ευρωπαϊκό. για όλες τις νομοθετικές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την εφαρμογή της αρχής ότι οι επιχειρήσεις πρέπει μία φορά να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε μία αρχή και όχι σε πολλές. Επίσης υποχρεώνοντας τα κράτη-μέλη να ε, ε, εφαρμόζουν σωστά τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Παράδειγμα, η ρύθμιση REACH Aver fatto pubblicare in tutte le lingue mm, έχουμε μειώσει, να και κάτι άλλο συγκεκριμένο, υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Μειώσαμε το στα, στα 60% από 90% το ποσοστό των ιτροδών ενώσεων έτσι ώστε να διευκολύνουμε την ε, υλοποίηση της ε, νομοθεσίας αυτής από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ακόμα και στα υλικά οικοδομής, όπως ξέρετε πολύ καλά, είχαμε και την ε, συζήτηση και πάλι εκεί οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις βοηθήθηκαν και διευκολύνθηκαν. Τώρα. Ancora le eh, Πριν να περάσω στις πρώτες ύλες, ε, νομίζω ότι απάντησα σε πολλές από τις ερωτήσεις που τέθηκαν. Ε, α, σε ό,τι αφορά και τη μείωση των εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να ζητήσουμε από τι δικέ μα επιχειρήσει στην Ευρώπη να πάνε πέρα από το όριο του 20% αν δεν υπάρξει παγκόσμια συμφωνία γιατί αυτό θα είχε αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα όλου του συστήματο. Ό,τι αφορά τώρα τι αυστηρέ αγορέ εργασίας, ναι, συμφωνώ. Στην Ευρώπη ισχύει κάτι τέτοιο και πάντοτε με την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων θα μπορούσαμε να σκεφτούμε τη συνέψη συμφωνιών μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων σε τοπικό επίπεδο ή σε επίπεδο επιχείρηση. Είναι αλήθεια όσα υπόθηκαν ότι πολλές φορές ποινικοποιούνται επιχειρήσεις που θέλουν να μεγεθυνθούν. Γι' αυτό πιστεύω εγώ στο σύστημα των κλάστερ ε, που έχουμε στην Ευρώπη και έτσι θα συνεχίσουμε σε ό,τι αφορά τώρα τις πρώτες για την Natura 2000. Εμείς καθόλου δεν αμφισβητούμε. Απλώς ε, έχουμε εκδώσει κάποιες ε, διατάξεις ερμηνευτικές σε ό,τι αφορά τώρα ε, τα αστικά ορχεία. Σίγουρα ξεκινήσαμε μια συζήτηση, υπάρχει μια σύμπραξη καινοτομία που προβλέπεται ε, για την εφαρμογή της ε, ανακοίνωσης για την καινοτομία. Το πρώτο, όπως ξέρετε, αφορά τη γύρανση του πληθυσμού ε, και το πώς θα προστατεύσουμε την υγεία των πολιτών μας και η δεύτερη σύμπραξη για την καινοτομία θα αφορά συγκεκριμένα την ανακύκλωση και την αντικατάσταση των πρώτων υλών. Αυτό φυσικά προστατεύει και το περιβάλλον. Εγώ θα ήθελα πολλές επιχειρήσεις και ιδιωτικές να συμμετάσχουν σε αυτή τη σύμπραξη ε, και όπως ε, ξέρετε έχουμε μέχρι τώρα ε, στις λάμπες ένα υλικό που δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε παραδείγματος χάρη δεν μπορούμε να κάνουμε ανακύκλωση των υλικών αυτών που έχουμε στις λάμπες, δεν έχουμε βρει ακόμη τον τρόπο και σε ό,τι αφορά την ενεργειακή αποδοτικότητα θεωρώ ότι η πρόταση της κυρίας Μέρκης με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο. Θα την υιοθετήσω και εγώ και έτσι θα προσπαθήσω να αντιμετωπίσουμε και το θέμα του ενεργειακού, της ενεργειακής αποδοτικότητας. Φυσικά το θέμα των πρώτων υλών δεν είναι κάτι που έχει ολοκληρωθεί. Χρειάζεται να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε συνεχώς γιατί εξελίσσεται η κατάσταση. Έτσι λοιπόν κάθε πρωτοβουλία και κάθε ιδέα ε, είναι ευπρόσδεκτες ε, στο τομέα αυτό το κοινοβούλιο. Μπορεί να συνεισφέρει είτε για το θέμα των πρώτων υλών, γιατί με τη συζήτηση που θα λάβει η χώρα για την έκθεση Μπιτικόφερ σίγουρα θα μπορέσουν να προκύψουν νέες ιδέες, εγώ είμαι πάντοτε ανοιχτός ε, στο να ε, λαμβάνω προτάσεις από τους ευρωβουλευτές. Τώρα για την πρώτη ερώτηση, τι μπορούμε να κάνουμε εμείς ε, και τι μπορεί να κάνει και το Κοινοβούλιο. Τι μπορεί να κάνει λοιπόν το Κοινοβούλιο, να συνεχίσει αυτό που έκανε μέχρι τώρα, να ασκεί πίεση στα κράτη-μέλη και στο Συμβούλιο, έτσι παραδείγματο χάρη η οδηγία που έχει μπλοκαριστεί στο Συμβούλιο για την Ευρωπαϊκή Εταιρεία, να μπορέσει να ακουστεί και η φωνή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να επιμένει έτσι ώστε τα κράτη-μέλη να επιταχύνουν την εφαρμογή τη οδηγία για την καθυστέρηση πληρωμών. Κοιτάξτε, ε, ε, μια πρωτοβουλία από πλευρά Κοινοβουλίου μπορεί να αναλυφθεί, να ασκηθεί μια πίεση για να γίνει ένα βήμα προς τα μπρος. Αν ε, το Κοινοβούλιο λοιπόν είναι πολύ προσεκτικό και επαγρυπνεί για το θέμα των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, για μένα πάντοτε θα είναι πιο εύκολο να θέτω στο επίκεντρο της συζήτησης το θέμα αυτό. Λοιπόν, ε, δεν θα με καλέσει ο πρόεδρος ε, σε δίπλα από ό,τι κατάλαβα, γιατί με ακρηγόρησα. Να σας ευχαριστώ τον Επίτροπο και να ευχαριστήσω ιδιαίτερα λέει ο πρόεδρος του Διερμηνής, οι οποίοι έμειναν λίγο παραπάνω μαζί μας. Ε, σας ευχαριστώ και κυρίες και κύριοι σας παρακαλώ να αποχωρήσετε ησύχως. Θέλω σε ένα λεπτό να ξεκινήσω την συνεδρίαση των συντονιστών. Θα μας κάνετε μεγάλη χάρη αν αποχωρήσετε γρήγορα γρήγορα.